Πριν να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, ε, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα οικογένειε των θυμάτων ε, του τραγικού ατυχήματος στην Αιθιοπία χθες. 157 άτομα έχασαν ε, τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Σήμερα είναι η 15η επέτειος ε, της ε, τρομοκρατικής επίθεσης στη Μαδρίτη που είχαμε πολλούς τραυματίες και νεκρούς. Η 11η Μαρτίου έγινε μια συμβολική ημερομηνία και αφιερώνουμε τη μέρα αυτή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Όπως ε, μας ε, υπενθύμισε και η επίθεση δηλή στο Στρασβούργο πριν από τα Χριστούγεννα, πρέπει πάντοτε να αγωνιζόμαστε για να υπερασπίσουμε τις αξίες μας ε, και τις ελευθερίες μας από τη βαρβαρότητα της τρομοκρατίας. Πριν πέντε χρόνια η Κρυμαία προσαρτήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία. Είχαμε διάφορα ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο και είδαμε ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας αποτελεί παραβίαση του διεθνού δικαίου. Και ε, έχουν υπογραφεί πάρα πολλές συμφωνίες από τη Ρωσία, ε, το Memorandum της Βουδαπέστης, ο Χάρτης του Ελσί λοιπά. Σήμερα υποστηρίζουμε και πάλι την εδεφική ακαιρεότητα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Από την Πέμπτη το βράδυ ένα μεγάλο μέρος ε, της Βενεζουέλας βρίσκεται χωρίς ρεύμα. Πρόκειται για την τέταρτη μέρα ε, στα σκοτάδια. Η κατάσταση αυτή είναι δραματική και πάρα πολλές ζωές, κυρίως ε, παιδιών, νεογέννητων, απειλούνται. Πολλά παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει ρεύμα στα νοσοκομεία. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνουμε κλίση έκτακτης ανάγκης στη διεθνή κοινότητα προκειμένου αυτή η άδικη κατάσταση να σταματήσει. Πρόκειται για, για μια κανονική, σε μια κανονική χώρα δεν θα πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Η ευθύνη της ε, έλλειψης ε, υποδομών ε, είναι της κυβέρνησης. Ο Μαδούρο επιδιδώνει την ανθρωπιστική κρίση και καταστρέφει τις ζωές του λαού της Βενεζουέλας. Θεωρώ ότι ξεκινά ε, εκ νέου η συνεδρίαση που είχε διακοπεί στις 14 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά ε, έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Τα πρακτικά λοιπόν, λοιπόν εγκρίνονται. Έτσι όπως έχουν υποβληθεί η Επιτροπή ε, των ε, νομικών θεμάτων έκνε τον έλεγχο της εντολής βιστερον σκούτσος ε, σε σχέση με τις 10 και 24 Ιανουαρίου φέτος υπάρχουν αντιρρήσεις έτσι λοιπόν η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προβαίνει στο έλεγχο της εντολής στις 20 Σεπτεμβρίου 1964 στην αποστολή που δόθηκε στον κύριο Λαμασούρ ε, σε σχέση με τη διδασκαλία στην Ευρώπη και θεωρείται ότι είναι συμβετό. Η Επιτροπή Συμμεταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1β του κανονισμού, ε, υπάρχει το κείμενο στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας ε, και θα δημοσιευτεί. Η ερμηνεία θεωρείται ότι εγκρίνεται αν μέσα σε 24 ώρες καμία πολιτική ομάδα δεν φέρει αντίρρηση σε σχέση με το αν φτάσει το λιγότερο καθόλου. Η Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει διοργανικέ διαπραγματεύσει σύμφωνα με το άρθρο 69C1 του κανονισμού. Ε, η εντολή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα τη Ολομέλεια και ο τίτλο θα δημοσιευτεί στα πρακτικά τη Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 69 ο παράγραφος 2 αριθμός των βουλευτών ή πολιτικών ομάδων ε, ίσο με το μέσο κατόφλι μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα 12 Μαρτίου να τεθεί σε ψηφοφορία ε, η έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αν όμως δεν παρουσιαστεί τέτοιο αίτημα ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο θα μπορέσει η Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 105 γάμα η διάσκεψη των Προέδρων της Επιτροπής με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει υπήρξε αντίρρηση στις συστάσει τη Επιτροπής ΕΚΟΝ να μην ε, φέρει αντίρρηση σε διάφορες κατοξιδότητε πράξει. ε, υπάρχουν διαθέσιμε συστάσεις αυτές στην ε, ιστοσελίδα τη Ολομέλειας αν μέσα 24 ώρες ε, καμία πολιτική ομάδα ή μέλη τουλάχιστον ίσο με το χαμηλό κατόφλι δεν φέρουν αντιρρήσει, τότε θα τεθεί σε ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 114 του κανονισμού έχω λάβει ε, τρία αιτήματα ε, να συζητηθούν κατ' επιδότως. Ε, έχουμε τους κανόνες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας λόγω της αποχώρησης του Ορειμένου Βασιλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, έχουμε την ε, δραστηριοποίηση των ε, πλοίων του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στο ύδατα της Ένωσης. Και επίσης έχουμε και το θέμα της σύνδεσης της υδροδρομικής. Επίσης, αύριο το πρωί θα έχουμε την ψηφοφορία για τα τρία αιτήματα στην έναρξη της συνεδρίασης. Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Σα ενημερώνω ότι την Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω 12 πράξεις που έχουν εγκριθεί δυνάμει τη τακτικής νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. τίτλοι των πράξεων θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης. Περνάμε τώρα ε, στην, ε, το σχέδιο μερική διάταξη που εγκρίθηκε στις 7 Μαρτίου, σύμφωνα με το άρθρο 149, έχει διανεμηθεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με το άρθρο 22.4 έχετε το προνόμιο να εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο επισήμως. Από τις 29 μέχρι τις 31 Μαρτίου θα λάβει χώρα στη Βερόνα το Παγκόσμιο Συνέδριο ε, Οικογενειών. Για όσους δεν το γνωρίζετε, διαδίδει ομοφοβία και ε, ε, επιτίθεται στη σεξουαλική αυτοδιάθεση. Επίσης, η SPRC την έχουν κατατάξει αυτή την οργάνωση ως ομάδα που μισεί τους LGBT. Και εσείς είστε ομιλητής εκεί κύριε Πρόεδρε. Μετά εξαφανιστήκατε από την ιστοσελίδα. Η ε, διακομματική ομάδα, το Intergroup των ΛΟΑΔΜ, σας έχει ρωτήσει επανειλημμένως τι θα κάνετε. Όταν αναλάβατε είπατε ότι θα εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο και τις θέσεις του. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει υπερψηφίσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και την ε, σεξουαλική αυτοδιάθεση. Εσείς θα ανταποκριθείτε σε αυτή την ε, δέσμευσή σας και θα υπερασπιστείτε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μεταβείτε και θα συμμετάσχετε σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα είμαι στο ΣΥΣΥ για, μαζί με τον πρόεδρο του Ιταλικού Συμβουλίου, τον κύριο Κόντε, και την καγκελάριο της Γεμαρλίας, την κυρία Μέρκελ. Για την ημερήσια διάταξη, μόλι είδα μια έκθεση, ένα δημοσίευμα ότι θα έρθει λέει στο Στρασβούργο η κυρία Μέη για να συναντηθεί με τον κύριο Γιούνκερ. Το γνωρίζετε ε, αυτό, κύριε Πρόεδρε, και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα την προσκαλέσετε να απευθύνει το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δώστε μου χρόνο να απαντήσω. Πρέπει να απαντήσω. Δώστε μου το χρόνο. Διαφορετικά δεν μπορώ να απαντήσω. Αν έρθει η κυρία Μέη, ενημερωθήκαμε ότι αν έρθει, θα έρθει να συναντήσει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα έρθει αργά το βράδυ. Και αν έρθει στο Κοινοβούλιο θα τη συναντήσω, πιστεύω, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει για αύριο το πρωί. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να απευθυνθεί στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να, να αναφερθώ στο κανονισμό 11.3. Στο άρθρο αυτό δεν μπορούν να προσβάλλουν βουλευτέ, άλλου βουλευτέ και κυρίω ανθρώπου που έρχονται να μιλήσουν στην Ολομέλεια. Στην προηγούμενη Ολομέλεια είδαμε ντροπιαστικό θέαμα από την πλευρά του συναδελφού Φερχόφστα, το οποίο προσέβαλε τον Ιταλό Πρωθυπουργό, ο οποίο εκπροσωπεί 60 εκατομμύρια Ιταλού πολίτε. Ζητώ λοιπόν ο κύριος Φερκόστατ, ο οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην αίθουσα αυτή, θεωρώ, να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν ναι, σα λέτε ότι δεν πρέπει ο Φερχόφστατ να προσβάλλει του άλλου, και εσεί δεν πρέπει να προσβάλλετε τον κύριο Φερχόφστατ. Τώρα, όποιο ε, έχει ε, εκλεγεί από το λαό είναι αξιοπρεπή. Ε, κοιτάξτε, εμένα μου φαίνεται ότι ήταν πολύ αρνητικό αυτό που έκανε. Ε, κοιτάξτε, ε, κυρία Μέρκελ, αυτό τι σημαίνει, ότι σε αυτό το κοινοβούλιο μπορούμε να δράμε με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, κυρία Ιντβελτ. I thought it was in the European Parliament. Apparently, it's the Italian Parliament. I would like to briefly come back to. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της κυρίας ε, Ρέινκε γιατί πάρα πολύ γρήγορα το ξεπετάξατε πράγματι. Είχατε μπει στον κατάλογο σε ένα από του κύριους ομιλητές στη διάσκεψη στην οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος και σας ζητήσαμε να το επισαφήνισετε αυτό με επιστολή. Και μετά αφού στείλαμε την επιστολή εξαφανίστηκε το όνομά σα από την ιστοσελίδα ω ομιλητή. και δεν λάβαμε καμία γραπτή εξήγηση. Επιμένω λοιπόν να μα δώσετε μια γραπτή επεξήγηση. Κύριε Βουλευτέ, αν θέλετε να σας στείλω γραπτός απάντηση, ήταν ήδη έτοιμη. Να το πω εδώ, ε, στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικότερο να το πούμε ότι θα σταλεί γραπτός ε, η επιστολή. Εγώ εκείνες τις μέρες θα είμαι στο Ασίσι και δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την πολεμική. Δεν θα πάω. Αν ε, έχω προσκληθεί και δεν πάω, δεν μπορείτε να με κατηγορείτε τώρα εδώ επειδή έχω προσκληθεί. Τώρα ποιο ο λόγο να συνεχίσουμε αυτή την πολεμική. Παρακαλώ. Κριμητικά. Η κυρία Ιντβελτ όμω. νομίζω το κάνετε χειρότερο, Πρόεδρε. Γιατί μπορεί να έχετε άλλε υποχρεώσεις εν τω μεταξύ, παράλληλα. Αλλά καταλαβαίνω ότι όχι μόνο προσκληθήκατε, αλλά αναφέρεστε και ως κεντρικός ομιλητής για μια οργάνωση ομοφοβική, σεξιστική, για ανθρώπου που μάχονται κατά των αξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να έβαλαν το όνομά σα στην ημερήσια διαταξή χωρί να το γνωρίζετε. Αυτό ίσω είναι εξήγηση, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε τη δική σα επιστολή. Να σα το επαναλάβω για νιωστή φορά. Θα στείλω την απάντηση γραπτό. Όμως ε, εδώ υπάρχει κυριαρχία στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι μετράει περισσότερο η απάντηση εδώ. Και καθώς εγώ θα πάω αλλού, δεν ξέρω τι να κάνουμε τελικά. Εγώ δεν είμαι ούτε υπουργό εσωτερικών που μπορεί να απαγορεύει διάφορες συνεδρία στη χώρα. αν πάω κάπου αλλού που είναι ο Πρωθυπουργό και είναι και η κυρία Μέρκελ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κανείς. Ο κύριος Μαριάς. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θέλω να μιλήσω για την ημερήσια διάταξη και θέλουμε ως ecr να κάνουμε την εξής πρόταση η θεομηνία που έπληξε την περιφερειακή ενότητα χανίων στην κρήτη το διήμερο 24 25 φεβρουαρίου προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε δημόσιες υποδομές και σε ιδιωτικές περιουσίες. επισκέφθηκα ήδη δύο φορές τις πληγείσες περιοχές και η περιοχή της ενότητας χανίων μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο γέφυρες κατεστραμμένες δρόμοι άνοιξαν στα δύο εκτεταμένες κατολιστήσεις αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδε καταστράφηκαν. την προηγούμενη εβδομάδα στην τεχνική σύσκεψη το ecr είχε ζητήσει να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας για συζήτηση το ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών και της αποζημίωσης των πληγέντων λόγω θεομηνίας στην περιφερειακή ενότητα χανίων προτείνουμε λοιπόν σήμερα μια και το αίτημά μας αυτό δεν έγινε δεκτό από τις άλλες πολιτικές ομάδες διότι δήθεν η ημερήσια διάταξη ήταν κορεσμένη προτείνουμε λοιπόν σήμερα δευτέρα ως τελευταίο θέμα να προσθεθεί το θέμα της και να εκδοθεί ψήφισμα για τη λήψη μέτρων στήριξης προς τους πληγέντες της θεομηνίας στην περιφερειακή ενότητα χανίων καθώς και για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης των καταστροφών. θεωρώ ότι είναι ένδειξη μιας αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας στην περιφερειακή ενότητα χανίων και καλώ τους συναδέλφους να κάνουν δεκτό το αίτημα του ecr να προσθεθεί ως όγδοο θέμα το ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών στην περιφερειακή ενότητα χανίων και να εκδοθεί και ψήφισμα. και παρακαλώ κύριε πρόεδρε να το θέσετε αυτό σε ψηφοφορία ζητώντας για άλλη μια φορά τη στήριξη των συναδέλφων. ευχαριστώ. Αυτή ήταν μια παρέμβαση για την ε, τροποποίηση της ημερησίας διάταξης. Ε, να προσθέσουμε μια συζήτηση με ψήφισμα για τις πλημμύρες στην Κρήτη. Υπάρχει κάποιος που να είναι κατά ή που να θέλει να τοποθετηθεί κατά και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε. Επομένω, έρχεται η ψηφοφορία για την πρόταση της ομάδας ECR. Ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρόταση. Ο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζήτησε ο τίτλος της ε, δήλωσης της ΥΠΑ ε, της εκπροσώπου. Τι θέλετε παρακαλώ. Thank you very much uh, for choosing... Ευχαριστώ πολύ. Η την τρίτη ζητούμε. Διακόπτη πρόεδρος. Αν κάνετε υπομονή, θα παρουσιάσω όλες τις προτάσεις όλων των ομάδων, αλλά με τη σειρά. Κυρία Μπεραστή, τι θέλετε. Δεν θέλω να διαταράξω τη διάταξη των εργασιών, απλώς ε, ήθελα να σημειώσετε ότι ήμουν κατά της πρότασης που έγινε και δεν έχω την κάρτα ψηφοφορίας μαζί μου. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, για την Τρίτη έχουμε μια σειρά προτάσεων ε, τροποποίηση. Ξεκινάμε από το ΕΛΚ, το οποίο ζήτησε ο τίτλο τη δήλωση τη εκπροσώπου για τις εξωτερικές υποθέσεις για ένα ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων ε, για τις παραδείγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλάξει ε, πράξη Μαγνής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρέντα για να παρουσιάσει το αίτημα της πολιτικής του ομάδας, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση ε, εύκολα γίνεται κατανοητή. Θέλουμε να προσθέσουμε αυτή τη βασική αναφορά στο Μαγνίτσκι, γιατί είναι αναγνωρισμένο αυτό, ήδη και στην κοινή μας γνώμη, ως αναφορά κοινώ ε, παραδεκτή. για το πώς επιβάλλουμε κυρώσεις και πώς τιμωρούνται όλες οι υποθέσεις διαφθοράς και προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευκρινίζει τη στράτευσή μας αυτή η αναφορά στην υπόθεση Μαγνίτση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η κυρία Σαρτζεντίνη θέλει να μιλήσει κατά. Yes, indeed, Chair. Would like... Ναι, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω κατά. Δεν βοηθάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε τον τίτλο ε, μιλούμε για ένα παγκόσμιο νέο καθεστώς κυρώσεων και δεν ε, επικεντρωνόμαστε σε μία χώρα. Προσπαθούμε να συνάψουμε και συμμαχίες και στα κράτη-μέλη και εδώ. Και αν βάλουμε στην επικεφαλίδα το όνομα του και δεν πρόκειται να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. Είναι και εκτός θέματος. Γιατί αυτό αφορούσε κυρίως τη διαφθορά και ε, τα οικονομικά εγκλήματα, ενώ εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία επώνυμη. Έχουν βαρετά ονόματα οι ευρωπαϊκοί νόμοι και δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει συμπεριλάβει τον όρο Μαγνίσκι. Ούτε ο Καναδάς, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η χώρα αυτή δεν επιτρέπει ε, ούτε αποζημιώσεις, ούτε δημοκρατική ε, ε, ε, επισκόπηση και ευλογία Εγώ θέλω και εμείς να παραμείνει όσο έχει ο τίτλος. Λοιπόν, να ψηφίσουμε την πρόταση του ΕΛΚ για τροποποίηση του τίτλου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται η πρόταση. Τρίτη. Πάντοτε ε, η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησε μια συζήτηση για την έκθεση Λόκεγκαρτ σε σχέση με τι απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε που προβλέπεται για ψηφορία Τετάρτη να προσθεθεί ω έκτο σημείο το απόγευμα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Συναλόβα για να παρουσιάσει το αίτημα τη ομάδα τη. Yes, indeed, the group Όντω, οι σοσιαλιστέ ζητούν συζήτηση, στον συζήτηση για την τοπική προσβασιμότητα και ο λόγος είναι διότι η οδηγία αναφέρεται σε άνθρωπους με αναπηρίες στην πρόσβαση σε καθημερινές ευκολίες και γι' αυτό ζητούμε συζήτηση διότι η οδηγία είναι πολύ σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνεται στην κοινή δήλωση εδώ και δύο χρόνια γιατί πρόκειται για δύο οργανική προτεραιότητα. Μετά από το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου, η συζήτηση ήταν ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι δεσμεύεται υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες και έτσι θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν πολύ περισσότερα στον τομέα αυτών. Θέλει κάποιο το λόγο για να μιλήσει κατά. Τότε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η πρόταση. Επομένως, μια συζήτηση για την έκθεση Λόκεγκαρτ για, που προβλεπόταν για ψηφορίες Τετάρτη προστίθεται ως έκτο σημείο το απόγευμα. Τρίτη πάλι η ομάδα Άλντε ζήτησε μία δήλωση της είπα της εκπροσώπου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα να προσθεθεί ως τρίτο σημείο το απόγευμα μετά την έκθεση κάτι πήρε για την έκθεση 2018 για την Τουρκία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση με ψήφισμα που θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νάρτη για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη Βενεζουέλα υπάρχει ανθρωπιστική καταστροφή και έχει ξεπεράσει τα όρια της τραγωδίας και τις τελευταίες πέντε μέρες είναι στο σκοτάδι μετά την ολέθρια διαχείριση της κλεπτοκρατίας στη Βενεζουέλα. Περάσαμε από το δράμα τώρα στην απόλυτη άβυσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να έθελο τυφλή μπροστά σε μια κατάσταση, σε μια χώρα που είναι τόσο κοντά μας. Γι' αυτό θέλουμε συζήτηση με ψήφισμα για την κρίση και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γκονζάλες ε, Πόνς, θέλετε να προστίθετε να προσθέσετε κάτι στην πρόταση του κυρίου Νάρτ. Θέλω να πω ότι η πολιτική μας ομάδα στηρίζει την πρόταση του κυρίου Νάρτ. Εκατό ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σημαίνει ότι έχουν χαλάσει όλα τα τρόφιμα, έχουν χαλάσει όλα τα φάρμακα. Και όταν συνταχθεί το ψήφισμα θα ζητήσει η ομάδα μου να ε, ενισχυθούν οι κυρώσεις πολύ έντονα κατά του Μαδούρου και κατά όλων των αρκοσυνεργατών του. Συμφωνείτε, θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο στο αίτημα του κύριου ε, Νάτ, ο κύριος Λαμπέρ. Πρόεδρε, μακριά από μένα το να υποτιμήσω την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη σοβαρότητά της. Ωστόσο, έχει γίνει συνήθεια εδώ στο Κοινοβούλιο να βάζουμε την κατάσταση στη Βενεζουέλα σε όλες τις συνόδους ολομέλειας στην ημερήσια διάταξη. Και διαπιστώνω ότι ορισμένοι από εμάς ε, χειραγωγούν την κατάσταση και την εργαλειοποιούν για να κάνουν πολιτική λεονταρισμό. Και εσείς κύριε Πρόεδρε δεν είστε τελευταίος μεταξύ αυτών. Τι να την κάνουμε άλλη μια συζήτηση εδώ. Δεν πρόκειται να λύσει τη βαριά κατάσταση και τη σοβαρή που ζει αυτή η χώρα. Και θα προσθέσω αν κάποιοι αγαπούν τόσο την κατάσταση στη Βενεζουέλα να μαζέψουν υπογραφές έτσι ώστε να συσταθεί ειδική επιτροπή για τη Βενεζουέλα και εκεί θα έχετε ε, την ευκαιρία να συζητήσετε ε, μέχρι κορεσμού τι γίνεται με το Μαρόκο, την Αίγυπτο λοιπά. Περιέργως το κοινοβούλιο μας είναι πολύ πιο σιωπηρό. Αλλά οι χώρες αυτές προφανώς μας είναι κοντινές και γεωγραφικά. Αλλά φαίνεται μάλλον ότι τις χρειαζόμαστε για να λύσουμε διάφορα ευρωπαϊκά προβλήματα. Ευχαριστώ. Επομένως, να περάσουμε στην ψηφοφορία της πρόταση της ομάδας των φιλελευθέρων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση, επομένως προστίθεται η δήλωση της ΥΠΑ της εκπροσώπου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα ως τρίτο σημείο το απόγευμα μετά την έκθεση Πύρη για την έκθεση 2018 σε σχέση με την Τουρκία. Πέμπτη ομάδα των Πρασίνων και η ομάδα FTD έχουν ζητήσει συζήτηση για την προφορική ερώτηση, κανόνες για την ευημερία των ζώων στην ιδετοκαλλιέργεια να κλείσουν με ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην επόμενη σύνοδο στις Βρυξέλλες. Κύριος Λαμπέρ. Κύριος Λαμπέρτς, άλλο θέμα που δεν συνηθίζουμε να συζητούμε εδώ είναι ε, τα δεινά που υφίστανται τα ζώα και η ευζοία και η ευημερία των ζώων. Όλο και πιο σαφές καθίσταται διαβάζοντας κανείς την επιστημονική βιβλιογραφία ότι τα ψάρια στις υδατοκαλλιέργειες υποφέρουν πάρα πολύ. Και γι' αυτό έχει σημασία επειδή ανησυχεί όλο και περισσότερο η κοινή γνώμη και οι πολίτες μας, καλό θα είναι να έχουμε ένα ψήφισμα μετά τη συζήτηση αυτή και προτείνω να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη ε, της δεύτερης συνόδου του Μαρτίου ψήφισμα το οποίο θα έρθει να επισφραγίσει τη συζήτηση της Πέμπτης που θα γίνει εδώ στην Ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί κατά της πρότασης. Παρακαλώ. Uważam, że ten parlament Το κοινοβούλιο οφείλει να συζητάει για τους ανθρώπους, όχι για τις υποθέσεις των ζώων. Είναι υποκριτικό. Βεβαίω, ε, τα ζώα υποφέρουν. Υποφέρουν όμως και στα σφαγεία. Τα ζώα δεν πληρώνουν ε, φόρους. Λοιπόν, ας το αφήσουμε το θέμα αυτό κατά μέρος. Ευχαριστώ. Ποιο είναι υπέρ τη πρόταση τη ομάδα των Πρασίνων και τη ομάδα Διευθυντή. Ποιο είναι κατά. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία κατά της πρότασης. Για να κάνουμε ένα έλεγχο για να είμαστε σίγουροι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρόταση. Έτσι λοιπόν, ορίστηκε η περισσία διάταξη να περάσουμε τώρα στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Είχα ζητήσει το λόγο νωρίτερα. Και εγώ βαστού. του άρθρο 11, μέρος 2. και που λέει ότι δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση των κρατών μελών. Η Μάρκο Πάκα άφησε την αίθουσα αφού ψηφίσαμε. Είχαμε λοιπόν ένα τύχημα, συνάδελφος έπεσε. Ήρθαν νοσηλευτές. Δυστυχώς ε, σημειώθηκαν σημαντικά τραύματα, σοβαρά τραύματα. Δεν θυμάμαι ποιο βουλευτής ήταν, Όμω, ε, θα ήθελα όλοι οι βουλευτέ να το έχουν αυτό στο μυαλό του, ε, αδειάζοντα, φεύγοντα από την αίθουσα, να έχουν ο ένας τον άλλον πιο πολύ κατά νου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν το έριξα καθόλου αυτό αν ε, υπήρξε ευθύνη, αν υπήρξε δόλο θα παρέμβουμε. Αν ε, όμως ε, ήταν κάτι μη θελημένο, θα το επαληθεύσω, θα ελέγξω τι συνέβη. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα σήμερα είναι η έκθεση του κύριου Ντάλτον. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου. Έκρης. Όσον αφορά φακέλους, ποινικούς φακέλους. Ζητώ πρώτα απ' όλα από τον κύριο Ντάλτο να λάβει το λόγο ως εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτείται για την καταπολέμηση του εγκλήματος. εγκληματίες ε, μετακινούνται, το έγκλημα εντείνεται. Είναι πιο εύκολο να κρύβονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για υπηκόους τρίτων χωρών. Το έκρηση δεν λειτουργεί αποδοτικά. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν προηγούμενε καταδίκε. Είναι εύκολο για Ευρωπαίου υπηκόου, αλλά όχι για του υπηκόου τρίτων χωρών. Αν κάποιο λοιπόν έχει προηγούμενε καταδίκε, ε, για να εντοπιστούν αυτέ οι καταδίκε, πρέπει να έρθει κανεί σε επαφή με όλα τα κράτη-μέλη, το οποίο σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον. Πρόκειται λοιπόν για ένα κενό, το οποίο σημαίνει λιγότερη ασφάλεια για του Ευρωπαίου. Η έκθεση λοιπόν αυτή κλείνει αυτά τα παραθυράκια. Ευνοούμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων και την διευκολύνουμε για, τον, για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Εν τέλει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν μια συνολική εικόνα κατά τη διενέργεια των καθημερινών τους καθηκόντων. Συμφωνούμε όλοι ότι οι υπηκοοί τρίτων χωρών δεν πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους υπηκόους και δι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνος όλους, όλες τις πολιτικές ομάδες. Μάλιστα αυτό θα αποτελούσε και διάκριση αν κάποιος είχε μια ε, ηθαγένεια τρίτου κράτους. Χρειάζεται επίση να συζητήσουμε το θέμα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ώστε να αποφεύγονται διακρίσει. Με την νομοθεσία αυτή, λοιπόν, κλείνουμε αυτό το παραθυράκι, όπω είπα, και εξασφαλίζεται η ισορροπία και έτσι οι προηγούμενε καταδίκε θα εντοπίζονται εύκολα. Προστατεύουμε επίση τα δεδομένα κατά την ανταλλαγή του. Δεν πρόκειται για κεντρική βάση δεδομένων στην οποία μπαίνει ο καθένα και κάνει ό,τι θέλει. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται με τρόπο ώστε να είναι στην ίδια μοίρα Ευρωπαίοι και άλλοι υπήκοοι. Έτσι, το αποτέλεσμα κάθε έρευνα θα είναι το ίδιο. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη εν τέλει και οι δικαστικέ του αρχέ θα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για να εντοπίζουν προηγούμενε καταδίκε από οποιοδήποτε άλλο κράτο μέλο για να το λάβουν υπόψη του όταν έρχεται η ώρα να δικαστούν αυτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Επίση, θα περιληφθούν και όσοι έχουν διπλή ηθαγένεια, ευρωπαϊκή και τρίτης χώρας. Έτσι κανεί δεν θα κρύβεται παρουσιάζοντα ένα μόνο από τα δύο διαβατηριά του. Επίση, για να ξεκαθαρίσω μερικέ παρεξηγήσει, παρανοήσει στην Άλντε, πρόκειται για προηγούμενε καταδίκε. Άρα, δεν μιλάμε για καταδίκε σε τρίτε χώρε, Μιλάμε για καταδίκε μόνο σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, οι Ευρωπαϊκέ αρχέ θα μπορούν να προβαίνουν σε ανάλυση χαρακτηριστικών με βάση τα εφιστάμενα δεδομένα. Επιπλέον, η συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα γίνεται, αποτυπωμάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο για του υπηκόου τρίτων χωρών όπω για του Ευρωπαίου. Επαναλαμβάνω ότι οι δικαστικέ αρχέ θα έχουν μια πλήρη λοιπόν εικόνα και θα εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα. Ελπίζω ότι θα ψηφίσετε για να μην αφήσουμε χωρίς προστασία τους ε, Ευρωπαίους υπηκόους, για να μην τους αφήσουμε σε δυσμενέστερη μοίρα, ούτε να δώσουμε τη δυνατότητα σε υπηκόους των χωρών να κρύβονται όταν έχουν καταδικαστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ η έκθεση υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ελπίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι μια καλή πρόταση, δεν δημιουργεί διακρίσεις. Να την υποστηρίξουμε, τη συνιστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σα σας καλώ να την υπερψηφίσετε και εσείς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ την κυρία Γιούροβα να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, τον κύριο Ντάλτον, τον εισηγητή και τις αντίστοιχες Προεδρείς του Συμβουλίου για το έργο τους επί των προτάσεων για κανονισμό και οδηγία για το ένα, σύστημα βελτιωμένης ανταλλαγής ε, πληροφοριών ε, ποινικού μητρώου για υπηκόρους τρίτων χωρών. τη ΙΕΝ Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συνομοθέτες ε, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την εξέβρεση μιας αποδεκτής λύσης για όλα τα μέρη. Η Επιτροπή πρότεινε το σύστημα ΕΚΡΙΣ της ΙΕΝ κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι το Νοέμβριο του 2015. Ο στόχος ήταν να κλείσουν ε, τα παραθυράκια στο εφιστάμενο σύστημα για την ανταλλαγή των ε, ποινικών μητρών, δηλαδή στο ΕΚΡΙΣ, έχοντα καλύτερη πρόσβαση για τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών ε, στα ποινικά μητρώα υπηκών τρίτων χωρών. Οι προτάσει συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο του των διαθεσμικών προτεραιοτήτων ε, του 2017 που θα έπρεπε να ελοπιθούν πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Με την αυριανή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο πετυχαίνει αυτό το στόχο. Ως αποτέλεσμα θα πετύχουμε ένα βελτιωμένο σύστημα για την εντελογή ποινικών μητρών που θα συνεισφέρει στο, ε, στον ευρωπαϊκό χώρο Ευρωπαϊκή ελευθερία, ασφαλεια και Δικαιοσύνης. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τι προσπάθειε του να επιλύσει κυρίω δύο ζητήματα. Καταρχήν, τι συνθήκε υπό τι οποίε μπορούν να συμπεριληφθούν τα αποτυπώματα στο σύστημα εκκριστησιέν. Και δεύτερον, την συμπερίληψη των ατόμων με διτή ηθαγένεια, δηλαδή πολιτών Ευρωπαϊκή Ένωση, που επίση έχουν την ηθαγένεια και τρίτη χώρα. Είμαι ικανοποιημένη γιατί θεωρώ ότι βρήκαμε μια ισορροπημένη λύση που να είναι αποδεκτή σε όλα τα μέρη και που θα διασφαλίσει ότι το σύστημα ECRIS της ε, πληρεί τους ε, στόχους του. Το νέο σύστημα θα επιτρέψει να κλείσουν τα παραθυράκια στην ανταλλαγή πληροφοριών για προηγούμενες καταδίκες. Και αυτό θα γίνει βάσει αξιόπιστων πληροφοριών ταυτότητα. και με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως το συμβιβασμό που έχει εξευρεθεί από τους συνομοθέτες και ανυπομονή για την αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλμελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εισηγητή της Αρμόδιας Επιτροπής για το έργο του, το οποίο είναι εξαιρετικό. Αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να ευχαριστήσω για την αγαστή μας συνεργασία. Αυτή είναι μια διαδικασία πληροφορικής που συζητούμε και χρειάζεται οπωσδήποτε ενημέρωση και διεύρυνση. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία ούτε αρκεί, δηλαδή δεν έχουμε ε, αρκετές αντιστοιχίες, ε, ούτε αρκετά ικανοποιητικές και από την άλλη είναι και αρκετά αναποτελεσματικό. Με κόστος μέχρι και 78 εκατομμύρια στα κράτη-μέλη, γιατί είναι τόσο περίπλοκο. Με τη νέα αυτή διαδικασία βέβαια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να δώσουμε 13 εκατομμύρια και άλλα τόσα τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτά είναι λεφτά που θα πιάσουν τόπο, διότι θα βελτιωθεί η διαδικασία και αυτό θα σημάνει ευξημένη ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις προϋποθέσεις για το κράτος δικαίου. Ανταποκρίνεται σε αυτές. Εδώ μπορεί να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι κάνει κάτι για τους πολίτες της. <clears throat> Ε, Ο κύριος ε, Παλτσάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάλτον για το έργο του. Είναι πολύ καλή η έκθεσή του και πάρα πολύ χρήσιμη. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή, μεταξύ των πολιτικών ομάδων εννοώ. Χαίρομαι που σε αντίθεση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση του 2016, Τώρα πρότειναν τα κράτη-μέλη ένα κεντρικό σύστημα. Εμείς πάντα ζητούσαμε ένα κεντρικό σύστημα και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Γιατί αυτό αποκλείει τα τεχνικά προβλήματα και ενδεχόμενες καταχρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε με νυφαλιότητα να ισχυριστούμε ότι ε, η δουλειά μας απέδωσε καρπούς έχουν αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος κατά των κακοποιών. Διότι τα σύνορα του Σέγγεν είναι ανοιχτά και είναι και ανοιχτά για τους εγκληματίες και για τους ε, κακοποιούς. Είναι καλό να μπορούμε να ταυτοποιούμε πολίτες τρίτων κρατών με πολύ λιγότερη ε, γραφειοκρατία. Ε, και η πιο ασφαλής μέθοδος είναι το δακτυλικό αποτύπωμα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν χωράει διαπραγμάτευση αυτή. Το σύστημα ECRIS έχει αποδειχθεί αξιόπιστο. Ε, ακόμα και στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. θα μπορούμε και θα πρέπει να αποθηκεύουμε όλες τις πληροφορίες ε, ε, για τους πολίτες των τρίτων χωρών, τις ίδιες πληροφορίες που συλλέγουμε και αποθηκεύουμε για τους δικούς μας πολίτες. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει την έκθεση αυτή γιατί συνιστά σημαντική και ουσιαστική πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε η κυρία Χέτ για τρία λεπτά. Thank you. Πρόεδρε, φτάνουμε στο τέλος αυτού του μεγάλου ταξιδιού. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμασταν. Ο στόχος ήταν τα πενικά δικαστήρια των κρατών μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί υπηκών τρίτων χωρών. Αυτό είναι καλό. Δεν έχουμε αντίρρηση το σύστημα έκρης να συμβάλλει στο να κλείσουν ορισμένα παραθυράκια. Υπάρχουν βεβαίως δυσκολίες. Για παράδειγμα το Συμβούλιο και η Επιτροπή θέλησαν κάποια στιγμή να τροποποιήσουν το σύστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δημιούργησε προβλήματα σε ό,τι μας αφορά όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ δηλαδή των της ΕΕ των υπηκών τρίτων χρόνων και αυτών που έχουν δύο ηθαγενείς, δύο διαβατήρια. Προβλήματα λοιπόν μη ισότιμης μεταχείρισης. Το σύστημα δυστυχώ επιτρέπει ακόμη τέτοια διακριτική μεταχείριση. Ε, επίσης, το σύστημα δακτυλοσκόπησης και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θέλουμε αντικειμενικά κριτήρια με την Γκουε και τους πράσινους. Κατά τη διάρκεια τώρα των διαπραγματεύσεων, η Κομισιόν έθεσε άλλους διαφορετικούς στόχους όσον αφορά συγκεκριμένα την ανταλλαγή πληροφοριών για προηγούμενες καταδίκες. Εκεί είχαμε προβλήματα λειτουργικής συμβατότητας και τούτο γιατί δεν γνωρίζουμε τα συστήματα όπως λειτουργούν σήμερα. Τώρα, ενώ ψυχλογών οι ακραίοι, δεξιοί θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε πίσω όσον αφορά τις αρχές μας. Σε κάθε περίπτωση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να την χάνουν διακριτική μεταχείρισης ει βάρο του σε σύγκριση με τους ευρωπαίου πολίτε. Ενώ, με άλλα λόγια, ότι αυτό το οποίο προτείνουμε εδώ είναι υπερβολικά αυστηρό. Εν πάση περιπτώσει, προτείνω να απόσχουμε κατόπιν όλων αυτών που ανέφερε. Ευχαριστώ. Η κυρία Στίβεν, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Το έκριση είναι μια τράπεζα δεδομένο όπου τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίε για ε, καταδικασμένου πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προσφέρεται για ανταλλαγή πληροφοριών για αλλοδαπού που έχουν καταδικαστεί. Γι' αυτό Τώρα υπάρχει ένας γολγοθάς γραφειοκρατικός για να μάθει ένα ε, κράτος μέλος ε, εάν έχει καταδικαστεί πολίτης τρίτης χώρας. Άρα 27 διαφορετικά αιτήματα θα πρέπει η δικαιοσύνη να συντάξει και να στείλει σε κάθε κράτος μέλος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η βαριά διαδικασία σχεδόν δεν ακολουθείται. Και ε, με ποινικό μητρό πολίτες τρίτων χωρών γλιτώνουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορεί ένας Βέλγος δικαστής να ενημερωθεί σωστά. Αυτό είναι παράδεκτη έλλειψη. Οι αλλοδαποί που έχουν ποινικό μητρό θα πρέπει να υφίστανται την ίδια σκληρή μεταχείριση όπως και οι Βέλγοι ή άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Με τη σημερινή πρόταση θέλουμε λοιπόν να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών για καταδικασμένους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι δυνατή και να ξέρουμε και σε ποια χώρα της Ένωσης έχουν καταδικαστεί ε, και να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να, να τρέχουν σε αυτή την τράπεζα δεδομένων. Είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόμμα μου, η ΕΝΒΑ, είναι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα ε, για να μπορούμε να ταυτοποιούμε καλύτερα τους πολίτες τρίτων χωρών και τους πολίτες που έχουν διπλή ηθαγένεια. Ε, στηρίζουμε απολύτως λοιπόν αυτή την νομοθετική δέσμη και σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. κυρία Μνίναρ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Στα αγγλικά. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω κατά πρώτον τον κύριο Ντάλτον και τους Κιώδης για το έργο τους επί ενός τεχνικού ευαίσθητου φακελού. Ήταν μακρά η πορεία που μας έφερε όμως σήμερα εδώ Δυστυχώ με λύπη μου σας ανακοινώνω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω, δεν μπορώ να υπερψηφίσω το αποτέλεσμα του τριμερού διαλόγου. Είμαι απογοητευμένη με την απόφαση να συμπεριλάβουμε ανθρώπους με διπλή υπηκότητα στο σύστημα, διότι από την αρχή αυτό ήταν για μας η κόκκινη γραμμή. Ε, για μένα ως τη της Άλτε. Είναι νομίζω ενισχυτικό ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να αποδείξει την αναγκαιότητα ούτε την αναλογικότητα του μέτρου. Το επιχείρημα ήταν υποτίθεται ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να κρυφτούν πίσω από το ευρωπαϊκό τους διαβατήριο. Αυτό είναι αβάσιμο. Ίσα ίσα τώρα δημιουργούμε ανισότητα στη μεταχείριση. Αυτό αποτελεί διάκριση, σαφέστατα. Είναι διαφοροποιημένη η μεταχείριση και με όλο το σεβασμό ε, αυτό αλλοιώνει τα γεγονότα. Δυστυχώ, παραβιάζουμε εδώ θεμελιώδη δικαιώματα, την αξία το δικαίωμα της ισότιμη μεταχείριση, που είναι δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν εγκριθεί ο κανονισμό ως έχει, ω προτείνεται, ένας μεγάλο αριθμός Ευρωπαίων υπηκόων θα την χάνουν μεταχείρισης ως εάν ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών. Γι' αυτό το λόγο και μόνο η πρόταση αυτή δημιουργεί πολίτε δύο ταχυτήτων. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε και καλό και του άλλου να καταψηφίσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φραντ για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μια τράπεζα δεδομένων ε, πανευρωπαϊκή, την οποία εμεί δεν απορρίπτουμε Λίβδιν όπως το PNR που δήλωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν είναι νόμιμο. Στο ΕΚΡΙΣ δεν πρόκειται για μαζική παρακολούθηση, αλλά για συλλογή πληροφοριών ε, για πολίτες που έχουν καταδικαστεί. Αυτό το ε, καθεστώς ισχύει για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατάλογος. Και τώρα θα δημιουργείται ε, και για πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά, εμείς πράσινοι ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τελικά δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Το έκρι για πολίτε τρίτων χωρών, όπως θέλει τώρα να αποφασιστεί και όπως ε, το διαπραγματεύτηκε ο κύριος Ντόλτον παρά την εντολή που του είχαν δώσει οι περισσότεροι συντονιστές δεν οδηγεί σε ίση μεταχείριση των πολιτών των τρίτων χωρών αλλά σε διπλή ανισότητα ενώ για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα δακτυλικά αποτυπώματα συλλέγονται μόνο όταν ε, έχουν ε, συλλεγεί σε κάποια δικαστική διαδικασία. Για τους πολίτες τρίτων χωρών αυτό γίνεται συστηματικά και πρόκειται για άνηση γεωμετρία και μια βάση δεδομένων για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών. Οι άνθρωποι που έχουν διπλή ηθαγένεια δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και κάποιο άλλο κράτος μέλους, συλλέγονται ε, τα στοιχεία τους ε, προληπτικά και καταλήγουν σε δύο βάσεις δεδομένων. Άρα, ορισμένοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο ίσοι από τους άλλους. Και αυτό παραβιάζει την αρχή της διάκρισης με βάση την ηθαγένεια. Ακόμα και αν επί της ουσίας και ε, καταρχήν θα συμφωνούσαμε με το έκρης το αποτέλεσμα μας απογοητεύει. Πρόκειται για συστηματική διάκριση εις βάρος πολιτών τρίτων χωρών και εκείνο με διπλή ηθαγένεια. Ευχαριστώ. Αποσιάζει ο κύριος Φερέιρα. Αν έρθει θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Ράντεφ. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, δεδομένης της τρομοκρατική απειλή, στην, ε, που πλανάται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, η ασφάλεια έχει γίνει πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για μας τους νομοθέτες, που έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι κάθε γωνιά της Ευρώπης παραμένει ασφαλής. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι το σύστημα έκρης Ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουμε την εβδομάδα αυτή. Ένα τέτοιο σύστημα ήδη υπάρχει και καλύπτει τους Ευρωπαίους πελίτες. Όμως ε, η έλλειψη ενός τέτοιου συστήματος που να καλύπτει τους υπηκόους τρίτων χωρών μέχρι τώρα αποτελούσε κενό στην ε, ευρωπαϊκή εσωτερική ασφάλεια. Η πραγματική, αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για τις ε, καταδίκες υπηκών τρίτων χωρών, καταδίκες από ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα σημαίνει ότι κανένας ε, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει της δικαιοσύνης, απλά μετακινούμενος από το ένα κράτος μόνο στο άλλο. Θέλω να είναι ξεκάθαρος η ελευθερία της κυκλοφορίας δεν απαλλάσσει κανέναν από τις ευθύνες του. Όλοι όσοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι Ευρωπαίοι πολίτες είτε όχι, υποχρεούνται να σέβονται την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να ε, υποστούν τις συνέπειες, όποιος και αν είναι. Για ένα λεπτό, η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. για πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως, χώρος ασφάλειας. Όμως, ε, λόγω της ε, μεταναστευτικής και οικονομικής κρίσης ε, δεν έχει μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες από τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Πολλές φορές διάφοροι εγκληματίες, τρομοκράτες επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός της Ευρώπης και ε, δυστυχώς τα μέτρα έρχονται πολύ καθυστερημένα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μία νέα πρόκληση στην ε, Ευρώπη. Ε, το ISIS έχει χάσει το μεγαλύτερο η εδαφική του επικράτεια. Όμως σήμερα προτείνουμε να ενισχύσουμε την τεχνική συνεργασία και να επιτρέψουμε στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταχύς αποφάσεις. Εγώ πιστεύω στους εθνικούς μας θεσμούς στη συνεργασία ε, των εμπειρογνώμων της ασφάλειας και ελπίζω ότι η πολιτική ορθότητα να μην σταθεί εμπόδιο στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις επιλέσεις. Περνάμε στη διαδικασία Κατζιά. Οι τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσουν το λόγο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Στρογεύσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος στην Επιτροπή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και υπέστησα την προσοχή των συναδέλφων σε πολλά ε, προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών και ε, χαίρομαι που ένα από τα παραθυράκια αυτά που υπήρχαν κλείνει σήμερα. Ε, δύο ζητήματα μας ενδιαφέρουν εδώ, να κλείσει επαναλαμβάνω αυτό το παραθυράκι, αλλά και να ενημερωθεί αυτό το σύστημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρουν όσοι ασχολούνται με την ασφάλεια. Ε, ταυτόχρονα καταργούμε και κάποιες διακρίσεις που υπήρχαν. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να υπερψηφίσουμε και με μεγάλη πλειοψηφία αυτό το φάκελο. Δεν είναι εδώ η κυρία Ζωάννα. Θα της δώσουμε το λόγο να έρθει ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, το ΕΚΡΙΣ, είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη εφαρμόζεται για ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με καταδικαστέντες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λοιπόν πάρα πολύ λογικό να επεκταθεί το σύστημα αυτό και για τους πολίτες τρίτων χωρών. δεν είναι δυνατόν αλλοδαποί να έχουν καλύτερη μεταχείριση από τους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης. τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ε, την διπλή υπηκότητα. θα πρέπει να επισημάνω στους συναδέλφους ότι διπλή υπηκότητα σημαίνει διπλά δικαιώματα αλλά και διπλές υποχρεώσεις. δεν μπορεί όταν είσαι πολίτης τρίτης χώρας και υπήκοος ευρωπαϊκής ένωσης απλά να έχει τα θετικά του πολίτη τρίτης χώρας και όχι τις υποχρεώσεις. έχουν λοιπόν τη δυνατότητα όσοι έχουν διπλή υπηκότητα να εγκαταλείψουν την υπηκότητα τρίτου κράτους ή εφόσον έχουν διπλή υπηκότητα θα έχουν και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. επομένως πρέπει να εφαρμοστεί η πρόταση του κυρίου ντάλτον. ευχαριστώ. Ε, Ολοκληρώσαμε εδώ τη διαδικασία Κατσδιάη. Κυρία Γιούροβα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω, να πω ότι συμφωνώ ότι είναι ευαίσθητο και σημαντικό το θέμα της ε, συμπερίληψης ε, των ατόμων με διπλή υπηκότητα για την Κομισιόν. Είναι ζωτικό να συμπεριλάβουμε στο σύστημα έκρηση της ΙΕΝ όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών και αυτούς ε, που είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών κρατών μελών. Διαφορετικά θα αφήσουμε ένα πολύ σημαντικό παραθυράκι και θα υποσκαφθεί ο στόχος της πρότασης αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι οι εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τις διάφορες εθνικότητες για να κρύψουν τις ε, περασμένες καταδίκες τους. Αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί διαφορετική προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών που έχουν μόνο μία υπηκότητα και μεταξύ αυτών που έχουν και την υπηκότητα τρίτης χώρας. Όμως θεωρούμε ότι αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε από αυτές τις υπηκότητες ε, όταν αντιμετωπίζουν δίωξη ή σε άλλες περιπτώσεις όταν το προηγούμενο ποινικό μητρό τους ε, μπορεί να τους θέτει εμπόδια. το χάρη, αν ε, Κάποια άτομα έχουν ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα. Δυνάμει τη ε, της εθνικότητάς τους, ως υπηκότητε της χώρας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διπλή του υπηκότητα όταν, ε, παραδείγματο χάρη, θα κάνουν αίτηση για να εργαστούν με παιδιά σε ένα άλλο κράτο μέλο. Ε, το να αποκλείσουμε αυτού θα σήμαινε ότι τα δεδομένα ταυτότητα κάποιων ανθρώπων με ποινικό μητρό που έχουν την υπηκότητα τρίτη χώρα δεν θα αποθηκεύουν στοχεύεται στο σύστημα ΙΕΝ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τι ε, παρεμβάσει. Θα ήθελα να σα ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε το συμβιβαστικό κείμενο και των δύο προτάσεων. Το νέο σύστημα ανταλλαγή ποινικών μητρών είναι σημαντική συνεισφορά στην ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Χώρου. Του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνη, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντάλτον, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και όλους τους κοιόδης ε, στο φάκελο αυτό, γιατί πράγματι κάναμε πολλή δουλειά, ήταν μακρά η διαδικασία και σας ευχαριστώ όλους ε, για το έργο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Χαβιέρ Νιτοπέρες, ε, ο οποίος είναι συμβουλός μου και τη Χαρίτη Κάρφης, για τις πολλές ώρες εργασίας τους. Τώρα, για τους κατόχους διπλής υπηκότητας, όλες οι νομικές υπηρεσίες μας είπαν ότι δεν αποτελούν διάκριση η συμπερίληψή του Για μένα ήταν κυρία μου προτεραιότητα αυτό. Εργαστήκαμε σκληρά για να τροποποιήσουμε το κείμενο, για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει εισαγωγή διακρίσεων και στου συναδέλφους από την ομάδα Άλντε και τους Πρεσίνου και κυρίως για την κυρία Μίλναρ που τη σέβομαι πάρα πολύ και συνεργαστήκαμε πολύ στενά, να πω ότι πιστεύω ότι κάνετε λάθο. Ε, αν ευθυγραμμίσουμε τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους θα διασφαλίσουμε ότι η μεταχείριση είναι ίδια. Δεν θα υπάρχουν εδώ πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τώρα, κάποιες ομάδες θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την νομοθεσία ως πολιτικό εργαλείο για να πούν στον κόσμο ότι μια ακαδημαϊκή συζήτηση είναι πιο σημαντική από την ευμερία των πολιτών μας. Όμως, λειτουργία ε, των δικαστικό συστημάτων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική εδώ. Ε, τι κάνουμε. Ε, μπορούμε να επιτρέψουμε, αν το αρνηθούμε, στους ε, ανθρώπους με υπηκότητα τρίτης χώρας να αποκρύψουν τις καταδίκες τους. Έτσι λοιπόν, έχουμε το εξή ερώτημα αύριο. Πιστεύετε ότι οι εγκληματίες ε, θα πρέπει να μπορούν να κρύβουν τις καταδίκες τους από τα δικά μας δικαστήρια, αν έχουν υπηκότητα τρίτης χώρας, ενώ οι δικοί μας πολίτες θα μπορούν να το κάνουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, στην έκθεση της κυρίας Σόντροβα, θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Και να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην κυρία Σόντροβα για τέσσερα λεπτά. Sorry for hearing it up, but yeah. it's okay. Συγγνώμη που σας πίεσα λίγο στην Επιτροπή. Κυρία uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Πέρασαν έξι μήνες από τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 18-20 και να είμαστε πάλι εδώ με ένα ενισχυμένο πρόγραμμα. Είχαμε μερικά προβλήματα διότι δεν είχαμε στοιχεία υλοποίηση από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Δεν είχαμε τα δεδομένα, αν θέλετε. Με τη βοήθεια όμω των εμπλεκομένων κατορθώσαμε να εντοπίσουμε του τομεί, τι περιοχέ όπου μπορούμε να βελτιωθούμε. Χαίρομαι, ε, διότι όλες οι πολιτικές ομάδες διατηρήσαν τον σκιώδη συγγητή τους και έτσι διασφαλίσαμε εξαιρετική περαιτέρω συνεργασία. Σα ευχαριστώ όλους. 332 τροπολογίες υποβλήθηκαν και τέσσερις επιτροπές εξέδωσαν γνωμοδοτήσεις. Κατατέθηκαν λοιπόν πολλές ιδέες στο τραπέζι. Ε, παρ' όλα αυτά κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ευρεία πλειοψηφία, μία μόνο ψήφο κατά και μία μόνο αποχή. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να εξασφαλίσει προπολογισμό ενό δισεκατομμυρίου 260 εκατομμυρίων ευρώ που αποδεχθήκαμε, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την χρηματοδότηση των δράσεων 350.000 συμμετεχόντων σε διάρκεια 7 ετών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, διότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα ενσωματώσει και το Σώμα Εθελοντών, το οποίο δρά σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κατεπίγουσες ανάγκες. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Σώμα θα μπορέσει να εκφράσει την αλληλεγγύη μας έναν τρίτων χρόνων με τρόπο απτό. Για να πετύχουμε όμως, το Ευρωπαϊκό Σώμα χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και το λέω αυτό διότι συζητώντας με νέους ανθρώπους συνειδητοποίησα ότι παρά το ότι ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά πράγματα δεν γνωρίζουν τον θεσμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελεγγύης προηγούμενους συμμετέχοντες, ε, προσώπους στα σχολεία. Να διαδώσουμε λοιπόν την ιδέα και να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Η ιδέα επίσης πρέπει να προβληθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε επίσης ε, ημερίδες ενημέρωσης ο σκοπός σε κάθε περίπτωση είναι, όπως είπα, να προβάλλουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, να πείσουμε να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι οργανισμοί, περισσότερες οργανώσεις, περισσότερες ομάδες, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την ποιότητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, να πολλά από τους νέους ανθρώπους, χρειαζόμαστε προγράμματα διαφορετικής φύσης, προγράμματα ποιότητας, δημιουργώντας και χώρο στους συμμετέχοντες για την υλοποίηση του προγράμματος. Ας μην ξεχνούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σχεδιάστηκε από την αρχή ως πρόγραμμα για νέους ανθρώπους. Το πρόγραμμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για άτομα ηλικίας έως 30 ετών. Καταλαβαίνω την επιθυμία ορισμένων να συμμετάσχουν πέρα από αυτήν την ηλικία, όμω ο βασικό στόχο είναι να κινητοποιήσουμε τη νεολαία. Και όταν μιλάμε για νεολαία, δεν μπορούμε να υπερβούμε το όριο των 30. Το πρόγραμμα επίση πρέπει να είναι ανοιχτό σε ανθρώπου με λιγότερε ευκαιρίε. Είμαι πεπισμένη ότι μαζί θέσαμε τα θεμέλια για καλύτερη συνεργασία με το Συμβούλιο. Περιμένουμε πολλά από την υλοποίηση του προγράμματος. Προσβλέπω και στην συνεχή υποστήριξη της Κομισιόν, διότι το Ευρωπαϊκό Σώμα είναι το εφαλτήριο για πολλές σημαντικές δράσεις. Πρέπει μάλιστα να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα αποτελεί συνέργεια με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους και προσβλέπω στην συνέχιση των συζητήσεων ώστε να καταλήξουμε σε μια επιτυχή θετική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς η κυρία Θεοχάρους από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε η σύσταση του ευρωπαϊκού σώματος αλληλεγγύης θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού και θα αναπτύξει το πνεύμα της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού ανάμεσα στους ευρωπαίους νέους. το esc program προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν σε προγράμματα αλληλεγγύης για αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας η σύστασή μα, ωστόσο είναι να μην εφαρμοστεί ω ανώτατο όριο ηλικία στα 30 έτη όσον αφορά τον τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια, για να επιτρέψουμε και σε πιο εμπειρά άτομα να συνδράμουν την προσπάθεια διότι πολλέ φορέ χρειάζεται ειδική κατάκτηση και γνώση πριν την ανάληψη καθηκόντων υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού στις διάφορες πτυχές και για τον λόγο αυτό εμείς εξ ονόματος της επιτροπής ανάπτυξης καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες προκειμένου να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για όλες τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας. οι αποτυχίες των προηγουμένων προγραμμάτων εθελοντικής δράσης της ευρωπαϊκής ένωσης δεν πρέπει να συνεχιστούν. θέλουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης χαιρετίζω τις προτεινόμενες απλουστευμένες διαδικασίες για την ετικέτα ποιότητας για τις συμμετέχουσες οργανώσεις καθώς και την κατοχύρωση των ήδη συμμετεχουσών. γνωρίζω από πρώτο χέρι τα τεράστια ζητήματα με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ελπίζω αυτές να απλουστευτούν. ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να συμμετέχω στη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτό το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι νέο, αλλά μεγαλώνει γρήγορα και οι νέοι στην Ευρώπη ανυπομονούν να συμμετέχουν. Το Ευρωπαϊκό Σώμα αλληλεγγύη. έχει τη δυναμική να γίνει ένα άλλο εμβληματικό πρόγραμμα όπως το Εράσμους. Η ελεγγύη μεταξύ των πολιτών και των κρατών μελών είναι μία από τις αξίες, τις βασικές τις οποίες οικοδομείται η Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης προσφέρει στους νέους ευκαιρίες να βιώσουν αυτή την ελεγγύη και να νιώσουν τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος. Ενυπομονούν να δράξουν τις ευκαιρίες αυτές. 130.000 νέοι έχουν τώρα εγγραφεί στην πρωτοβουλία αυτή. Περίπου 12.000 έχουν ήδη ξεκινήσει στις δραστηριότητές τους στα πλαίσια της ελληνικής. Αυτό που δεικνύει ότι το πρόγραμμα απαντά σε πραγματικό αίτημα επιτόπου. Οι νέοι κάνουν τη διαφορά, υποστηρίζουν άτομα και ολόκληρες κοινότητες που είναι σε ανάγκη. Γι' αυτό τον Ιούνιο του 2018 η Κομισιόν πρότεινε να συνεχίσει και να διευρύνει περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υπό το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θέλουμε να διατηρήσουμε τα κυρία στοιχεία του σημερινού προγράμματο, αλλά να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή μετά το 2020 για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και επιχειρήσει ανθρωπιστική βοήθειας πέρα από τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίες μου για τη μεγάλη αφοσίωση με την οποία η κυρία Σόντροβα και σκιώδη εισηγητές ε, ανέλαβαν αυτό το φάκελο. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την κυρία Θεοχάρου ε, για το έργο τη ω εισηγήτρια στην Επιτροπή Ανάπτυξη, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τις νέες επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Κομισιόν καλωσορίζει την ισχυρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την πρόταση και σημειώνει τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που βλέπω ότι συμφωνούμε σχεδόν σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης και που πρέπει να βρούμε συμφωνία είναι το νέο σκέλος ανθρωπιστικής βοήθειας και η επιθυμία σας να το ανοίξετε σε ανθρώπους όλων των ηλικιών να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί ένα πρόγραμμα για την νεολαία που έχει σχεδιαστεί ακριβώ να προσφέρει ευκαιρίε στη νέα γενιά να επενδύσει στη δική του ανάπτυξη, στι δεξιότητέ του και τα όνειρά του. Και η ιδέα είναι όλε αυτέ οι ευκαιρίε ε, να ομαδοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα. Οι δραστηριότητε του προγράμματο ε, αφορούν ανθρώπου μέχρι 30 έτη για έναν συγκεκριμένο λόγο, για να τους βοηθήσουν ε, στο να να προσαρμοστούν και να κατακτήσουν την ανεξαρτησία τους, αλλά και να μπουν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας και μια εμπειρία αλληλεγγύης. Η ηλικία του 30 βασίζεται σε αποδείξεις, δεν είναι κάτι ευθέρετο. Πέρα από αυτήν την ηλικία, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ουσιαστικά παγιώσει ε, την επαγγελματική και ιδιωτική της ζωή. Ε, Τώρα το να άρουμε αυτό το όριο ηλικία σημαίνει ότι θα φερούσαμε ευκαιρίες για τους νέους και κινδυνεύουμε ε, αντικατάσταση των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που εμπίπτουν ε, στο νέο σκέλος ανθρωπιστικής βοήθειας ε, θα αφορούν μόνο 4.500 από τους 350.000 που θέλουμε να προσφέρουμε κατά τα 7 έτη και μόνο 500 από αυτού ε, θεωρείται ότι θα αναλυφθούν από ανθρώπου ε, πάνω από τα 30. Το να βάλουμε διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητα για ένα τόσο μικρό σκέλο δραστηριοτήτων θα οδηγούσε σε επιπρόσθετο διοικητικό κόστο, δυσανάλογο και θα καθιστούσε το πρόγραμμα πιο πολύπλοκο. Και σίγουρα θα παίκλει αυτού που πρέπει να ωφεληθούν περισσότερο, δηλαδή του νέου. Επομένω, απευθύνω έκκληση σε εσά να διατηρήσουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελληνική σε ένα πραγματικό πρόγραμμα για του νέου, λεχθέντο αυτού. Κομισιόν. Θα ήθελα να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει μαζί σα αμέσω, όπω και το Συμβούλιο. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση και προσφορά μου σε εσά. Είμαι έτοιμο να συνεργαστώ μαζί σα για την επίτευξη μια συμφωνία πριν το τέλο τη σημερινή θητεία. Μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, η μερική συμφωνία πρώτη ανάγνωση έχει ήδη επιτευχθεί για πολλά προγράμματα. Θα ήταν κρίμα αν ε, για αυτό το νέο πρόγραμμα ε, δεν τα καταφέρναμε είμαι σίγουρος ότι ένας καλός συμβεσμός που πετεύχθη μόλις πρόσφατα θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Μία ταχεία συμφωνία θα βοηθούσε την Κομισιόν να κάνει όλες τις προετοιμασίες για να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα πλήρως μπορεί να εφαρμοστεί και αποτελεσματικά από την αρχή του 2021. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη νέα γενιά ότι επενδύουμε σε αυτούς παραμένει προτεραιότητα για μας και ότι θα βάλουμε τη δυνατά μας για να τους βοηθήσουμε να οικοδομήσουν μια καλύτερη Ευρώπη για το μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Βράτσιτς. και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φόλκιν για ένα λεπτό από την Επιτροπή Προπολογισμών. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί νέοι, ε, που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Ήδη από το 2016 Χάρη στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, δίνεται ευκαιρία σε νέους να συνεισφέρουν ε, πανευρωπαϊκά στην κοινωνία με εθελοντισμό, άσκηση ή και εργασία για να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους στην πράξη είναι κάτι παραπάνω από ένα σώμα αλληλεγγύης. Ε, δημιουργεί ταυτότητα και αξίες πέρα από σύνορα. Και αυτό είναι σημαντικό. Στην επόμενη περίοδο να δώσουμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τους νέους για να στηρίξουμε το πρόγραμμα αυτό. Αυτό θέλουμε. Και τώρα τι χρειαζόμαστε. Περισσότερους νέους Ευρωπαίους και νέες Ευρωπαίες που να βιώνουν τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Γι' αυτό χαίρομαι που οι νέοι βγαίνουν στο δρόμο και διαδηλώνουν για περισσότερη προστασία του κλίματος, κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της ελευθερίας. Ε, οι νέοι λοιπόν δεν είναι ρομπότ, ε, είναι σκεπτόμενοι νέοι και με το πρόγραμμα αυτό ε, υποστηρίζουμε τους νέους και χαίρομαι που θέλουμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλετιτς για ένα λεπτό, εξ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με μικρόφωνο παρακαλώ. κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, επίσης να συγχαρώ τους εισηγητές Πολύ συχνά οι νέοι ε, ρωτούν πώς μπορώ να προσφέρω, ε, να κάνω κάτι εθελοντικά, γιατί έχω ελεύθερο χρόνο. Είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, ε, είτε για άλλες μορφές ανθρωπιστικής δράσης. Στον προϋπολογισμό 2021 έως 2000 27 έχουμε αυξήσει τα κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό 1,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου τριπλάσια πλέον τα κονδύλια σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να απλουστευτούν οι κανόνες επιλεξιμότητας και συμμετοχής καθώς επίσης και να απλουστευτεί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το κόστος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα πρέπει να αποζημιώνονται για όλες τις δαπάνες τις οποίες έχουν υποβληθεί. Ε, είναι σημαντικό να είναι νέοι, το ακούσαμε αυτό ήδη, αλλά ιδιαίτερα τους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο κύριος Τρογιάσκη για 1,5 λεπτό εξ ονόματος της ε, Επιτροπής του. Το Ευρωπαϊκό Σώμα είναι προσφορά προς τους νέους. Τους νέους της Ευρώπης. Έχουμε πείρα από άλλα προγράμματα και πιστεύω ότι η εξέλιξη αυτή είναι θετική. Με τη νέα πρόταση μειώνουμε την γραφειοκρατία, επιταχύνουμε τις διαδικασίες, εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη διαφάνεια το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο. Προσοχή όμως δύο σημαντικά θέματα. Το πρόγραμμα πρέπει να προβληθεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρέπει να προβληθεί στους νέους ανθρώπους κυρίως, να καταλάβουν ποιες είναι οι προοπτικές που τους ανοίγονται και χαίρομαι που ήδη έχουμε δεσμεύσει προπολογισμό για την επόμενη ετία. Βεβαίω το πιο δύσκολο είναι η εφαρμογή. Η πρόκληση είναι η εφαρμογή στην πράξη. Θα δούμε λοιπόν αν θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Με την ευκαιρία συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έχουμε πολλές, έχουμε περίπου 300 ε, τροπολογίες. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα να πάρει το λόγο για 3,5 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε κυρία Σόντροβα και κύριοι και ηγητές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τι θέλουμε να στείλουμε ως μηνύματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ότι είναι πολύ ισχυρό το θέμα της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της ελεγγύης και αυτό θα πρέπει να είναι ένα σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για την νέα γενιά. Και στην ε, συνέχεια ότι για τα επόμενα 7 έτη σταθεροποιούμε αυτή την εμπειρία που έχει ξεκινήσει ήδη και ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, θα συνεχιστεί, γιατί δείχνουν συμμετέχει σε αυτό 20.000 νέοι. Θέλουμε να είμαστε πιο τολμηροί με την ευριανή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, εγώ όμως και όδηση κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος, γιατί θα δημιουργήσουμε ένα σταθερό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζω οι υπουργοί να δεχτούν την πρόταση του Κοινοβουλίου και ως προς τον προϋπολογισμό. Σχεδόν ε, για το σύνολο του 86% του προϋπολογισμού θα αφορά την ελληνική και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για νέους 18-30 και θα έχουμε και ένα μέρος την εργασία, αλλά πάντοτε θα είναι μη κερδοσκοπική δραστηριότητα και ένα 6% για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ε, πρόκειται για ένα πολιτικό ε, μήνυμα που θα πρέπει πραγματικά να το φυγηθούμε στους νέους που δεν το γνωρίζουν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το εξής. Συμβολικά αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία εγώ θέλω ε, να υπενθυμίσω ότι μετά από ένα τρομερό σεισμό είχαμε ε, ένα πυρήνα νέων που προέρχονταν από 12 χώρες. Επάνω από 70.000 ε, άνθρωποι έχουν εγγραφτεί, 7.000 επιτρέπουν στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, στη διαφύλαξη πολιτικής κοινωνίας κτλ. Είναι σημαντικό ότι έχουμε κονδύλια πάνω από ένα δισεκατομμύριο για την επόμενη επταετία και έτσι επιβεβαιώνεται αυτή η θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και για να απαντήσουμε κυρίως στις ανάγκες της κοινωνίας ε, και των κοινοτήτων. Ε, δίνοντας ε, φυσικά και έμφαση ε, στους λιγότερο ευνοημένους. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ε, μικρότερες ευκαιρίες, που μπορεί να έχουν και δυσκολίες στο σχολείο ή μπορεί να προέρχονται από μεταναστευτικό background. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πτυχές. Καταρχήν, η ευρωπαϊκή διάσταση της εμπειρίας. Ε, όλες αυτές ε, οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ε, έναν διακρατικό χαρακτήρα και θα πρέπει να υποστηρίζουμε και την αναγκαιότητα να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτός ο διακρατικός χαρακτήρας και το γεγονός ότι έχουμε περιλάβει και κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά πάντοτε για μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες και θα πρέπει να υπάρχει και ένα διαφοροποιημένο σήμα ποιότητα Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια νέα εμπειρία όπου συλλέγονται τα καλύτερα διδάγματα του παρελθόντος αλλά και τη βούληση να οικοδομήσουμε μια ε, ηθαγένεια από τα κάτω. Μιλήσαμε σήμερα για τη θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρώπης, για την πολιτική ολοκλήρωση και για την οικοδόμηση διαδικασίας συνεργού συμμετοχής των πολιτών. Ευχαριστώ. Κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με την εκδοχή του ως ενιαία θηρίδα που συνενώνει όλες τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε προγράμματα αλληλεγγύης είναι μια πραγματικότητα για την οποία θα σταθούμε περήφανοι σε πολύ λίγα χρόνια. Μια σπουδαία ιδέα όπως ήταν και το πρόγραμμα Εράσμους γιατί εξισώνει τις ε, δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης στα προβλήματα στα προγράμματα μάλλον, και έτσι θα γίνει καλύτερη αξιολόγηση και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για να δούμε ε, και πώς ε, αποδίδει. Συστηματικά λοιπόν οι πιο ευγενείς αξίες της Ένωσης γίνονται πραγματικότητα. Οι νέοι μας θα συνεισφέρουν στη συνοχή της κοινωνίας μας, θα βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα γνωρίζουν πραγματικότητες ε, που θα τους κάνουν να είναι πιο συνειδητοποιημένοι, πιο αλληλέγγυοι και θα εμβολιαστούν κατά στερεοτύπων και ε, προκαταλήψεων. Έτσι, αυτό θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι πολίτες και να μπορούν να βρουν και καλύτερη δουλειά. Και πιστεύω λοιπόν θα πρέπει η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός να ενισχυθούν, να συγχωνευθούν και να υπάρχουν περισσότεροι πόροι. Και θα πρέπει να δίνεται και κάποια πιστοποίηση στους συμμετέχοντες και συμμετέχοντες να είναι και οι συνοδοί ε, που υλοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Είναι σημαντικός ο ρόλος τους για να ε, πάνε όλα καλά. Και εδώ πρόκειται για διπλή αλληλεγγύη προς τους τελικούς αποδέκτες του προγράμματος και προς τους νέους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Τρούπελ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νέο πρόγραμμα ε, Εράσμου Σώμα Αλληλεγγύης, έχει ε, μεγάλες δυνατότητες να δίνει άλλη μια ιστορία επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει αίτημα για μεγαλύτερη και περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται κυρίως για νέους ηλικίας 18 με 30 ετών που θέλουν να προσφέρουν στο θέατρο, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στο περιβάλλον, στην κλιματική πολιτική, παντού όπου υπάρχουν εθελοντικές ενώσεις ή όπου έχουν και οι ίδιοι ιδέες τι μπορούν να προσφέρουν και να κάνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαθαίνουν γλώσσες, μαθαίνουν άλλες χώρες, γνωρίζουν άλλες χώρες, γνωρίζουν ε, να συμπονούν τους άλλους, την συνέστηση και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουν και κάτι για τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους. Πραγματικά είναι αμοιβαία επωφελής αυτή η κατάσταση. Και τώρα επιτέλους και ευτυχώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα αυτό που ήταν 375 εκατομμύρια να ε, πολλαπλασιαστεί ο προπολογισμό και να φτάσει στα 1,2 δισεκατομμύρια. Άρα υπάρχει πολιτική βούληση σαφής να κάνουμε περισσότερα για τους νέους και για τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και να κατανοούν όλοι ότι έχει νόημα να αγωνίζεσαι για τους άλλους ανθρώπους στους Δήμους και κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Ένωση είναι θετική και η Ένωση είναι αλληλέγγυα. Είναι πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μόνο εργαλειακά και κατ' το πρόγραμμα φτιάχτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η ίδια η έννοια της αλληλεγγύης να διαστρεβλώνεται. θεσμοθετεί μια επικίνδυνη σύνδεση μεταξύ του εθελοντισμού και της απασχολησιμότητας ενώ τη της ουσίας προσπαθεί να επιβάλλει και καλυμμένη εργασία προωθώντας ταυτόχρονα και τη συμμετοχή κερδοσκοπικών εταιριών σε αυτό. στόχοι του προγράμματος αλληλεγγύη δεν μπορούν να είναι η επιχειρηματικότητα τα κέρδη και η επισφαλής εργασία των νέων. ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να ενισχύει την κοινή αξία της αλληλεγγύης και όχι να οδηγεί στην αποδόμηση του περιεχομένου της να ενεργοποιεί τους πολίτες και να βοηθάει τους νέους στην προσωπική τους ανάπτυξη και όχι να ενισχύει τα κέρδη των πολυεθνικών. το ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης αγαπητοί συνάδελφοι όπως συγκροτείται αποτελεί έναν ακόμα ιδεολογικό και πολιτικό μηχανισμό υπό τον έλεγχο τη νεοφιλελεύθερη ευρωπαϊκή ένωση. η σημερινή ευρωπαϊκή ένωση έχει αποδειχθεί ότι αδυνατεί να απαντήσει στι πραγματικέ ανάγκε στι ανάγκε των νέων για μόρφωση για δουλειά για αξιοπρέπεια. αδυνατεί να αντιμετωπίσει τι τεράστιε οικονομικέ και ανθρωπιστικέ κρίσει που γεννούν οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ τη πολιτικέ οι οποίε πρέπει να ανατραπούν και όχι να αντιμετωπιστούν με αυτά τα μπαλώματα που συζητάμε σήμερα. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Έθεριτς ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και τι, πώς ήταν ε, μια έναρξη της εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς ένα ολοκένουργιο πολύ ακριβό πρόγραμμα. Τι ωραία που επιστρέφουμε μου αρέσει ότι τώρα οικοδομείται πολιτική ε, με αυτόν τον τρόπο. Είναι εξαιρετική ιδέα. Τι έχουμε εδώ, το Big ε, Brother και ε, έχει ντυθεί με στολή έτσι λοιπόν ότι επιτρέπεται να δώσετε ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια ευρώ σε καιρούς που λέμε ότι όλοι πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας και αυτά τα χρήματα πάνε σε πολύ ωραία εθελοντικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να μάθει κανείς να είναι λιλέγγυο. Είμαστε όλοι πολύ καλοί Ευρωπαίοι που εργαζόμαστε από κοινού και ε, ακόμη και ο, ο πρόεδρος ήταν υπέρ. Όμως είναι πολιτικό το πρόγραμμα αυτό. Ε, διασυνορική ελληνική. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά ε, υπάρχουν φιλανθρωπικά ιδρύματα που μπορείτε να προσφέρετε την εργασία σας και κάνουν πολλή δουλειά χωρί να υπάρχει και πολιτική σκοπιά. Όπω είπαν και άλλοι ομιλητέ, αυτό είναι ένα ακόμη Εράσμου. Ναι, ένα ακόμη Εράσμου, ένα ακόμη πρόγραμμα όπου κάτι που είναι καλό στην ε, εκπαίδευση τον τίνουμε με προπαγάνδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο μεγάλο βαθμό που αδυνατούμε να δούμε από τι αποτελείται. Ε, μία τέτοια ιδέα είναι ακριβώ το είδο τη ιδέα ε, που ε, κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν γιατί προσπαθείτε να χειραγωγήσετε τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν θέλετε τους ε, μεγαλύτερου ηλικία. Θέλετε να χειραγωγήσετε τα μυαλά των νέων. Ε, όμως ε, πραγματικά πολύ ωραία έναρξη για την εβδομάδα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Δέχεστε μπλε κάρτα από τη συνάδελφο Γκραπίνη. Παρακαλώ κυρία Γκραπίνη. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, προσπαθήσατε ε, να καταφερθείτε ε, απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. Πολύ ωραία μας τα είπατε, όμως εσείς ε, τι εννοείτε με τον όρο αλληλεγγύη, πιστεύετε, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη και μας είπατε ότι ανησυχεί τους ανθρώπους αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ανησυχεί τους ανθρώπους, είναι ένα πολύ καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα το οποίο θέλει να εκπαιδεύσει τους νέους όσο σε Αυτό το σώμα παρακαλώ να μου απαντήσετε. Σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι η ελεγγύη είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοείτε εσεί. Ε, η αλληλεγγύη που βασίζεται στο πλαίσιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ όλων εμά ε, Εγώ ε, θα ήθελα να δω την πραγματική χρήση του όρου ελληνικής, δηλαδή όταν ε, ε, έχουμε δύσκολες στιγμές και πρέπει να συνεργαστούμε. Όμως αυτού του είδους η ελληνική απλώς καταγγέλει και αρνείται την ατομικότητα, τα έθνη, κράτη και όλα όσα αποτέλεσαν μεγαλύτερα στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό η ευρωπαϊκή ένωση παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ενάντια στους λαούς επιστρατεύοντας βομβαρδισμούς εμπορικούς πολέμους δασμούς κυρώσεις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απειλές το ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης αποτελεί ένα ακόμα αντιδραστικό πολυεργαλείο υποστήριξης των πολυπλόκαμων στρατιωτικών δομών της ευρωπαϊκής ένωσης όπως η πεσκο. πρόκειται για ένα σώμα ανέργων όλων αυτών που κατά εκατομμύρια προκαλεί η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεών της που θα περιμαζεύουν τους νεκρούς τους πρόσφυγες και τα συντρίμια των υπερελεστικών επεμβάσεων της ευρωπαϊκής ένωσης και των συμμάχων της επίσης. από χώρα σε χώρα ακόμα και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης θα πηγαίνουν για να μαζέψουν πιστοποιητικά εθελοντισμού και ολιγόμενης μαθητείας με χαρτζηλίκι ίσα ίσα για τα έξοδά τους με εργολάβους μκο και επιχειρήσεις. με ένα σπάρο λοιπόν πολλά τριγώνια υπερελιστικές επεμβάσεις διείσδυση ευρωμονοπωλίων επέκταση των εργασιακών σχέσεων γαλέρας ανακύκλωση της ανεργίας εμπόριο δίθεν αλληλεγγύης μονάζιγα όλα για το μεγάλο κεφάλαιο. οι νέοι εργαζόμενοι με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα μπορούν να δώσουν απάντηση στα υπερελεστικά σχέδια και στην εργασιακή ζούγκλα. Ευχαριστώ κύριο Γκερέρο Σαλόμ. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ω εισηγητή, μόνιμο εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαιρετίζω αυτή την νομοθεσία για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που έρχεται να ενταχθεί στην ανθρωπιστική πρωτοβουλία που υπάρχει ήδη από το 2014. Προσωπικά πιστεύω ότι ενώνονται εδώ ή συναντώνται δύο πεδία. Από τη μια έχουμε την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανθρωπιστικές κρίσεις, οι οποίες αυξάνονται και πληθύνονται ανά τον κόσμο. Και οι περισσότερες είναι ανθρωπογενείς μετά από πολέμους, συγκρούσεις κλπ. Αλλά όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι είναι απορία της κλιματικής αλλαγής, ξηρασίες ε, σε πολλά μέρη του κόσμου, ε, πλημμύρες, ε, πυρκαγιές, τυφώνες, κυκλώνες και από την άλλη ε, ε, θα πρέπει να οικοδομηθεί η ε, έννοια του ανήκειν, της αλληλεγγύης για τους νέους και τους όχι τόσο νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να επεμβαίνουν για να απαλύνουν λίγο τα δεινά και τον πόνο εκεί που χρειάζεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Άκουγα προηγουμένως να γίνεται λόγος για εράσμους και έτσι με τρόπο περιφρονητικό. Το Εράσμο είναι από τα καλύτερα προγράμματα και οικοδομήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο δόμος δεν είναι Εράσμο. Το Εράσμο είναι υπέρ των νέων που ε, μορφώνονται. Αυτό είναι αλληλεγγύη των νέων προς τους άλλους που έχουν ανάγκη και είναι μεγάλη διαφορά. Καθόλου ευκαταφρόνητη, απόλυτη διαφορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ward για ένα λεπτό παρακαλώ. το Σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης στην ουσία του αντιπροσωπεύει τις ίδιες τις αρχές και αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ειρνευτικό πρόγραμμα που επενδύει στο δυναμικό των νέων πολιτών. Εγώ υποστηρίζω την πρωτοβουλία αυτή και χαίρομαι πολύ ε, για την έκθεση όπως προέκυψε από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ζήτησα αύξηση του προπολογισμού έτσι ώστε το πρόγραμμα να ανοίξει για όλους τους ε, νέους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες το να μπορεί να προσφέρεσαι ως εθελοντή και ως νέος έχει πολλά ωφέλη. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Λεγγύη θα δώσει ευκαιρίες ε, για νέους ηλικίας 17 με 30 ετών για να βοηθούν ε, ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αποκτώντας προσόντα και δεξιότητες, αλλά ακόμα και αυτοπεποίθηση και ταυτότητα. Ως Ευρωβουλευτής από το Ηνωμένο Βασίλειο λυπούμε που οι νέοι από την εκλογική μου περιφέρεια μπορεί να στερηθούν αυτό το φανταστικό πρόγραμμα λόγω του Brexit. Τώρα που τόσο ε, ε, πολλοί νέοι αισθάνονται απογοητευμένοι από την πολιτική, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να τους εμφυσίσει αυτές τις ιδέες και τις αρχές και να τους ενισχύσει το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. Είναι μια ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Είναι πολλές ε, οι ευκαιρίες και τα ωφέλη που μπορεί να χάσει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από ε, ένα δημοψήφισμα το 2016 όπου ψήφισαν κάποιοι πικραμένοι ηλικιωμένοι για λόγους του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Νέκοφ ότι τον Ευρωπαϊκό Σώμα θα είναι μια καλή εξέλιξη τα επόμενα, τα επόμενη Όμως, υπάρχουν δύο άλλα πράγματα. Να φροντίσουμε πρώτον ότι υπάρχει ικανός προπολογισμό. έτσι ώστε περισσότεροι νέοι να μπορέσουν να εκφράσουν τον εθελοντισμό τους και να είναι χρήσιμοι. Επίσης να φροντίσουμε να είναι προσβάσιμο από όλους τους νέους, ανεξαρτήτως προέλευσης, ε, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, να συμμετάσχουν και άνθρωποι φτωχοί από απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι είναι σε χειροτερή μοίρα. Αυτό θα κρίνει εν τέλει την επιτυχία ή όχι του προγράμματος. Επίσης, ε, πιστεύω ότι το πρόγραμμα θα βάλει και μια τάξη στα της χώρας μου, θα οδηγήσει στην δημιουργία αντίστοιχης νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Catch Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο της Επιτροπής Πολιτισμού ορίζει την ελληνική ως την έννοια της υπευθυνότητας απέναντι όλο, από όλους απέναντι σε όλους και εκφράζει το κοινό του καλό που εκφράζεται μέσω ε, συγκεκριμένων δράσεων χωρίς αντάλλαγμα. Με το Ευρωπαϊκό Σώμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προωθεί την ελληνική ως αξία μέσω του εθελοντισμού και ταυτόχρονα αυξάνει τη συμμετοχή των νέων ε, για να συνεισφέρει ε, το θέμα της αλληλεγγύης, της παγίωσης της δημοκρατίας, ε, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην Ένωση και στο εξωτερικό. Οι στόχοι αυτοί μας βρίσκουν σύμφωνους μέσω με σε ό,τι αφορά το να συμπεριληφθούν και οι νέοι με ανεπηρίες και επίσης κατά τη διάρκεια του εθελοντισμού να προσφέρονται δυνατότητες εκμάθησης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητε αυτές σε μελλοντική εργασία. Οι νέοι λοιπόν θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν μέσω δραστηριοτήτων εθελοντισμού, στάζ και εργασία σε τέτοια προγράμματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαριάς ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη πραγματικά είναι σημαντικές αξίες στη σύγχρονη κοινωνία. το θέμα είναι όμως ότι παρατηρώντας την πρόταση για το περίφημο ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι διότι ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία γίνεται χωρίς αμοιβή. εδώ βλέπουμε ότι θα διατεθούν ένα δισεκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον περίφημο εθελοντισμό. είναι εθελοντισμός με αμοιβή δηλαδή δεύτερον είναι εθελοντισμός στη βάση της αλληλεγγύης; πολύ το αμφισβητώ διότι έχουμε δει το πώς έχουν δράσει οι περίφημες μη κοιο σε σχέση με τη στήριξη για το προσφυγικό είδαμε ένα μεγάλο πάρτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες. επομένως αξιοποιείται η περίπτωση του εθελοντισμού της αλληλεγγύης στην πράξη για να συνεχιστεί το περίφημο πάρτι το οποίο γίνεται στον τομέα του προσφυγικού του μεταναστευτικού και άλλων δράσεων της κοινωνίας και βέβαια να συγκαλυφθεί το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. αν θέλουμε να πάρουμε μέτρα ας δοθούν αυτά τα χρήματα υπέρ της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή και παρακαλούμε τον Επίτροπο κύριο Ναυράσης να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ καλό που ε, αισθανόμαστε την ευρεία στήριξη για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ήταν μια πρωτοβουλία πολύ επιτυχής. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ρυθμό της, πρέπει να επιταχύνουμε και να αρχίσουμε τους τριμερείς διαλόγους, έτσι ώστε πραγματικά να διατηρήσουμε αυτή την επιτυχία και για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήθελα και πάλι να σας εκφράσω και να σας δηλώσω την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσουν το συντομότερο τριμερείς διάλογοι και σας καλώ να είστε εταίροι μας εκεί και να είναι μια μόνιμη και διαρκής αυτή η επιτυχία. Ευχαριστώ την κυρία Σόιντροβα για την έκθεσή της. Και ήθελα πραγματικά να σας επενέσω για το έργο σας, αλλά και για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για τη συζήτηση αυτή που νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ γόνιμη σχεδόν συμφωνούμε απολύτως και το εκτιμώ αυτό. Και πιστεύω ότι οι αλλαγές που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βελτιώσουν το πρόγραμμα και ελπίζω να τις δεχτεί και το Συμβούλιο και να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία. Όλοι θέλουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να προσφέρει ευκαιρίες ε, στους νέους εθελοντές ε, υψηλής ποιότητας. και να εξακολουθούν να συμμετέχουν ε, εθελοντικά οι προηγούμενοι συμμετέχοντες. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μία αρχή για εκατομμύρια νέους για να μπουν σε νέους αγώνες, ε, σε νέες εμπειρίες και βιώματα και να αποκτήσουν νέες γνώσεις. Ελπίζω η αλληλεγγύη να μην είναι μόνο ε, κάτι το οποίο ε, θα αφυπνήσει και θα κάνει τους ε, αποδέκτες να συνειδητοποιήσουν όλες αυτές τις αξίες, αλλά και για τους εθελοντές. Η αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να θεωρείται είδος πολυτελείας στην κοινωνία μας, αλλά ως κάτι που ο καθένας μας θα έπρεπε να προσπαθεί να εντάξει στη ζωή του. Αυτό το πρόγραμμα πραγματικά μας φέρνει πιο κοντά στην υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας σας. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτησή μας και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η κοινή συζήτηση ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, έχουμε την έκθεση της κυρίας Νίμπλερ ε, πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και έκθεση της κυρίας Ρέντα, Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Τεχνολογικό και Ερευνητικό Κέντρο Εκανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Συντονισμού. Έχει έρθει και ο Επίτροπος για να περάσουμε στη συζήτηση. Για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Επίτροπε, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα καταρχά να σας ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που είχαμε με όλους τους κοιόδης ηγητέ από τις πολιτικές ομάδες, αλλά και την εντατική συνεργασία στον τριμερή διάλογο που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψυγεία, καφετιέρες, ε, ενεργειακά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ε, δίκτυα συγκοινωνιών, τα πάντα θα είναι στο μέλλον συνδεδεμένα μεταξύ του. Τι σημαίνει αυτό ότι η ασφάλεια στον χώρο είναι από τις ύψιστες πολιτικές προτεραιότητες και οφείλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να θυμάστε πριν από δύο χρόνια ε, είχαμε μια μεγάλη ε, κυβερνοεπίθεση πάνω από 200.000 ε, υπολογιστές και συστήματα στο Ενωμένο Βασίλειο τα νοσοκομεία. Στη Γερμανία στόχοι ήτανε ε, οι ε, πίνακες με τα δρομολόγια των τρένων στους σταθμούς και ε, στην Ισπανία ορισμένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών παρέλυσαν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια πανευρωπαϊκή επίθεση, επίθεση, μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες. Και καλά θα κάνουμε εμείς Ευρωπαίοι να προετοιμαστούμε για τέτοιου είδους επιθέσεις. Γνωρίζοντας λοιπόν όσα έγιναν τα περασμένα χρόνια και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά οπλισμένοι πλέον. Υπάρχει μια στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ευρωπαϊκή στρατηγική. Πριν από λίγα χρόνια εγκρίναμε την οδηγία για τις κρίσιμες υποδομές. Αύριο θα εγκρίνουμε την αντίστοιχη πράξη και θα διασυνδέσουμε τα κέντρα δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Ε, αυτή είναι νομίζω η σωστή απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις. Περί τίνος πρόκειται σε αυτή την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αφενός, να ενισχύσουμε την ΕΝΙΣΑ, τον αντίστοιχο οργανισμό που έχουμε και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια θαραλέα πρόταση. Αυτός ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ πρέπει να ενισχυθεί και ως προς το προσωπικό αλλά και προς τους οικονομικούς πόρους του. Και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δώσει και άλλες αρμοδιότητες Θέλαμε να το κάνουμε στην Ενίσα και αυτό ήταν από τα σημεία τριβή στη συζήτηση που είχαμε με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να έχουμε ισχυρές ε, αρμοδιότητες και κέντρα εθνικά αλλά για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ σημαντική ενίσχυση του οργανισμού μας, Ενίσα και να μην είναι απλώς ένα κέντρο συντονισμού των Εθνικών Κέντρων Ασφαλείας, αλλά να έχει και ίδιες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση. Στην Ευρώπη θέλουμε ένα ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο πιστοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό και τεράστιο πλεονέκτημα και για τις δικές μας εταιρείε. Δηλαδή κάποιο να έχει πιστοποίηση όχι μόνο σε μια χώρα, αλλά ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας το Κοινοβούλιο λοιπόν ήταν σημαντικό να έχουμε επίπεδα ασφαλείας για τις έξυπνες συσκευές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Και επίσης για αυτές τις έξυπνες συσκευές θα πρέπει να δίνουμε πληροφορίες, προϊόντος, οδηγίες στους καταναλωτές. Θα πρέπει να ξέρει ο πολίτης αν είναι ασφαλής η συσκευή του και να γνωρίζει πώς μπορεί να ε, ρυθμίζει ε, την ασφάλεια της συσκευή. Όλα αυτά θα τα δούμε στο τριμερή ε, διάλογο και ελήφθησαν υπόψη μάλλον ήδη. Εγώ θα ήθελα να είχαμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω για τις κρίσιμες υποδομές ας πούμε να υπάρχει ένα υποχρεωτικό πλαίσιο πιστοποίησης. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε ένα καλό συμβιβασμό. Θα κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενίσα, με ένα πρόγραμμα ετήσιο θα πρέπει να κάνουν μελέτες για το αν χρειάζεται ένα υποχρεωτικό τέτοιο πλαίσιο όπως το ζητούσαμε. Πάση περιπτώσει, ένα πρώτο βήμα είναι σημαντικό, τα επόμενα θα ακολουθήσουν. Τελειώνω, Πρόεδρε. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κρισιμότατο θέμα, ιδιαίτερα για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι ε, που θα προχωρήσουμε γρήγορα στις διαβουλεύσεις και στις διαπραγματεύσεις ε, μάλλον που το κάναμε ήδη, συγγνώμη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και αύριο θα ψηφίσουμε, ελπίζω, με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Και Ρέντα, τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε Άντσεπ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε την πρόταση για την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλεια στην βιομηχανία και την ίδρυση ενό κέντρου τεχνογνωσίας καθώς και τη δημιουργία εθνικών κέντρων συντονισμού. Συντονίζοντα την προστασία στον κυβερνοχώρο, το κέντρο, το νέο κέντρο συμπληρώνει το έργο του ΕΝΙΖΑ και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε απλώς να αγοράσουμε ένα προϊόν προστασίας και τέλος, η προσπάθεια σημαίνει συνεχή προσπάθεια εναντί διαρκών απειλών. Χρειάζεται η υποδομή μας, τα συστήματά μας να γίνουν πιο ασφαλή. Η κυβερνοασφάλεια είναι λοιπόν διαδικασία, είναι διαρκής διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος. Όμως δεν αρκεί να έχουμε ασφαλή προϊόντα αν δεν έχουμε ασφαλείς υποδομές. Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πλεονέκτημα η κατανομή της τεχνογνωσίας στην Ευρώπη. Πρέπει να ανταλλάξουμε γνώσεις, εμπειρίες στο πλαίσιο ενός νέου οικοσυστήματος κυβέρνου Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη πρέπει και αυτοί να προσπαθήσουν μαζί μας, μαζί με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με τους κατασκευαστές ε, συσκευών για τους καταναλωτές και να συνεργαστούμε και με τους ε, καλόβουλους hacker. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δημορφώσουμε το μέλλον της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Η διανομή της τεχνογνωσίας θα είναι πλεονέκτημα, αλλά θα είναι και πρόκληση. Χρειάζεται συντονισμό. Για αυτούς τους λόγους πάντως θα ενθαρρύνουμε συνεργατικά σχέδια και την επένδυση σε κοινού πόρους. Υπάρχει ζήτηση για εμπειρογνώμονες Μάλιστα έχουμε έλλειμμα εκεί και οι εταιρείε μας δεν πρέπει να υποτιμήσουν τις ανάγκες αυτές. Χρειάζεται λοιπόν η δημιουργία και του απαραίτητου εργατικού προσωπικού που θα υποστηρίξει την τεχνογνωσία στο διαδίκτυο. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητα, αλλά είναι και υπέρ τη ισότητα. Οι συνάδελφοι του περασμένου μήνε και χρόνια έκαναν μεγάλη προσπάθεια, τράβηξαν την προσοχή του κοινού στο πρόβλημα και στις πιθανές επιπτώσεις από την τεχνολογία της πληροφορικής. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον διάλογο αυτόν εν ώψη της ανάγκης προστασίας της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο. Πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον, να δούμε τους μελλοντικού κινδύνους. Δεν έχει νόημα να περιορίσουμε την αντίδρασή μα. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τι κοινωνικέ επιστήμε. Οι κοινωνικοί επιστήμονε πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί. Η Επιτροπή Ήτρε κατέληξε σε μια ισορροπημένη, θα έλεγα, γνωμοδότηση. Και όλα αυτά υπέρ τη δημοκρατία, του κράτου δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτέ τι τεχνολογίε και να θυμάμαστε και την συνθήκη. Όταν η συζήτηση έρχεται και στις στρατιωτικέ εφαρμογέ. Υποστηρίζω λοιπόν τι τροπολογίε που καταθέσαμε όσον αφορά την άμυνα. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις πρωτοβουλίες κάθε είδου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να προστατεύσουμε και τις κρίσιμε υποδομές μας. Το κέντρο αυτό εμπειρογνωμοσύνης πρέπει να υπερασπιστεί την Ευρώπη, αλλά όχι να κατασκευάζει όπλα για τον κυβερνοχώρο. Θυμίζω ότι δεν είναι μόνο οι εφαρμογές κρυπτογράφησης. Πρέπει να ενισχύσουμε το εφιστάμενο πλαίσιο για τις λεγόμενες διτές τεχνολογίες για πολιτικές και στρατιωτικές χρήσεις. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και τους κοιοδησηγητές για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ. And thank you. Εγώ σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Ντάντι έχει το λόγο από την Επιτροπή εσωτερικής αγορά και προστασίας καταναλωτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε, σε έναν όλο και πιο ψηφιασμένο και συνδεδεμένο κόσμο, η κυβερνοασφάλεια είναι πραγματική πολιτική προτεραιότητα με την έγκριση τη πράξη για την κυβερνοασφάλεια. Αποκτά αρμαρμονισμένα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τι επιθέσει στο διαδίκτυο. Η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και συντονισμού τη ενίσχυση και δημιουργία ενό ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού ε, σχήματος επιστοποίησης αποτελούν την προσθέμενη αξία του κανονισμού. Πρέπει όμως να κάνουμε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο βήμα ένα μηχανισμό υποχρεωτικό για την πιστοποίηση για τα προϊόντα της οποίας ε, η χρήση ε, προορίζεται για ε, κρίσιμους φορείς. Παραδείγματο χάρη, ε, κάποιοι με στο μέλλον με ένα κινητό ή με ένα τόμπλετ θα πρέπει να μπορούν να ελέγξουν αν φέρει την πιστοποίηση αυτή. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον προς για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη ε, στην ευρωπαϊκή αγορά των συναφών αγαθών και υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Κύριος Άνσιπ για την Κομισιόν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και την κυρία, τις εισηγήτριες, την κυρία Νίμπλερ και την κυρία Ρέντα όλους τους και ε, και τις ε, επιτροπές που ασχολήθηκαν με αυτούς τους πολύ σημαντικούς νομοθετικούς ε, φακέλους. Θα ενισχύσουν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απεκτικότητά μας να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ως τμήμα της οικοδόμησης ψηφιακών νέων αγορών. Σε ό,τι αφορά τώρα την πράξη, για την ασφαλεία στον κυβερνοχώρο. Υποστηρίζει η Κομισιόν την πολιτική συμφωνία που πέτυχαν οι συνομοθέτε. Αυτή η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα καλής συνεργασίας ε, μεταξύ των ε, συνομοθετών για το μέλλον της ΕΝΗΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και για τη σύσταση της επιστοποίησης ε, της κυβερνοασφάλειας για τις ψηφιακές αγορές. Θα ενδυναμώσει τον κανονισμό σε πολύ σημαντικούς τομείς. Συγκεκριμένα θεσπίζει ένα εύρωστο και ξεκάθαρο πλαίσιο για την ε, πιστοποίηση στην κυβερνοασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ε, συμφωνήσει επί προγραμμάτων πιστοποίησης που θα ε, διατηρούν την ασφάλεια των πολιτών, θα φροντίζουν για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και θα καλύπτουν τις ανάγκες των ομιλητών και των αγορών. Θα δώσει στην ΕΝΗΣΑ μια ισχυρότερη εντολή για να συνεισφέρει στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΕΝΗΣΑ e χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη της ε, προκειμένου να βοηθήσει να διασφαλιστούν ε, οι μελλοντικέ ευρωεκλογέ. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό είναι το εξή. Θέλω να καλωσορίσω την έκθεση για το κέντρο ικανοτήτων ε, και ε, για το Δίκτυο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού. Αυτή η πρόταση αποτελεί στοιχείο κλειδί για να οικοδομήσουμε μία ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να οικοδομήσουμε τις ικανότητές μας ε, στον κυβερνοχώρο συμπεριλαμβάνει όλη την έρευνα που υλοποιήθηκε δυνάμει του ορίζοντα 2020 ναι. αλλά και στο μελλοντικό πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Είναι προ το στρατηγικό συμφέρον τη Ευρώπη να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε θα είναι στην πρώτη γραμμή στο να αναπτύξουν νέε ψηφιακέ τεχνολογίε έχουμε προτείνει το πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης για να χρηματοδοτήσει την ε, ανάπτυξη νέων ε, ικανοτήτων στην Ευρώπη και για να υπάρξουν ε, επενδύσεις και από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για την ανάπτυξή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα ομαδοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο να αναπτύξουν τις νέες ικανότητες για την ψηφιακή νέα αγορά. Ο, και, και δημόσιο τομέα θα συμμετέχουν, αλλά και ο ακαδημαϊκό τομέα. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο συμφωνεί με το όραμά μας ε, για ε, το μέλλον ε, για το σημασία του να διασφαλίσουμε πρόσβαση ε, στα οικονομικά μέσα βάσει προτεραιοτήτων που θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Το Κοινοβούλιο έχει εργαστεί σκληρά επί του φακέλου αυτού σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το ευχαριστώ ενδυναμώνοντας ε, τις ικανότητες ασφάλειας του κυβερνοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την αλυσίδα αξίας, διασφαλίζουμε ότι η ψηφιακή ε, μια αγορά που έχουμε οικοδομήσει θα είναι ισχυρότερη και θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις κυβερνοαπειλές. Εν υπομονώ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ένα λεπτό κύριος Χάουαρθ. Επιτροπή Προϋπολογισμού. Madam President, cyber attacks are not... Κυρία Πρόεδρε, οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι κάτι της μόδας το οποίο σύντομα θα εξαφανιστεί πάλι και είναι κάτι που έχει να κάνει με πολλά χρήματα και τη σοβαρή πολιτική. Η μόνιμη εντολή του οργανισμού που θα αντισταθεί σε αυτές δεν είναι πολυτέλεια, είναι κάτι απολύτως απαραίτητο. Επίσης, ε, είναι γεγονός ότι η κακοί άνθρωποι της πληροφορικής πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν από καλούς. Θα πρέπει λοιπόν να επανδρωθεί ο οργανισμός με τους καλύτερους ανθρώπους στο πεδίο αυτό. Θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά ο οργανισμός και συζητιέται το αν η διπλή έδρα είναι ε, ε, σκόπιμη. Πάντως ε, επικροτούμε την έκθεση διότι ε, το κυβερνοέγκλημα ποτέ δεν κοίταζε τα σύνορα και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διασυνοριακά. Σας ευχαριστώ. Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, η κυρία Γκραπίνη, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα συζητάμε μια έκθεση η οποία πρέπει να υιοθετηθεί γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. 80% του πληθυσμού της Ένωσης είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Και η οικονομία βεβαίως εξαρτάται από το διαδίκτυο, από την ψηφιακή τεχνολογία. Βεβαίως αυτό σημαίνει και κινδύνους όπως οι κυβερνοεπιθέσεις. Θεωρώ λοιπόν πως ε, η συζήτηση και η έκθεση για την ίδρυση αυτού του κέντρου είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και τα εθνικά κέντρα συντονισμού. Τα ανέφερε και ο Επίτροπος γι' αυτό. Έχει μεγάλη σημασία να λειτουργούν αυτά σωστά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έγιναν δεκτές οι τροπολογίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο ευπαθείς από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχουν ειδικού για την κυβερνοασφάλεια Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κέντρα για να μπορέσουν να υποστηριχθούν ε, σωστά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Σας ευχαριστώ για την Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Για να λεπτό, ο κύριος Φραντς. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εξ ονόματος της Επιτροπής μας συγχαίρω τον συνάδελφο Νίμπλερ για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νέα εντολή της ΕΝΙΖΑ. Βεβαίω όλα αυτά είναι πολύ ωραία και σημαντικά, αλλά δυστυχώς εθελοντικά το άρθρο 48α που ήθελε να εισαγάγει η Επιτροπή μας θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί θα προέβλεπε ένα υποχρεωτικό ε, στάνταρ για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Εδώ λοιπόν στο Κοινοβούλιο μιλάμε πάντα για περισσότερη ασφάλεια και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι ε, για ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζουν οι πολίτες γιατί οι συσκευές τους μπορεί πολύ απλά να χακαριστούν και έτσι να υπάρξει επίθεση σε άλλες ε, Κρίσιμε υποδομέ. Για να κάνω μια παρομοίωση, μιλάμε για μια έγκριση τύπου σε αυτοκίνητα τα οποία δεν θα είχαν τα κατάλληλα συστήματα ταχυτήτων ή φρένων. Αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και δεν ε, συζητάμε άδικα αυτή την εβδομάδα για την ασφάλεια των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΝΙΖΑ ή και πιο πριν ε, στην ε, οδηγία περί ασφάλειας των προϊόντων να συζητήσουμε το θέμα. Η κυβερνοασφάλεια είναι βασικό ζήτημα πλέον της ασφάλειας της κοινωνίας. Πρέπει να το πάρουμε τόσο σοβαρά όσο απαιτείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πάμε στις πολιτικές ομάδες. Κύριε Ρούμπιχ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Αγγέλικα Νίμπλερ για τη συζήτηση αυτή. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στα συστήματα. Θέλουμε ε, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές μας ε, με εμπιστοσύνη. Δεν θέλουμε όμως προτεξιονισμό. Θέλουμε ασφάλεια για τους πολίτες κατά την χρήση των του εξοπλισμού τους και δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα από τον πολιτικό ή τον αμυντικό τομέα. Ε, και πράγματι όχι μόνο η Κίνα είναι το πρόβλημα. Πρέπει γενικά να ασχοληθούμε με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικός τομέας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Ρέντα. 28 κράτη-μέλη μπορούν με συντονισμό να πετύχουν πολύ περισσότερα από ό,τι κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Και ευχαριστώ και για την τροπολογία για τον τριμερή διάλογο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν τις εκλογές ε, να παρουσιάσουμε αποτελέσματα στους πολίτες μας. Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων και η ε, οδηγία για την ε, για την κυβερνοασφάλεια πρέπει να εφαρμοστούν και να δημιουργηθούν κέντρα αριστείας στα πανεπιστήμια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές διαδίκτυο. Η ε, διευκόλυνση ε, ε, συνδέοντας την Ευρώπη καθώς και τα σχετικά ταμεία θα έχουν μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά ο κύριος Κουρουμπάσεφ. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε για το θέμα αυτό, ιδίως την κυρία Νίμπλε, τον κύριο Τέλισκα. Έχουμε διπλασιάσει τον προϋπολογισμό της ΕΝΙΖΑ, έχουμε μόνιμη εντολή και τις δικές μας τεχνικές ικανότητες της ΕΝΙΖΑ που ελπίζω ότι αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση και ότι θα αυξηθούν οι ικανότητες αυτές ε, επιτρέποντας η Ελληνίσα να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη. Όπως και άλλοι εδώ, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ικανοποίησή μου με την ρύθμιση για την εθελούσια πιστοποίηση. Την, η ιδέα της υποχρεωτικής πιστοποίησης θα οδηγούσε σε ένα ανταγωνιστικό πλονέκτημα για κάποιους και όχι μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών εν τέλει. Υπάρχει η αντίφαση αυτή στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού ένα, ε, τα εθνικά κέντρα ικανοτήτων, ένα απαιτεί η πιστοποίηση να αφορά κατοίκους της Ένωσης. Αν περάσει κάτι τέτοιο δεν θα επιτρέψει στις θηγατρικές ε, επιχειρήσεις από τρίτες χώρες να μετάσχουν στις διαδικασίες αυτές, μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στην κύβερνο ασφάλεια. Επιπλέον δώσαμε εξουσίες για έρευνα και ανάπτυξη στην, ε, και στον κανονισμό για τα κέντρα ικανοτήτων έχουν δοθεί αντίστοιχες αρμοδίτες. Αυτό μπορεί να υπάρξει να οδηγεί σε μια επικάλυψη και υπάρχει βέβαια πάντα και ο κίνδυνος υπερβολικής νομοθετικής ε, ρύθμισης χωρίς ουσιαστική ε, υλοποίηση. Τρία εργαλεία πάντως έχουμε τα ΚΕΤ, το, το, την πράξη για την ε, κυβερνοασφάλεια, τα κέντρα ικανότητας και τα το, δίκτυο, το οργανισμό για τα δίκτυα εθνικών και συντονισμού. Η ΕΝΗΣΑ θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα αμέσως για να δημιουργήσει μια διαδικασία πιστοποίησης, κάτι που είναι αναγκαίο ακόμα και σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κρασνοντεύσκη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι το θέμα της πιστοποίησης είναι ζωτική σημασία, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, μόνο σε θελούσια βάση προ το παρόν. Η Επιτροπή ωστόσο μπορεί να επαναξετάσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής σε ένα στο εγγύς μέλλον. Όπως ξέρετε η σημασία της κυβερνοασφάλειας είναι τεράστια. Ανά τον κόσμο έχουμε πέντε δις μηχανήματα που ανά πάσα στιγμή βρίσκονται στο ίντερνετ. Κάποιοι υπολογίζουν ότι τα μηχανήματα αυτά το 2021 θα είναι 21, θα είναι 15 δις. Ωστόσο, τα μηχανήματα αυτά δεν έχουν πάντα την σωστή ασφάλεια. Ξέρουμε ότι οι επιθέσεις hacker μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σε ένα νοικοκυριό ή σε έναν ιδιοκτήτη. Μια τέτοια επίθεση σε πολλά εργαλεία και μηχανήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κυβερνο, ε, από κυβερνοεπιτιθέμενους για να καταστρέψουν μία ολόκληρη χώρα μπορούν να κλείσουν όλες τις ηλεκτρικές γεννήτριες σε μία περιοχή. Η ασφάλεια λοιπόν των οικοκυριών συνδέεται στενά με την στρατηγική ασφάλεια. Αρκεί, για παράδειγμα, λένε οι ερευνητές, να επηρεάσεις 90 μηχανήματα κλιματισμού που συνδέονται με την πηγή ηλεκτρισμού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την σωστή ασφάλεια για κρίσιμες, για κρίσιμες υποδομές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέλιτσκα, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Νίμπλερ οπωσδήποτε και τους Κουρούμπασεφ και Ντάντε για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στο θέμα μας τώρα. Δεν είναι μυστικό νομίζω ότι οι κυβερνοεπιθέσεις και η κυβερνοασφάλεια είναι σημαντικές προτεραιότητες για την κοινή γνώμη και δικαίως, γιατί είμαστε ευάλωτοι. Σήμερα είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε επιθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και άλλα σοβαρά ζητήματα, αλλά ακόμα διαχειρίσιμα. Αλλά αύριο, τέλο πάντων τώρα δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή απειλή που θα αφορά την υγεία, την ασφάλεια, ευρεία τη ενία κτλ. Και αυτά τα οποία καταφέραμε εδώ και με την ενίσα είναι ε, το να μπορούμε να αντιδράσουμε. Βεβαίω, εντάξει, πάντα μπορούμε να συζητάμε το εάν επαρκεί ή όχι, αλλά είναι αυτό το οποίο είναι εφικτό την ημέρα που ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα ήθελα κάποια κράτη-μέλη να αντιληφθούν ότι είμαστε τόσο ισχυροί όσο ο ασθενέστερος κρίκος. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό ακριβώς θα ήθελα εδώ πέρα να επισημάνω την τελευταία δήλωση του Προέδρου Μακρόν και της Προέδρου του Τσεντεού που μίλησε για ε, την απειλή προς την δημοκρατία. Διαφορετικό ζήτημα, αλλά πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Και βεβαίως ε, έχουμε μία βάση στην οποία μπορούμε να βασιστούμε και ε, εγώ θα φροντίσω να δω τι έκανε ο κύριος Μακρόν για αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Σας ευχαριστώ κύριο Συντελούντε για λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι κοινωνίες μας γίνονται όλο και πιο ψηφιακές και γι' αυτό γίνονται όλο και πιο ευάλωτε. Ε, και γι' αυτό είναι ε, ιδιαίτερα ε, θετικό ότι αύριο θα ψηφίσουμε για να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια, για να ενισχύσουμε τα ψηφιακά μας συστήματα. Με πιο αυστηρούς κανόνες πιστοποίησης μπορούμε να χρησιμοποιούμε με ασφαλή τρόπο τα κινητά μα τηλέφωνα, του υπολογιστές και τα άλλα ψηφιακά προϊόντα με την ομοθεσία αυτή θα ε, ενισχύσουμε την ψηφιακή μας ε, ανθεκτικότητα και θα έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις στον τομέα αυτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριο Σκόλιτσεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυβερνοασφάλεια είναι επίκαιρο θέμα τα τελευταία χρόνια. Τον Αύγουστο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μία πρώτη δέσμη μέτρων ε, για το θέμα αυτό ε, με στόχο την ενίσχυση του ΕΝΙΖΑ. Τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού και το δίκτυό τους θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν διότι αυτά θα εκπονήσουν τμήματα ε, του, της ψηφιακής Ευρώπης και του Ορίζον Ευρώπη και θα διευκολύνουν τις εργασίες του συνολικού δικτύου που ασχολείται με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Έχω συμφωνήσει ήδη με ε, τους εισηγητές να ε, στηρίξουμε ε, το ανοιχτό λογισμικό και το δωρεάν λογισμικό. Έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Δεν θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε σε ε, προϊόντα διπλής χρήσης ε, για ε, την άμυνα. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση και είναι σημείο κλειδί της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεσεβαλία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η νέα αυτή πρωτοβουλία επιτρέπει στις εθνικές αρχές να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες. Για να είναι αποτελεσματική ωστόσο η κυβερνοασάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σεβασμό των, κρατών, των κυρίαρχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Η παραβίαση, από την παραβίαση της ιδιωτικής ε, ζωής μέχρι την, τις οικονομικές ατασφαλίες, οι, οι κυβερνοεπιθέσεις πλήττουν την καθημερινότητά μας ε, Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Πέραν της ε, συνεργασίας, η εθελούσια πιστοποίηση επιτρέπει στον καταναλωτή καλύτερη ενημέρωση για την προστασία που, έχει, που έχουν τα προϊόντα που αγοράζει. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μόνο μία υποχρεωτική πιστοποίηση θα επιτρέψει την εξασφάλιση την μεγαλύτερη ασφάλεια του ίντερνετ των πραγμάτων που αυξάνεται ε, εκθετικά. Η κυβερνοασφάλεια μετατρέπεται έτσι σε τεράστιο ζήτημα και είναι λογική αύξηση του σχετικού προπολογισμού. Ωστόσο, μια αύξηση 40% του προπολογισμού τη ΕΝΙΖΑ μέχρι το 2022 δεν πρέπει να μα οδηγεί να ξεχάσουμε ότι πρέπει να μειώσουμε συνολικά το προπολογισμό τη Ένωση λόγω του Brexit. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κέιλ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την συνάδελφο, την κυρία Νίμπλερ, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Νομίζω πως η συμφωνία πέτυχε αυτό το οποίο θέλαμε και θα μας προστατεύσει από κυβερνοεπιθέσεις. μια εύρωστη στρατηγική είναι σημαντική για να αποθήσουμε κυβερνοεπιθέσεις κατά της ενέργειας, της αεροπορίας, του εμπορικού τομέα και των κρατών πλέον ε, στοχεύουν ε, τέτοιες υποδομές οι εγκληματίες για σκοπούς ε, τρομοκρατικούς και εγκληματικούς. Και κάνουμε ένα βήμα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις υποθέσεις, όπως επίσης και το κακόβουλο λογισμικό και τις απάτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε τις κρίσιμες υποδομές, την υποδομή ενέργειας δηλαδή, την βιομηχανία, αλλά και άλλες υποδομές από τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, το να πέσουν τα δίκτυα ενέργειας ε, θα προκαλέσει τεράστιες ζημιές οικονομικές και μη. Επίσης σημαντικό είναι ότι ενισχύει το ρόλο της ΕΝΙΖΑ και η δικιά μου η χώρα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας κόμβος κύβερνο ασφάλειας για την Ευρώπη καθώς έχει ήδη το εκπαιδευμένο δυναμικό και ε, φιλοξενεί ήδη τις μεγαλύτερες εταιρείες όπως την VMware και άλλες οι οποίες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά για να προλάβουν τέτοιες επιθέσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοιες υπηρεσίες και να παίξουμε παγκοσμίω ηγετικό ρόλο. Και ελπίζουμε να αναπτυχθεί ο κλάδος τα επόμενα χρόνια. Τέλος, ήταν τιμή μου το ότι πέρσι πήγα στην Silicon Valley με μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω πως και η βοήθεια αυτών των ανθρώπων θα είναι σημαντική. Σας ευχαριστώ κύριος Γκάιερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είχα την χαρά να είμαι σκιώδης εισηγητής για την πολιτική μου ομάδα για το ε, Κέντρο Ικανοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια. Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την επικροτούμε καθώς ε, και την ε, θέση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία. Η πολιτική μου ομάδα ε, SND, ε, βρίσκει ιδιαίτερα σημαντική την συνεκτικότητα στις δομές που περιλαμβάνουν τον οργανισμό ΕΝΙΖΑ. Θέλαμε να πετύχουμε σωστή διατύπωση για να εξασφαλίσουμε μια καλή συνεργασία. Το θέμα της διακυβέρνησης ε, είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ο οργανισμός να λειτουργεί ε, καλά μαζί με τα εθνικά κέντρα για να έχει πρόσβαση στην απαραίτητη εμπειρογνωσία και ε, για να ευνοηθούν ευρωπαϊκοί φορείς από το πρόγραμμα αυτό. Επίσης, προγράμματα στρατιωτικά θα πρέπει ε, να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Πολιτικά προγράμματα θέλουμε να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα μη στρατιωτικής χρήσης και γι' αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε απολύτως με την διατύπωση ε, στην θέση της Ήτρα. Όσον αφορά το να πάμε κατευθείαν σε τριμερή διάλογο, έχω την εντύπωση ότι όσον αφορά ε, τη χρηματοδότηση την στάθμιση των ψήφων κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με τη θέση του ε, Συμβουλίου. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι την Τετάρτη καλό είναι να λάβουμε σχετική απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάκετ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης αυξάνεται και η σημασία της κυβερνοασφάλειας. Και βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις μας δεν είναι επαρκώς θωρακισμένες για αυτές τις απειλές. Γι' αυτό τώρα φέραμε το νομοθέτημα αυτό. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική με πολλά και διάφορα μέτρα για να επενδύσουμε στην ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από κυβερνοεπιθέσεις. Και όχι μόνο αυτό. Αφήνουμε χώρο σε κράτη και επιχειρήσεις για να κάνουν τις μεταξύ τους διευθετήσεις και να βασιστούν στην καινοτομία. Βεβαίω, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή. Ελπίζω λοιπόν να τα παρακολουθήσει όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη όπως το Βέλγιο από μόνα τους να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα. Ας γίνει λοιπόν η Ευρώπη ασφαλής στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Μιλινάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σήμερα συζητάμε ένα καθοριστικό βήμα στον καθορισμό μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας για την σύσταση ε, δυνατοτήτων τελευταίας τεχνολογίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πραγματική απάντηση στην ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών των κρατών μελών με τον κλάδο έτσι ώστε οι πολίτες και οι καταναλωτές να έχουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς να βασίζονται σε εισαγόμενες λύσεις από τρίτες χώρες. Χάρη στις ε, έντονες διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή και την ε, συνεργασία που είχαμε με την Γιούλια Ρέντερ και τους άλλους και έχουμε τώρα ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό Αυτοκέντρο Αριστείας θα συντονίζει τις προτεραιότητες και δεν θα γίνονται διπλές προσπάθειες στα κράτη-μέλη. Και πάντα σε σχέση με τη νέα εντολή της ΕΝΙΖΑ. Δεύτερον, το κέντρο αυτό θα παρέχει χρηματοδότηση από τα προγράμματα Ορίζοντας και Ψηφιακή Ευρώπη σε καινοτόμους πρωτοβουλίες. Και τρίτον, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενε προσεγγίσει των κρατών μελών μέσω της συνέργεια στρατιωτικών και πολιτικών εφαρμογών για να χρησιμοποιηθούν πλήρως και αποδοτικά υφιστάμενοι πόροι. Τέλος, ως ε, εισηγητή του σχετικού προγράμματος ε, χαίρομαι ιδιαίτερω για την δομή διοίκηση του κέντρου. και την σχέση με τα κέντρα ψηφιακής καινοτομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ματίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, η ζωή μας γίνεται online. Γι' αυτό τα προσωπικά μας δεδομένα αποτελούν ένα αγαθό που αποκτά και αποκομίζει όλο ένα και μεγαλύτερη αξία και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί εγκληματίες που θέλουν να κλέψουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε σαφείς ενδείξεις και αποδείξεις γι' αυτό, το Facebook μεταξύ άλλων. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις δράσεις μας με κέντρο την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι άνθρωποι στο, στη μάχη αυτή. Χρειαζόμαστε να δώσουμε δυνατότητες στις πολίτες να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις για την προστασία των δεδομένων τους. Όχι μόνο η ΕΝΙΖΑ, αλλά όλες οι αρχές πρέπει να συμβάλλουν στη μάχη αυτή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάμπ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την εξαιρετική της δουλειά την συνάδελφο Αγγέλικα Νίμπλερ. Ε, ελπίζω η Επιτροπή μας, η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά να μπόρεσε να συμβάλλει σημαντικά στην έκθεση αυτή. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σε 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται, υπολογίζεται η ζημιά παγκοσμίω ε, για ε, από τη, θέματα από κυβερνοεπιθέσεις ε, και αυτό δείχνει την σημασία του ΕΝΙΖΑ. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αμέσως να καθορίσει στόχους και να προστατέψει έτσι μια σημαντική πτυχή της εθνικής ασφάλειας. Για το... Μέχρι το 2020 απολογίζεται να επενδύσουμε 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, πρόκειται να επενδύσουν 22 δισεκατομμύρια. Ε, μένουμε πίσω λοιπόν στο θέμα αυτό. Και θα πρέπει όχι μόνο να δώσουμε νέες αρμοδιότητες ε, στον Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην κυβερνοασφάλεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Σωρίνιο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ασφάλεια σήμερα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, είναι κομβική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την προστασία των πολιτών της από τις απειλές των νέων τεχνολογιών. Ε, πρέπει λοιπόν και ταυτόχρονα μπορούν να φτάσουν σε πραγματικές ε, αποφάσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις ικανότητες της ΕΝΙΖΑ δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό χώρο κατά, τις, ε, των κυβερνοεπιθέσεων με γρήγορη ανταπόκριση ταυτόχρονα υιοθετώντα ένα σύστημα πιστοποίησης προϊόντων και διεργασιών. Τα εθνικά κέντρα γνώση, ικανοτήτων θα έχουν ε, μεγάλο ρόλο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδίως στην ψηφιακή Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας τις δυνατότητες με ένα σύστημα που επιτρέπει να ε, αντικατοπτρίζονται σωστά οι ε, διάφορες ανάγκες που υπάρχουν σε εθνικό πλαίσιο. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλερ, αλλά λείπει. Θα δώσω λοιπόν το λόγο για ένα λεπτό στην κυρία Καϊλή. Yes. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διαπραγμάτευση και την ευτυχή κατάληξη του τριλόγου αυτό είναι το επόμενο σημαντικό βήμα μετά την οδηγία ε, nis για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην ευρωπαϊκή ένωση που προστατεύει και την οικονομία και την κοινωνία μας αλλά και τη δημοκρατία μας. καθημερινά έχουμε κυβερνοεπιθέσεις ε, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τρίτες χώρες και η ψηφιακή μας οικονομία εξελίσσεται εκθετικά και αυτές οι επιθέσεις θα εξελίσσονται επίσης εκθετικά. είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ένωση στην αντιμετώπιση με εργαλεία και πολιτικές ε, όχι όμως μόνο στη συνεργασία αλλά και στο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και στην ανταλλαγή πληροφοριών γιατί είναι ένας κινούμενος στόχος η κυβερνοασφάλεια ο ΕΝΙΣΑ λοιπόν που εδρεύει στην ελλάδα είναι σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας αυτής. με την ψήφιση του eu Security act ενισχύεται πολύ αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες και στελεχώνεται με ειδικού για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών. ωστόσο οφείλουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά τις επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια στηρίζοντας την καινοτομία και μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της ευρωπαϊκής ένωσης επενδύουμε γύρω στα δύο δισεκατομμύρια για το 2021-2027 θεωρώ ότι είναι στο σωστό δρόμο και ελπίζω ο νέος κανονισμός για τα competence Center και networks που επίσης ψηφίζουμε να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει και ο τρίλογος ώστε με αυτή τη σύνθεση του ευρωκοινοβουλίου να μπορέσουμε ουσιαστικά να ολοκληρώσουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο για την κυβερνοασφάλεια. Ε, θεωρώ λοιπόν πως πετυχαίνουμε πολλά σήμερα ε, έχουμε λίγο ε, δρόμο ακόμα μπροστά μας έχοντας ολοκληρώσει και το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνουμε ότι οι απειλές είναι διαρκώς και αυξανόμενες. σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καϊλή. Καλησπέρα σε όλους σας. Μπαίνουμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Στο Γεύσκι ήταν ο πρώτος, λείπει ωστόσο. Μπόγκοβιτσε μετά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. ο κόσμος είναι όλο και πιο διασυνδεδεμένον, όλο πιο ψηφιοποιημένος και έτσι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί σημαντική πρόκληση. Τα συστήματά μας ε, στον τομέα της ενέργειας, ε, στον τραπεζικό τομέα, ε, οι εκλογές, ακόμα και η ασφάλεια του ατόμου διακυβεύονται. Ήμουνα θύμα κλοπής ταυτότητας και γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο ή και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στηρίζω αυτή τη δέσμη μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει ενωμένη το θέμα αυτό, διότι κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του να προστατευτεί από τις κυβερνοεπιθέσεις. Επισκέφθηκα το Ισραήλ και είδα εκεί τι μπορεί να καταφέρει ένα κράτος με 10 εκατομμύρια πολίτες. Στηρίζω τη δέσμη μέτρων αυτών, διότι το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την κυβερνοασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καπούτο. E ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα δίκτυα και τα, τα δίκτυα πληροφορική είναι πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης, εξού και η σημασία μείωση στο δυνατό των κινδύνων που ενέχουν ε, παρέχοντας τους καταναλωτές την εμπιστοσύνη που χρειάζεται. Ο κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια θα δώσει στην Ευρώπη μια, ένα όραμα μακροπρόθεσμα ενισχύοντα ε, τις δομές της ΕΝΙΖΑ και εισάγοντα ένα σύστημα πιστοποίησης ε, κυβερνοασφάλειας, μειώνοντας έτσι την δαπανηρή, το δαπανηρό κατακαιρματισμό υπηρεσιών και διαργασιών. Μέσω Συμφωνώ με την εθελούσια προσέγγιση της πιστοποίησης με βασικές εγγύσεις ωστόσο για τα προϊόντα ή διαργασίες που υπάγονται σε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας καλύτερο θα ήταν ένα υποχρεωτικό σύστημα. Οι παραγωγοί και κατασκευαστές προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για την πιστοποίησή της ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει επαρκή στοιχεία τη στιγμή που επιλέγει το μηχάνημα που θα αγοράσει, τη συσκευή που θα αγοράσει. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Μιλούμε για την κυβερνοασφάλεια, τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Τι μέτρα όμως κύριε Επίτροπε κύριε ansip θα λάβει η ευρωπαϊκή ένωση ενάντια σε ένα κράτος μέλος το οποίο παρακολουθεί τους πολίτες του διότι προ λίγων ημερών στις 4 μαρτίου είχαμε προληπτικές συλλήψεις στην πόλη των γιάννητσών οπαδών ελλήνων πολιτών οι οποίοι διαφωνούν με την κατάπτυστη συμφωνία των πρεσπών και τους συνέλαβε προληπτικά η αστυνομία και η υπουργό προστασία του πολίτη η κυρία γεροβασίλη είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τα social media παρακολουθεί το facebook μαζεύει πληροφορίες για τους πολίτες και κάνει προληπτικές συλλήψει και στέλνει τον κόσμο στα δικαστήρια Όσου αγωνιστές παλεύουν ενάντια στο ξεπούλημα της μακεδονίας μα και τη ιστορία μα. αυτά είναι καταγεγραμμένα. τι μέτρα θα πάρετε λοιπόν; είναι δυνατόν να έχουμε παραβίαση τη νομοθεσία παραβίαση του κανονισμού gdpr και να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και παρακολουθεί το διαδίκτυο και κάνει προληπτικές συλλήψεις παράνομες. θέλω την άποψή σας κύριε επίτροπε να καταγγελθεί αυτή η πρακτική στέρησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ελλήνων πολιτών. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σδροϊεύσκη, επέστρεψε και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω τι είχαμε πει εδώ πριν από πέντε χρόνια, όταν ξεκινούσε η θητεία μας. Τότε ε, ο κόσμος αγνοούσε την κυβερνοασφάλεια. Υπήρχαν πολλές απειλές που αγνοούσαμε παντελώς. Αυτό άλλαξε. Βρισκόμαστε στην περίεργη κατάσταση να θεωρούμε ότι αυτό είναι καλό, διότι ενισχύουμε το θεσμικό μας πλέγμα και δημοσιονομικά αυξάνουμε το προσωπικό και διευρύνουμε τις δυνατότητες που έχουν οι υπηρεσίες. Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, χάσαμε χρόνο και αυτό είναι κρίμα. Ο κόσμος προχώρησε, έγιναν πράγματα, εξελίχθηκαν διαδικασίες. Ε, αυξήθηκαν οι απειλέ. Πρέπει να υποστηρίξουμε ωστόσο την έκθεση γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλειά μα. και ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια γι' αυτό. Τελειώσαμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Δίνω το λόγο τώρα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Άνσιπ, να κλείσει την παρέμβασή του. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωβουλευτές για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις απόψεις που εκφράσατε σήμερα. Η πράξη για την κυβερνοασφάλεια θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο πιστοποίησης και θα δώσει μόνιμη εντολή στον ΕΝΙΖΑ. Έτσι, η ψηφιακή ενιαία αγορά θα γίνει πιο ισχυρή και πιο ασφαλής. Όσο ε, αυξάνεται και μεγαλώνει η ψηφιακή εσωτερική αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά και τους κινδύνους ε, και τα ωφέλη. Έχουμε λοιπόν συλλογική ευθύνη να διασφαλίσουμε την σωστή αντιμετώπιση των κινδύνων και την ε, διασφάλιση των προϊόντων και υπηρεσιών του, του ψηφιακού κόσμου και η πράξη για την κυβερνοασφάλεια ε, συνδυάζεται με άλλα νομοθετήματα και τα ε, κέντρα ε, ικανοτήτων θα διασφαλίσουν την ύπαρξη ευρωπαϊκού δυναμικού και ευρωπαϊκών πόρων για μια ψηφιακή εσωτερική αγορά. Λογικά θα πρέπει τώρα να έχουμε αρκετούς πόρους για να διασφαλίσουμε την κυβερνοασφάλεια. Και τώρα την εμπειρογνωσία αυτή και την πείρα θα πρέπει να την μετατρέψουμε σε καινοτόμα προϊόντα και να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να φροντίσουμε το ψηφιακό οικοσύστημα να παρέχει τα μέσα ώστε να ανταγωνιζόμαστε στι ε, διεθνεί αγορές τεχνολογίας. Αυτό απαιτεί συντονισμένες εργασίες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και ε, απαιτεί και συνδυασμό προσπάθειων ε, και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι πολύ ευγνώμων για τον γρήγορο ρυθμό της νομοθετικής δουλειάς και με την ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα όπως ε, έχετε δηλώσει ότι είναι η πρόθεσή σας, ε, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός της παρούσας εντολής και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει πόσο ε, μεγάλη είναι η πολιτική σημασία του θέματος αυτού για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα κυβερνοασφάλειας που βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Προσβλέπω στις προσεχείς διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχω, έχει τώρα η κυρία Νίμπλε, η συγγήτρια. Liebe Kollegen, verehrter Herr Vizepräsident, nur ein herzliches Dankeschön von meiner Seite für die ähm, für mich sehr inspirierende. Heute mich freut es, dass wir τους συναδέλφους για την συζήτηση αυτή. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι για την τεράστια σημασία της κυβερνοασφάλειας. Και βεβαίως σας ευχαριστώ και για τις ε, πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις σας στην έκθεση. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη στο θέμα αυτό και θεωρώ ότι τα καταφέραμε. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερος σήμερα για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματο. Για εμένα είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ακόμη μια φορά ότι έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να θέσουμε διεθνείς προδιαγραφές. Λοιπόν, είναι σημαντικό το ότι έχουμε αυτήν την δυνατότητα. Και αν καταφέρουμε για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές, για όλο αυτό το οικοσύστημα να δημιουργήσουμε εμείς τις προδιαγραφές, θα έχουμε καταφέρει πραγματικά κάτι. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν. Νομίζω δεν ήταν επιφανειακή η συζήτηση. Ε, καταλήξαμε σε κάποιες καλές λύσεις και κάποιοι ε, συνάδελφοι ήθελαν να είναι πιο φιλόδοξοι ε, ειδικά όσον αφορά την υποχρεωτική πιστοποίηση κρίσιμων υποδομών αλλά ας κάνουμε το πρώτο βήμα και βλέπουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όσους συνεργάστηκαν και θα δούμε ποια θα είναι και εφαρμογή στα κράτη-μέλη για να έχουν οι πολίτες περισσότερη ασφάλεια στα προϊόντα τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα η κυρία Ρέντα, η άλλη Σας ευχαριστώ. Όπως βλέπετε από τη συζήτηση υπάρχει μια ευρεία συνένεση για την ουσία του κέντρου αυτού, αλλά υπάρχουν ε, και διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω την προσέγγιση μου. Πρώτα απ' όλα, ήδη στην Επιτροπή μας ε, καταφέραμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, ε, να κατευθυνθούν οι πολιτικές δαπάνες σε στρατιωτικές εφαρμογές. Αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν, χρηματοδοτούμε και δραστηριότητες που θα υπονομεύουν την κυβερνοασφάλεια όπως τις πίσω πόρτες στα συστήματα και άλλα τέτοια παρόμοια. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχει μια συνένεση η οποία θα φανεί στην ψηφοφορία της Τετάρτης και αν γίνει αυτό ε, και εγώ θα βοηθήσω να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου ε, με μια πολιτική συμφωνία εντός της θητείας αυτής. Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές διαφορές οι οποίες παραμένουν και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τελικά η θέση του Συμβουλίου. Και βεβαίως δεν θέλουμε συμφωνία με κάθε κόστος. Και ακριβώς λόγω της ευρύτατης στήριξης του Κοινοβουλίου και των αλλαγών που επέφερε το Κοινοβούλιο ε, θα απαιτήσουμε και μεγαλύτερη ευελιξία από Συμβούλιο και Κομισιόν. Οπότε, αν υπάρξει αυτή η συνενετική προσέγγιση, νομίζω ότι έχουμε ελπίδες για κάποια συμφωνία εντός αυτής της ε, θητείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου για τη συμμετοχή μου στην συζήτηση αυτή. Γιατί είμαι και επικεφαλής ε, της ομάδας εργασίας για την ε, κυβερνοασφάλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να, ευχαριστώ το, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Άνσιπ και τον Επίτροπο Κίνγκ επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο ε, για την έκθεση Νίμπλερ και την Τετάρτη για την έκθεση της κυρίας Ρέντα. Περιμένουμε τώρα τον Επίτροπο Χόγκαν. θα έρθει τώρα να πάσα στιγμή. Underway. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Καθίστε. Βλέπετε το Κοινοβούλιο λειτουργεί πάντα αποτελεσματικά και είναι στην ώρα του. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε μαζί. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση δεκαστού για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο κύριος Δεκάστρο, εισηγητής, που έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέκα χρόνια συζητήσεων χρειάστηκε 20 κράτη έπρεπε να νομοθετήσουν για το θέμα αυτό. Χρειάστηκε να επιμείνει το Κοινοβούλιο και με δύο ψηφίσματα, ε, το τελευταίο από τα οποία ε, βοηθήθηκε πάρα πολύ από την κυρία Μαγκίνες και που εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία τον Ιούνιο του 2016. Χρειάστηκαν όλα αυτά για να φτάσουμε σήμερα στην τελική ψηφοφορία της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στον τομέα της ε, ε, αλυσίδα διατροφή. Εξαιρετικό αποτέλεσμα που κατέστη δυνατό χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου μα. που υλοποιήθηκαν με τις σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση. Να αναφέρω κάποιες μόνο. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής που καλύπτει πλέον 100% των γεωργών και πάνω από 95% των, επιχειρήσεων στην Ένωση, περνώντας από 50 σε 350 ε, ε, εκατομμύρια, ευρώ ε, τζίρο. Μείωση, καθορισμό της των, υπο, υποκειμένων στην οδηγία και επιχειρήσεων εκτός Ένωσης. Προστασία στρατηγικών των, των νέων, ζωοτροφές εκτός των άλλων η ενίσχυση και ο διπλασιασμό των απαγορευμένων πρακτικών που πέρασαν από 8 σε 16 με τη συμπερίληψη για παράδειγμα καθυστερήσεων πληρωμών για μη αλλοιώσιμα προϊόντα, άρνηση παροχής ε, γραπτών συμβάσεων, απειλή εμπορικών ε, κυρώσεων σε περίπτωση καταγγελίας, προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του καταγγέλλοντος, για να ξεπεραστεί ο παράγοντα φόβο που συχνά υποχρεώνει του παραγωγού μα να δεχθούν τέτοιε πρακτικέ με το δικαίωμα καταγγελία να, να επεκτείνεται σε όλε τι επιχειρήσει, Υποχρέωση δράση για να τεθεί τέλος σε αθέμητες ε, πρακτικές από εθνικές αρχές, στις οποίες δώσαμε περισσότερες εξουσίες, τόσο ερευνητικά όσο και κυρωτικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, που θα πρέπει να συναντιούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και να ανταλλάσσουν πληροφορίε και βέλτιε πρακτικές για να εξασφαλίσουν μια ομοιογενή και φιλόδοξη εφαρμογή τη οδηγία. Αξίζει να θυμίσουμε ότι μιλάμε για εναρμόνιση στο ελάχιστο όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να βελτιώσουν μέσω των εθνικών τους ε, ρυθμίσεων, μπορούν να διευρύνουν και τον κατάλογο των πρακτικών και τις οργανώσεις που καλύπτονται. Για να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό, συνάδελφοι, χρειάζονται κανένα 11 μήνες από την πρόταση της Επιτροπής, παρά τις προσπάθειες να εμποδιστεί η οδηγία αυτή ακόμα και τώρα. Χρειάστηκε μια ισχυρή πολιτική βούληση από πλευρά όλων. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι κατέστησαν το αποτέλεσμα αυτό δυνατό, ξεκινώντας από τους συναδέλφους της Επιτροπής βέβαια. Τον Επίτροπο κύριο Χόγκαν που ευχαριστώ τους σκιώδεις ηγητές, όλη η ομάδα των, της διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου, τις υπηρεσίες, την Αυστριακή Προεδρία, την Υπουργό κ. Κόστιγκερ, ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε την πολύ καλή δουλειά που έκαναν όλε τι τεχνικέ ομάδε και η δική μου ομάδα βεβαίω. Πρόεδρε, συνάδελφοι, η οδηγία αυτή δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί και θέλει να είναι δίπλα στου πιο αδύναμους, τους γεωργούς, όλους τους πολίτες. Η αλυσίδα αυτή χαρακτηρίζεται από αθέμητες πολιτικές και πρακτικές και κακή χρήση των πόρων. Η βάρος των γεωργών, με μείωση της ε, τιμής που κερδίζουν οι γεωργοί, αλλά και της ποιότητας, διώνοντας, οδηγώντας σε σε εκμετάλλευση της εργασίας των γεωργών. Εμείς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις θευλώσεις αυτές και η οδηγία θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για να φτάσουμε σε μια πιο δίκαιη, ανοιχτή και αποτελεσματική αγορά που μπορεί να δώσει κέρδη σε όλη την κοινωνία, ιδίω δε στον καταναλωτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. Για την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά, ο κύριο Ταραμπέλα έχει το λόγο. Πρόεδρε, η, η έκθεση αυτή είναι μία από τις μεγάλες ε, πρόοδους της θητείας μας. Είναι υποχρέωσή μας να καταπολεμήσουμε τις ανισορροπίες που αντιμετωπίζει ο μικρός γεωργός μπροστά στη συγκέντρωση των μεγάλων επιχειρήσεων διανομής τροφίμων. Αυτό οδηγεί σε προβλήματα στον σημερινό κόσμο. Η διατροφή ωστόσο έπαιρνε μεγάλη προτεραιότητα. Η οδηγία καταργεί τις αφέμητες πρακτικές στην αλυσίδα διατροφής, ενισχύει τη διαφάνεια, κατά την εκβο... την... τους εκβιασμούς των πολυεθνικών. Η εξαιρετική δουλειά του συναδέλφου και φίλου κ. Ντεκάστρο βοήθησε σε μεγάλο βαθμό συνεργαστήκαμε πολύ στενά για να μπορέσει το κείμενο, το τόσο σημαντικό αυτό κείμενο να κλείσει πριν, κλείσει θητή, πριν τελειώσει η θητεία μας. Θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν παραπέρα στην εθνική του νομοθεσία για να ξεριζώσουν άπαξ διαπαντό αυτέ τι βλαβερέ, αθέμητε πρακτικέ, όχι μόνο για του γεωργού, αλλά και για του καταναλωτέ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Χόγκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε, ε, κύριοι συγητές, ε, κύριοι ευρωβουλευτές. Ε, όπως είπε ο κύριος Δεκάστρο, είναι πολύ ε, σημαντικές οι μικρόμεσες επιχειρήσεις και με την πρόταση αυτή αναγνωρίζουμε ότι ε, έχουν βρεθεί σε μειονεκτική θέση οι μικροί γεωργοί. Ε, η ψηφοφορία αυτή θα προστατεύσει τους ε, γεωργούς που βρίσκονται κατάντι στην αλυσίδια εφοδιασμού. Είναι πολύ σημαντική η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσε να μην βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Η και γι' αυτό χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά ανταποκρίθηκε θετικά ε, με μια νομοθετική πράξη που να απαγορεύει τις αθέμητες πρακτικές. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, καθώς και την Προεδρία του Συμβουλίου. Ιδιαίτερα να συγχαρώ τον κύριο Ντεκάστρο και την κυρία Κέρστινγκερ από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές, τον κύριο Ταραμπέλα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, την κυρία Μακέιβαν από την ΔΕΒΕ και την κυρία Αγιούσο από την ΕΝΒΗ καθώς και την κυρία Μαγκίνε, σε σκιώδη η συγγήτρια, την Ανθέα Μάκενταερ την ε, Μαρία Χάιπερ, ε, Κατάινεν, Μαρκοσούρο, Τζάκι Κορνμπέρ, όλοι σας έχετε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να συζητάμε σήμερα αυτή την ε, νομοθεσία ορόσημο. Ο κύριος ε, Ντεκάστρο μας θύμισε ότι μόνο 8 μήνες ε, έχουν περάσει από την έναρξη των εργασιών. Και αυτό δείχνει ότι με πολιτική βούληση όλα μπορούν να γίνουν. Τώρα εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία και σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά την διαδικασία και είμαι βέβαιος ότι και το Κοινοβούλιο θα το κάνει αυτό. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε τον στόχο, δηλαδή να προστατεύσουμε τους αδύναμους ε, απέναντι στους ισχυρούς. Πρώτη φορά έχουμε τέτοιους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι προστατεύονται όλοι οι γεωργοί ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι περισσότερες επιχειρήσεις ε, στον ε, αγροδιατροφικό τομέα. Έτσι θα έχουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού και προστασία από αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, εφόσον το, επιθυμεί, να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα με βάση τους κανόνες εσωτερικής αγοράς. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες ε, πρακτικές οι οποίες επιβάλλονται μονομερώς ε, από τον ε, ένα συμβαλόμενο. Η συμφωνία που θα επιτευχθεί τον Δεκέμβριο θα ισχύει για όλους στην αγροδιατροφική αλυσίδα με, με τζίρο μεγαλύτερο από 350.000 ευρώ. Έχουμε την ειδική ομάδα για τις ε, γεωργικές αγορές ε, που ε, έχει ζητήσει καλύτερο νομικό πλαίσιο και βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς. Γι' αυτό χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο και στους δύο αυτούς τομείς με τον κανονισμό Omnibus και το γνωρίζει αυτό ο κύριος Δεκάστρο και ο κύριος Σεντές καθώς και το παρατηρητήριο της αγοράς. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θέλει να αυξήσει την ε, διαφάνεια ε, στον λιανικό τομέα. Πολύ σύντομα ελπίζω να μπορέσω να σας ανακοινώσω λεπτομέρειες ε, αυτών των πρωτοβουλειών. Μαζί λοιπόν αυτές οι τρεις πράξεις θα βελτιώσει τις ευκαιρίες των γεωργών και θα τους υπερασπίσει από αθέμητες πρακτικές. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι τους συζητητές ε, και την Αυστριακή Προεδρία για τις εργασίες πάνω στην πρόταση αυτή που θα προστατεύσει τους ε, γεωργούς και όπως είπε ο κύριος Ταραμπέλα, κανένας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ε, από την πρόταση αυτή στον αγροδιατροφικό τομέα εφόσον φέρεται σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, ήδη καλέσατε την κυρία Αγιούσαν να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέσα στην αλυσίδα διατροφής η γεωργή σίγουρα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος που πρέπει να προστατευτεί. Αν θέλουμε μια επαρκή γεωργία με καλά τρόφιμα, ο μόνος τρόπος είναι να προστατεύσουμε τους γεωργούς. Διότι όπως η καθώς η διανομή είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη, η γεωργική παραγωγή είναι εξατομικευμένη και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια. Εγώ λοιπόν θέλω πρώτα να συγχαρώ την Επιτροπή που έκανε την πρόταση, το Συμβούλιο και τον κύριο Ντεκάστρο, καθώς και όλους τους κοιόδη ηγητέ, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν αυτή την έκθεση. Παρά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήταν πολύ πιο αυστηρή στο ξεκίνημα, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια καλή τελικά, τελική συμφωνία και για τους γεωργούς και για τη γεωργία. Στην Ισπανία υπάρχει νομοθεσία για την αλυσίδα διατροφής που λειτουργεί πολύ καλά. Χρειάστηκε, καταφέραμε έτσι να υιοθετήσουμε κάποιους στόχους. Ωστόσο, τα, οι στόχοι που αναφέρετε εσείς παραμένουν σημαντικοί. Γι' αυτό το λόγο ένα λεπτό έχω νομίζω. Θέλω απλά να συγχαρώ το Κοινοβούλιο, τον εαυτό μου και όλους μας, διότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και θα προχωρήσουμε. Πριν από πολλά χρόνια, η κυρία Μακίνη ήταν επικεφαλή μια ομάδα εργασία που τελικά καρποφόρησε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλου. Ευχαριστώ. Για τις πολιτικές ομάδες, η κυρία Μαγκίνες πρώτη, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Γεγονό είναι πως οι εκκλήσεις των γεωργών ε, επιτέλους ε, εισακούστηκαν. Το πήρατε σοβαρά και φέρατε μία πρόταση και σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως και θα δούμε τι θα γίνει στα κράτη-μέλη. Και είναι ευπρόσδεκτο τα σχόλιά σας ε, για το ότι θα προσέξετε την εφαρμογή, γιατί βλέπω ήδη κάποια αμφισβήτηση στα κράτη-μέλη, κάποιο δισταγμό για το πώς θα εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς γραφειοκρατία και αποτελεσματικά, έτσι ώστε όσοι έχουν πραγματικά παράπονα να μπορέσουν να έχουν αποτελέσματα. Αλλά για μένα η σημερινή ημέρα είναι πολύ πιο σημαντική από το σύνολο των αθέμητων εμπορικών πρακτικών που θα απαγορευτούν. Ε, πρόκειται ακριβώς για την βιωσιμότητα της διατροφικής αλυσίδα. Ακούμε πολλά πράγματα για την αλλαγή του κλίματος, βιοπικιλότητα, τα εδάφη και τα ύδατα. Και ο κύριο Δεκάστρο είχε δίκιο όταν είπε ότι το τρέχον σύστημα λειτουργεί με τρόπο λανθασμένο και καταλήγει στο να έχουμε χαμηλή ποιότητα και τιμές. Οπότε καλωσορίζω το πρώτο αυτό βήμα προς μια πιο βιώσιμη διατροφική αλυσίδα. Η Άρλα μας λέει ότι θα προχωρήσει προς μια πιο βιώσιμη γεωργία και ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να την επιβραβεύσουν. Ελπίζω να συμβεί αυτό και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ καταναλωτών και αγροτών να φροντίσουν οι αγρόντες να έχουν μια βιώσιμη τιμή για τα προϊόντα τους. Είχα και εκπροσώπους την προηγούμενη εβδομάδα των Ιρλανδών αγροτών και ζητήσαμε για, συζητήσαμε με για ζητήματα ευζοίας, περιβάλλοντος και πραγματικά ε, απευθύναν έκκληση για τι λέγανε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να βρουν άκρη. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας ακούσατε όταν οι άλλοι δεν ακούαν και νομίζω ότι μαζί θα κάνουμε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαγκίνης για τους σοσιαλιστές και οι δημοκράτες τώρα ο Νικόλα Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ επίτροπε. Με την οδηγία για τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στις αλυσίδες διατροφής φτάνουμε επιτέλους ε, ε, αποτελέσματα που περιμένουμε 10 χρόνια και συγχαίρω τον εισηγητή κύριο Ντεκάστρο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε ε, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο τριμερή διάλογο βελτιώνει σημαντικά την προστασία των γεωργών για τις μικρές και μεσαίες ε, αγροτικές επιχειρήσεις, ε, αυξάνει τις παράνομες, τις αθέμπτες πρακτικές που απαγορεύονται, που οδηγούν από την ακύρωση τελευταία στιγμή των παραγγελιών μέχρι τις μονομερείς τροποποιήσεις των συμβολέων από πλευράς των μεγάλων επιχειρήσεων αγορών. Αυτό ε, που ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της οδηγίας είναι η ανώνυμη καταγγελία, επιτρέποντας την ε, έρευνα χωρίς να εμφανίζεται η ταυτότητα του καταγγέλλοντος, ε, που είναι συχνά πολύ ευάλωτος. Οι κανόνες που περιλαμβάνει η οδηγία υποκαθιστούν την αξιοπρέπεια του, της αγροτιάς της Ένωσης, φέρνοντας τους γεωργούς στο ίδιο επίπεδο με τους ε, μεγάλη με τις μεγάλα, μεγάλα κέντρα διανομής. Ευχαριστώ. Τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, η κυρία Μακιντάερ. Ευχαριστώ. Επί πολύ καιρό βρίσκονταν σε επισφαλή θέση η γεωργοί στην ε, αλυσίδια εφοδιασμού τροφίμων ε, και για πολύ καιρό οι μεγάλοι λιανοπολιτές μπόρεσαν να καταχραστούν την ε, ισχυρή τους θέση. Αυτή η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές χρησιμοποιεί ως βάση της τον κώδικα πρακτικής του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι νομικά δεσμευτικός κώδικας το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψε ότι τα προαιρετικά συστήματα δεν λειτουργήσαν καλά. Οι προαιρετικοί κώδικε συμπεριφορά ε, δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά και γι' αυτό χρειάζεται δεσμευτική νομοθεσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μα Παόλο Δεκάστρο και του άλλου εσκιώδει εισηγητέ, καθώ και τον Επίτροπο Χόγκαν για τη δουλειά που έκαναν πάνω στην οδηγία αυτή για να ε, έχουν σωστή μεταχείριση οι γεωργοί μας. Ε, κατόπιν ε, επιμονής του Κοινοβουλίου η οδηγία αυτή περιλαμβάνει όλα τα γεωργικά προϊόντα, όχι μόνο τα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα τα άνθη, τα οποία είναι εξίσου αλλοιώσιμα με με, τον, ε, με τα τρόφιμα. Καλύπτονται έτσι όλοι οι γεωργοί της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι καλύπτονται οι επιχειρήσεις με μέχρι, με κύκλο εργασιών μέχρι 350 εκατομμύρια. Στον κόσμο μετά το Brexit θέλουμε να διασφαλίσουμε την συνεχή προστασία και των ε, γεωργών ε, του Ηνωμένου Βασιλείου όταν θα πολλούν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να στήξω την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Άλτε ε, Κατάινεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Ντεκάστρο και όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για, αυτό το, για να πετύχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο που σημαίνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να κλείσουμε ένα σύνθετο φάκελο χωρίς ε, να χάνουμε τις προθεσμίες μας. Τα τα θέματα γεωργίας, ε, τα θέματα θέμη του ανταγωνισμού πάντα είχαν δημιουργήσει, είχαν προβλήματα στην αλυσίδια φύση, ιδίως για τους γεωργούς που ήταν οι πιο ευαίσθητοι και που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν συχνά περικοπές. Ξέρω ότι ζητούμε όλο και περισσότερο να σέβονται τους κανόνες αγοράς. Αλλά τι, σημαίνουν τι σημαίνει αυτή η οδηγία ουσιαστικά για τον για τον παραγωγό. Πρώτα πρώτα, ο παραγωγό μπορεί να κάνει καταγγελίε στις αρχέ τη χώρας του, έστω και αν ο αγοραστή ή ο συναλλασσόμενο προέρχεται από τρίτη χώρα και ασκεί αθέμητες εμπορικέ πρακτικές. Αυτό διασφαλίζει και βελτιώνει τις εξαγωγές. Δεύτερον, υπάρχει ένα αποτρεπτικό στοιχείο στην οδηγία αυτή, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κυρώσεις κατά των αθέμητων αυτών πρακτικών. Τρίτον, περνάμε λοιπόν ένα μήνυμα και στα εθνικά κοινοβούλια που νομοθετούν και πρέπει να νομοθετήσουν και πηγαίνοντα παραπέρα και από τα, τις διατάξεις της οδηγίας. Ελπίζω να υποστηριχθούν οι ρυθμίσεις αυτές από όλους σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για τους πράσινους, η κυρία Χόιμπουχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει έναν ενιαίο κανονισμό για να περιορίσει την δύναμη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ τον Πάολο και όλους τους συμμετέχοντες για την πολύ καλή συνεργασία τώρα. Το σημαντικό είναι να μην καθίσει να παρακολουθεί η Ευρώπη γιατί δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Οι αγρότες και οι εργάτες στα χωράφια, στα θερμοκήπια, οι εργάτες στα σφαγεία. Όλοι αυτοί υφίστανται πιέσεις από διαφορετικές πλευρές, όχι μόνο από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και από την πλευρά ε, των ε, αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών, ε, ζυζανιοκτώνων. Χρειάζεται λοιπόν και εκεί πέρα να δούμε κάτι, γιατί υπάρχει μια συγκέντρωση της αγοράς. Σε τελευταίο παράδειγμα η συγχώνευση Bayer Monsanto. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν ένα δίκαιο εισόδημα οι αγρότες, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται και με τα αγροτικά εφόδια και να καταπολεμήσουμε και εκεί τη συγκέντρωση της ε, αγοράς. Και αυτό γίνεται μόνο με ρύθμιση του δικαίου του ανταγωνισμού. Κύριε Χόγκαν θα πρέπει ε, να δείτε το θέμα αυτό. Είστε διατεθειμένοι να το κάνετε. Είστε διατεθειμένοι σε προσεχείς συγχωνεύσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία αλλά και το εισόδημα των αγροτών να τα λάβετε αυτά υπόψη. Γιατί ακριβώς αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση Μονσάντο Μπάιερ. Θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη. Και εδώ μπορούμε να κινηθούμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ΓΚΟΕ, ο κύριος Μακάρθη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι ντροπή ότι αυτοί που ε, παράγουν ε, το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μας να λαμβάνουν το λιγότερο κέρδος και η κατάσταση αυτή χειροτερεύει συνεχώς. Εργάζονται με όλο και πιο περιορισμένα περιθώρια κέρδους και συχνά με ζημία. Επιτέλους, ε, λοιπόν, ε, προσφέρουμε μια νομοθεσία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που θα ε, εξισορροπήσει πάλι την πλάστιγκα. Αυτή ήταν μια ευκαιρία, την οποία όμως δυστυχώς χάσαμε και δεν μπορώ να στήριξω την πρόταση αυτή, διότι δεν πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση των γεωργών με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. μπορούν ε, να συνεχίσουν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές εφόσον τα σούπερ μάρκετ τις ε, συμπεριλαμβάνουν ε, στις συμβάσεις. Ελπίζω να αλλάξει την κατάσταση η νομοθεσία αυτή. Φοβάμαι όμως πως όχι και φοβάμαι ότι θα επανέλθουμε στην πρόταση αυτή, διότι αλλιώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε γεωργούς να εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές. Χρειάζεται μια πιο φιλόδοξη πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ από το EFDD Μάρκο Τσούλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Η έγκριση της οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπρο. Μπορούμε να έχουμε μια αναδιανομή της οικονομικής αξίας πιο δίκαιη στην ε, αλυσίδα εφοδιασμού τροφινών, δίνοντας ε, ε, καλύτερο εισόδημα στις μικρές επιχειρήσεις και καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται. Η οδηγία ήταν οφειλόμενη για να αποκαταστήσει την ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις, προστατεύοντας αυτούς που λόγω του μικρού τους μεγέθου παραμερίζονται συχνά από τις καταχρήσεις των μεγάλων. Ε, η, υποχρέωση, συμβατική, η υποχρέωση ε, υποχρεώνει τις μικρές επιχειρήσεις να υποκύπτουν σε πιέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Χάρη στους σαφείς κανόνες που δίνει οδηγία τώρα, ε, ε, καταδικάζονται ξεκάθαρα αυτές οι εμπορικέ πρακτικές και των ε, επιχειρήσεων χωρίς των ανενδίαστων επιχειρήσεων εις βάρος των μικρών γεωργών. Όταν κυρών, όταν κυρώσεις και α, να καλούνται οι εθέμητες αυτές πρακτικές βελτιώνεται το πλαίσιο. Η πληρωμή οι υπηρεσιών που δεν, που δεν παραχωρούνται οδηγούν σε απόκτησε εκ νέου τις αξιόπιες των μικρών επιχειρήσεων προς όφελος ολόκληρου του κλάδου της γεωργίας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας των Εθνών, ο κύριος Άγνιο. Καλησπέρα σας ε, κύριε Επιτροπέ. Ε, μήπως καθυστερήσατε επειδή προσγειώνεται η Τερέζα Μέη και σας είχε πάρει κατά μέρο ε, για να στηρίξετε την αποχώρηση και της Ιρλανδίας για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως είναι υπερβολικό αυτό. Ίσως αναρωτιέστε, καθώς έχουν απομείνει 18 μέρες, ε, τι κάνω εγώ εδώ πέρα ε, ως Βρετανός Ευρωβουλευτής. Ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η σημαία θα είναι εδώ και σε ένα χρόνο, το πιστεύω. Γι' αυτό θα ήθελα να πω κάτι για την έκθεση αυτή. Χαίρομαι για το συνέστημα της, αλλά με ανησυχεί το ότι έχουμε την κυρία Κριστίν Τέικον στην Βρετανία, η οποία είναι η συνήγορος ε, για τα θέματα αυτά και φοβάμαι ότι θα υπονομευτεί η δουλειά της γιατί θα τους πούν τα σούπερ μάρκετ «Α, ναι, ξέρετε κυρία Τέικον, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει το χ και το ψ» και θα πάνε στο δικαστήριο να υπονομεύσουν το έργο της. Το προσωπικό σας με έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό δεν θα συμβεί, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια η Κομισιόν κατά φρικτό τρόπο πάντα φροντίζει να υπερισχύει η νομοθεσία της, ε, της Βρετανικής νομοθεσίας. Αποδείξτε μου ότι κάνω λάθος. Εγώ προτιμώ αυτό το οποίο έχουμε ήδη στη Βρετανία. Σας ευχαριστώ κύριε Άγνιου. Ο κύριος Επίτροπος ήρθε πάνω στην ώρα και ήταν ιδιαίτερος ε, αποτελεσματικό και ήμασταν και αποτελεσματικοί υπό την ε, προεδρία της κυρίας Μαγκίνε. Γι' αυτό τελειώσαμε γρήγορα και τον περιμέναμε μόνο κάτι δευτερόλεπτα. Κύριε Άγνιο, δέχεστε μια μπλε κάρτα από την κυρία Μαγκίνε. Βεβαίω. Ο κύριος Άγνιο ξέρει ότι ε, αντιδρώ σε προκλήσεις. Ε, μην ε, ανησυχείτε για την ε, κυρία Μέη, όμως είναι ισχυρή η γυναίκα. Πάντως είπατε σχεδόν με χαρά ότι θα βρίσκεστε σε ένα χρόνο εδώ. Θα σας λείψουμε αν φύγουμε. Μήπως μας αγαπάτε παρόλα αυτά. Σας παρακαλώ το διευκρινίστε αυτό. Μαρέι, Πολύ ευχαριστώ θα το διευκρινίσω. Αυτό που με διασκεδάζει είναι η απόλυτη ανικανότητα των πολιτικών μας σε τρία χρόνια και κατόπιν από, ε, του δημοψηφίσματος δεν έχουν καταφέρει ε, την αποχώρηση. Αυτό με διασκεδάζει. Ε, έθιξε σε ένα άλλο θέμα και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Α, ναι, είπες ότι η Τερίζα Μέη είναι ισχυρή γυναίκα. Όχι, εγώ μιλώ για την ε, για την κρίση Αλλά, εν πτώση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σόσνιας, μη εγγεγραμμένος. Ο Στέφαν Κισελεύσκη είχε πει κάποτε ότι ο σοσιαλισμός λύνει τα προβλήματα που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα τα κράτη προσπαθούν ε, να συλλέξουν όσο δυνατόν περισσότερους ε, τρόπους, ε, φόρους, οπότε βάζουν χέρι στον τζίρο, επιβαρύνουν τους πάντες, γιατί θέλουν να ξέρουν τι φόρους μπορούν να επιβάλλουν. Οπότε δημιουργείται επιπλέον κόστος, είναι δύσκολο μετά οι επιχειρηματίες να τα βγάλουν πέρα, νέοι κανονισμοί, συγκεντρώνεται η αγορά είναι εύκολο να αντλήσουν φόρους ε, τα κράτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν επιτρέπεται μετά στους αγρότες να πουλήσουν απευθείας στους ανθρώπους. Μετά έχουμε κακές συμβάσεις και χαμηλές τιμές. Το αποτέλεσμα, ε, λοιπόν, εσείς λέτε ότι δεν είναι να αποσύρουμε αυτόν τον κανονισμό, αλλά να επιβάλλουμε περισσότερους κανονισμούς ε, και ε, περιμένετε να πέσουν τιμές περιμένω και εγώ να δω τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ κύριο Σικερσκή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αν θέλει ο προλαλή σα ε, να με ρωτήσει, να του τα εξηγήσω. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια έχουμε επιτέλους ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες ε, πρακτικές στην ε, διατροφική αλυσίδα. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τον κύριο Ντεκάστρο για την ε, δουλειά που έκαναν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα περάσει σε αυτή τη θητεία. Να ευχαριστήσω επίσης ε, την κυρία Μαγκίνες που είχε προετοιμάσει μια γνωμοδότηση πριν από τρία χρόνια η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ένας λόγος για τον οποίο έχουν ίδια διαπραγματευτική θέση οι αγρότες. Είναι μικρή. Γύρω στο 10% των εκμεταλλεύσεων έχουν την δυνατότητα να είναι μεγάλοι παίκτες στην αγορά. Για να βελτιωθεί λοιπόν η θέση τους στην αγορά θα πρέπει να μπορούν οι αγρότες να ενώνονται σε ομάδες παραγωγών. γιατί με μικρές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούν να οργανωθούν. Επίσης ε, υπάρχει ανάγκη διαλόγου μεταξύ των διαφόρων μερών της ε, διατροφικής αλυσίδας. Φαίνεται ότι ο τομέας της ε, μεταποίησης προτιμάει να μιλάει με τους αγρότες μέσω των ΙΝΙΕ αντί για απευθείας. Αυτό πρέπει να το αλλάξει η Κομισιόν. Λοιπόν, η οδηγία αυτή είναι ένας πολύ εκτεταμένος συμβασμό που επέτυχε ο κύριος Χόγκαν και βεβαίως έτσι είναι οι συμβιβασμοί, δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, παρόλα αυτά είναι μια καλή αρχή. Ας δούμε τώρα αν θα πάει η Εθνική Νομοθεσία παραπέρα και να λύσει και άλλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε Κέρσκι μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σόσνιαρς. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επανειλημμένα είχαμε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου που λένε ότι αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είπατε ότι είναι ασθενής η θέση των γεωργών. Πώς ψηφίζεται λοιπόν όταν το Κοινοβούλιο ε, ψηφίζει προτάσεις για να διατηρήσει την κατάσταση. Απάντηση. Ναι, πράγματι. Ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Ήμουν εισηγητή στην έκθεση για τι μικρέ εκμεταλλεύσει. Πρέπει να στηρίξουμε τι μικρέ επιχειρήσει. Είναι σημαντικέ από μόνε του. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε δει μια ε, διαδικασία ενοποίησης που βελτιώνει τις ευκαιρίες των παραγωγών. Όταν συνεργάζονται μεταξύ τους μπορεί να επηρεάσουν περισσότερο την αγορά, να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην αγορά από ότι ε, ως μεμονωμένη γεωργοί. Είναι μια διαδικασία συνεχιζόμενη και την οποία πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την καλή γεωργική πρακτική, θα πρέπει ε, να στηρίξουμε και τη μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή. Η κυρία Αγγελέρα Γκρασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως όλοι και εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία να ευχαριστήσω τον και να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντεκάστρο και όλους τους σκιώδης ηγητές και από την ΕΜΒΙ και από την ΙΜΚΟ και ιδίω τον Επίτροπο Χόγκαν διότι μετά από 10 χρόνια και άλλα για πρώτη φορά ένας ε, Επίτροπος Γεωργίας το, τολμά να προχωρήσει μια τέτοια οδηγία. Με άλλους δεν ήταν δυνατό. Έχει λοιπόν αξία αυτή η απόφαση που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Υπήρξε ένα μεγάλο λάθος ότι έπρεπε, <coughs> ότι η αλυσίδα διατροφής ήταν καλή, άρα διότι έπρεπε να περιορίσουμε τις τιμές για το καταναλωτή. Αυτό είναι ψέμα η αλυσίδα είναι στρεβλωμένη λόγω αθέμητων πρακτικών που πρέπει να διορθωθούν και πρέπει να προστατεύσουμε τους πλέον αδύναμους. Και αυτό γίνεται. Και ξέρετε, Επίτροπε και συνάδελφε Πάολο, σήμερα πρέπει να περάσει ένα μήνυμα προς όλους. Η Ευρώπη πάει με τους γεωργούς και τους καταναλωτές. Είναι μαζί τους. Αυτό δεν ήταν δυνατό μέχρι τώρα η, το σφάλμα αυτό πρέπει να, να πάψει να υπάρχει και πρέπει, γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε υλοποιώντα πολύ ευρύτερα την οδηγία. Αλλά πρόκειται για ένα πολύ καλό ξεκίνημα και συγχαρητήρια. Ο κύριος Νίκολσον. Ναι, λειτουργεί το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ. Δεν θα περίμενα από τον Παύλο Τεκάστρο μια τέτοια έκθεση. Θα ήθελα να συγχαρώ και όλους όσοι συμμετείχαν στην εργασία και για την ταχύτητα των εργασιών. Η διαπραγματευτική δύναμη των ισχυρών ε, έχει ε, οδηγήσει σε πολύ δύσκολη θέση τους γεωργούς σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό είναι λογικό να εισάγουμε μέτρα προστασίας των μικρών γεωργών. Επί πολύ καιρό βλέπαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε την ε, εξουσία να συγκεντρώνεται στα χέρια των ε, αγοραστών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, έχουν μειώσει το περιθώριο κέρδους των γεωργών. Οι γεωργοί ε, παίρνουν μόλις το 21% της τελικής τιμής του γεωργικού προϊόντος. Τα μέτρα στον τομέα αυτών ε, για τα αλλοιώσιμα είδη θα αποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία για να μπορέσουν οι γεωργοί να συνεχίσουν να παράγουν ε, τρόφιμα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε όταν ολοκληρώσουμε τι εργασίε αυτέ. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχή ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι η λανθασμένη εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών, όχι στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο κρατών μελών. Και εδώ πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Το κλειδί λοιπόν είναι η εφαρμογή και η παρακολούθηση. Ο πρόεδρο σε διακόπτη έχει λήξει ο χρόνο σα. Αλλά ε, ο μιλητή συνεχίζει. Πρέπει να, κάνει, να προχωράει κανεί βήμα-βήμα. Ε, να, πρώτα μαθαίνει κανεί να μπουσουλάει και μετά να περπατάει. Πρόεδρο. Τζαν Κάρλο Σκότα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Ντεκάστρο. Η έγκληση τη οδηγία για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων είναι ένα πρώτο βήμα. Ανεπαρκέ προ την αναγνώριση ενό γεγονότο ότι έχουμε μια εσωτερική αγορά γεμάτη ανισορροπίε μεταξύ περιπίν γεωργών και προμηθευτών και ενδιάμεσων. Α ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αθέμητες πρακτικές αυτών που ε, κυριαρχούν εις βάρος των μικρών που αυτό αυτό συχνά σημαίνει ότι κάποιοι από τους πιο αδενούς είναι υποχρεούνται και καλούνται να πληρώσουν κόστη αποθήκευση, αποθεματοποίησης. Στην Ιταλία έχουμε μια μακρά τέτοια παράδοση όπου ε, οι μηχανισμοί που φερρυπίν καλύπτουν ε, προϊόντα ντόκ όπως το πεκορίνο αλλά και άλλα προϊόντα τα οποία ε, έχουν πολύ χαμηλότερο ουσιαστικό κόστος από το κόστος παραγωγής λόγω της πίεσης των ενδιάμεσων. Υποστηρίζουμε κατά συνέπεια την διάταξη αυτή ελπίζοντας ότι στην επόμενη θητεία θα υπάρξουν ακόμα περισσότεροι κανόνες στην εσωτερική αγορά, ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει με, το, τη σωστή αξία τα γεωργικά προϊόντα και τις διάφορες παραμέτρους της γεωργίας, ιδίως τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντά. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητέ Παόλο, Κάναμε μεγάλο δρόμο. Ο ουσιαστικός στόχος της επανεξισορρόπησης των σχέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίνων και, και η βελτίωση της θέσης των γεωργών ήταν ο στόχος μας. Τα δύο τελευταία χρόνια περάσαμε τρία κείμενα. Τη μεταρρύθμιση του δικαίου ανταγωνισμού στην εφαρμογή του στη Γεωργία, την αναθεώρηση των κανόνων συμβατοποίησης με γραπτά συμβόλαια και την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών. Νομίζω ότι μπορούμε να γυρίσουμε στους γεωργούς με, ψηλό κεφάλι, με ψηλά το κεφάλι. Το θέμα είχε μπλοκάρει εδώ και χρόνια. Ωστόσο το Κοινοβούλιο έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στη μάχη αυτή μπροστά στη, στο φόβο και τη δηλία αλλά και τη διέρεση στο Συμβούλιο. Πρέπει στο μέλλον να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό που είναι εξαιρετικά ουσιαστικό αυτή τη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε χωρίς την ε, κρίση του 16 και την task force ε, της ε, Κομισιόν για την οποία σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, γιατί αυτή η ομάδα εργασία ήταν ουσιώδης για να προχωρήσουμε εκεί που φτάσαμε σήμερα. Ένα τελευταίο θέμα παραμένει ακόμα επιτάπητος, η διαφάνεια των αγορών. Η Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό και τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εκ νέου, κύριε Επίτροπε, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο προς όφελος μιας υπόθεσης που και εσείς και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας ευγενό, ευγενής στόχος που τον χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ερίκ Ανδρία. Πατήστε το κουμπί όμως. Ευχαριστώ πρόεδρε. 350 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το εισόδημα ενός γεωργού στους τρεις, στη χώρα μου, τη Γαλλία. 260 γεωργικέ εκμεταλλεύσει εξαφανίζονται κάθε εβδομάδα. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του χρόνου ο κόσμος των επιχειρήσεων της ε, διατροφή αυξάνουν τα κέρδη τους δίνοντας μερίσματα στους ε, μετόχους τους. Αυτό είναι άδικο. Χρειάζεται, το ξέρουμε όλοι, να, ζήσει ο να ζει ο παραγωγός από την παραγωγή του. Είναι αναγκαίο να παρεύουμε και γι' αυτό ευχαριστώ τον Παρόλη Κάστρο, τους σκιώδη συγγητέ και εσάς κύριε Πίτροπε που επιτρέψατε να κλείσει αυτό το φάκελο, αυτός ο φάκελος της οδηγίας. Με μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Όντως πρέπει να αυξηθεί όπως αναφέρθηκε η διαφάνεια, να υλοποιηθεί ένα παρατηρητήριο σε όλο αυτό τον κλάδο. Αλλά η υλοποίηση της οδηγίας αυτής πρέπει να ενθαρρυνθεί και να πιεστούν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν παραπέρα από το κείμενο που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθυστερημένες πληρωμές, αλλαγές των συμβάσεων είναι κάποιες από τις πρακτικές που αντιμετωπίζουν καθημερινά η παραγωγή. Και αυτή την εβδομάδα ψηφίζουμε να τις απαγορεύσουμε. Ένα σημαντικό βήμα και θα ήθελα και να συγχαρώ τον ε, εισηγητή, τους και οδησηγητές και τον Επιτροπό. Θα πρέπει λοιπόν οι παραγωγοί να μπορούν να κάνουν εμπιστευτικές καταγγελίες. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία και να υπάρχουν υπηρεσίες που να επιλαμβάνονται. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε ε, μια υπηρεσία η οποία θα είναι ανεξάρτητη και θα μπορεί να λαμβάνει μέτρα, θα έχει την εμπιστοσύνη του κλάδου και θα έρχεται να ακούει το τι πραγματικά συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Φιλίπ Λαζό. Ευχαριστώ. Η έκθεση για τι αφέμετε εμπορικέ πρακτικέ στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στετσίδε φοδιασμού τροφίων έρχεται επιτέλου στην Ολομέλεια. Χρειάστηκε ένα χρόνο από τη δημοσίευση ε, τη νομοθετική πρόταση επιτροπή για να μπορέσει να ψηφιστεί το κείμενο αυτό στο Κοινοβούλιο παρότι καθυστερήσαμε για την έγκριση της ε, έκθεσης, οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε βελτίωση της κατάστασης και του κινέμου. Αυξήθηκε ο αριθμός των αθέμητων πρακτικών. Αγοραστέ από τρίτε χώρε προστέθηκαν στο πεδίο επαφαρμογή οδηγία. Οι οργανώσεις παραγωγών και οι αντιπροσωπευτικέ ενώσει έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία εξ ονόματο παραγωγών. Η ταυτότητα των καταγγελόντων προστατεύεται για να μην υφίστανται πιέσεις και τέλος η ο ίδιος ο καταγγέλων θα επιλέξει την, ε, το φόρουμ στο οποίο θα ε, θα εξεταστεί η καταγγελία του. Γι' αυτό υποστηρίξαμε εμείς ε, την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Γεωργία και θα την υποστηρίξουμε στην Ολομέλεια. Η δουλειά βέβαια μπορεί να βελτιωθεί. Το έργο μπορεί να βελτιωθεί μέχρι ότου ε, υποκαταστήσουμε την θέση των γεωργών. Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια λύση θαύμα. Παρά τις προσπάθειες κάποιων χωρών όπως η Γαλλία για το θέμα αυτό, διαπιστώνουμε ότι παραμένει η επίδραση ε, η εξαιρετικά αδύναμη επίδραση των παραγωγών στις εμπορικές σχέσεις. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των γεωργών, κάτι που είναι εξαιρετικά αναγκαίο για τη διατήρηση ολόκληρου του κλάδου. Ευχαριστώ. Μπούντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Χόγκαν και τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους. Η Κομισιόν παρακολουθεί ε, εντατικά τις ε, αθέμητες πρακτικές των ε, μεγάλων παικτών της αγοράς οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα. Η μικρή παραγωγή συχνά είναι θύματα αυτών των καταχρηστικών πρακτικών. Αναβάλλονται οι πληρωμές, μονομερείς αλλαγές ε, συμβάσεων, επέκταση του πεδίου ε, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν για να καλύψει όλους τους συμμετέχοντες ε, στην αγορά για να προστατευτούν οι αγρότες ε, και να παράγουν προϊόντα υψηλής αξίας σε προσιτές τιμές για να οδηγηθούμε σε μια σταθεροποίηση των τιμών ε, έτσι ώστε να εκπροσωπηθούν ε, τα συμφέροντα 11.000 αγροτών και 300.000 συνεργατών και επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης οι Ρουμάνοι αγρότες να πιστούν για την ανάγκη των ενώσεων παραγωγών. Θα πρέπει λοιπόν η εφαρμογή των ε, μέτρων αυτών σε εθνικό επίπεδο να είναι συνεπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Γκαμπριέλα Ζωάννα έχει κατόπιν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη και μέσω αυτής της ε, θέσης ισχύω ε, και των αθέμητων εμπορικών πρακτικών ε, δημιουργούν πολλά προβλήματα. Διαπιστώνουμε συνεχώς ότι υπάρχουν μεγάλες αδικίες και όσον αφορά τη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ αγροτών ε, και εμπόρων και διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλοι και ισχυροί αλλάζουν κάποιες ρήτρε ε, ή τις επιβάλλουν. Βεβαίω, ε, αν συμφωνούν και οι δύο πλευρές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά εδώ πέρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, στις οποίες ε, αναγκάζονται οι αγρότες να υπογράψουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν σαφείς συνθήκες στις συμβάσεις. Πρέπει όλοι να φροντίσουμε να τηρούν οι έμποροι τις ε, προδιαγραφές ε, και να αποφεύγονται οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Νοτσέντο Λεοντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να εκφράσω την εκτίμησή μου για την σκληρή και αποτελεσματική δουλειά του συναδέλφου Ντεκάστρο. Το κείμενο που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο για την πρόταση οδηγία σε ό,τι αφορά τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ένα εργαλείο θεμελιώδου σημασία και οφειλόμενο σε ένα πλαίσιο γεωργικής πολιτικής που προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά. Η καλή διαχείριση της αλυσίδας διατροφής ε, είναι σημαντική, ιδίως για τους μικρούς γεωργούς που είναι ιδιαίτερα τροτοί έναντι αθέμητων πρακτικών, γιατί συχνά στερούνται συμβατικής δυνατότητας που έχουν αυτοί οι εταίροι τους, οι αντισυμβαλόμενοι. Τούτο οφείλεται στι περιορισμένε εναλλακτικέ που έχουν για να προωθήσουν στον τελικό καταναλωτή τα προϊόντα του και στι διαφορετικέ ελλείψει του συστήματο. Η οδηγία προσπαθεί να πλήξει τις αθέμητες πρακτικές με την εισαγωγή μέσων προστασία από κοινού σε όλη την Ένωση και που απαριθμεί τι απαγορευμένε πρακτικέ. Ο στόχος είναι σωστός και θα τύχει της θετικής υποστήριξης από πλευράς μας προσπαθώντας γιατί προσπαθεί να πετύχει έναν από τους βασικούς στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής, την προστασία των γεωργών. Αυτό είναι σημαντικό και για τους Ιταλούς και ιδίω τους Σικελούς γεωργούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση Ντεκάστρο επιδιώκει να καταπολεμήσει τις αθέμητες πρακτοχέ των μεγάλων δομών διανομής που πιέζουν και επιβάλλουν δεσμεύσει στους μικρούς γεωργούς. Αυτό, γι' αυτό θα την υποστηρίξω. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει των ευθυνών της την Ευρωπαϊκή Ένωση που στη σημερινή κρίση οδηγεί τους γεωργούς στην απελπισία και στην αυτοκτονία μερικές φορές. Οι, οι δυνατότητες που έχουν οι, μεγάλοι, οι μεγάλες χώρες γεωργίας όπως Καναδάς, Νέα Ζηλανδία ε, ε, είναι εις βάρος μας οι γεωργοί μας πρέπει να σεβαστούν μια σειρά εργατικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών καμονών που δεν επιβάλλονται στους γεωργούς των άλλων χωρών. Αυτός ο τρελός υπερφιλελευθερισμός οδήγησε την Ένωση να, μειώ, να, να καταργήσει τις ποσοστώσεις στο γάλα και τη ζάχαρη πρόσφατα. Εμείς, ε, βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού, αντισταθήκαμε σε αυτή την κατάργηση και έχουμε δίκιο, διότι βλέπουμε τώρα τις φρικτέ ε, φρικτές συνέπειες οι, ε, δύο, ε, δύο επιχειρήσεις παρασκευής ε, ζάχαρης στη Γαλλία έκλεισαν ε, οδηγώντας σε απολύσεις 132 παραγωγών ζάχαρης και, και 1320 παραγωγών τεύτλων. Οι Βρυξέλλες πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να, διορθώσουν την ε, πολιτική τους υποστηρίζοντας ένα νέο πλαίσιο γεωργικής πολιτικής, ε, την οικογενειακή ποιοτική παραγωγή εις βάρος της μαζικής παραγωγής που, είναι, που πλήττει και την υγεία μας. Ευχαριστώ. Σβάμπ. Λείπει όμως ο κύριος Σεράου Σάντος έχει το λόγο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάολο Δικάστρο για τις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο. Για τους γεωργούς αυτή η οδηγία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Θα βελτιώσει τη θέση τους και θα τους προστατεύσει από τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Τώρα θα υπάρχει ελάχιστο επίπεδο προστασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που θα ξεπερνάει την προστασία που παρήχε μέχρι τώρα η Πορτογαλία, για παράδειγμα. Ε, αποφασιστικός ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχει διευρυνθεί σημαντικά ο κατάλογος των ε, αθέμητων πρακτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόκοβιτς. Please wait Κύριε Σπάπ, παρακαλώ περιμένετε λίγο. Ο κύριος Μπόγκοβιτς, ευχαριστώ πολύ. Στο εμπόριο βλέπουμε εκμετάλλευση των μικρών γεωργών, ε, μεγάλες τάσεις συγκέντρωσης και τα προβλήματα των καταναλωτών ε, έχουν ενώσει το Κοινοβούλιο. Με την υπερψήφιση της έκθεσης αυτής επιβεβαιώνεται και το ψήφισμα της κυρίας Μακίνες. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη δική σας συμβολή. επιδείξατε τόλμη και επιμονή. Με την πρώην συνάδελφό μας, την κυρία Κέστιγκερ, ε, από πλευράς της Αυστριακής Προεδρίας, Εργαστήκατε γρήγορα ώστε να έχουμε την πρόταση αυτή. Τώρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη εντός δύο ετών να μεταφέρουν στην ομοθεσία τους την οδηγία αυτή, ώστε να προστατευτούν οι γεωργοί και οι καταναλωτές. Πολλές ε, αντίστοιχες οδηγίες ήδη έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Στο μέλλον θα μπορούμε έτσι να έχουμε μια βιώσιμη αλυσίδια εφοδιασμού τροφίμων. Πολλοί γεωργοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ε, τον τομέα λόγω της ε, κακής κατανομής του κέρδους. Μόλις το 21% της τιμής του τελικού προϊόντος ε, φτάνει στον γεωργό και αυτό είναι καταστροφικό μήνυμα θα πρέπει να καλέσουμε τους εμπόρους ε, να φροντίσουν για καλύτερη κατανομή του κέρδους στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μωρά. Είναι εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι. Παντού στην Ευρώπη ο γεωργικός κλάδος ζει αβέβαιες στιγμές. Γι' αυτό θέλω και εγώ να συγχαρώ την εξαιρετική δουλειά του συναδέλφου Παύλο Ντεκάστρο με την υποστήριξη Επιτροπής. Συγχαρητήρια για αυτή τη συμφωνία που βρέθηκε μεταξύ των διαφόρων πλευρών που θα επιτρέψει στους γεωργούς να ζήσουν καλύτερα τον καρπό της δουλειάς τους και για προϊόντα που ε, είναι αλλοιώσιμα και για τις συμβατικές υποχρεώσεις. Ε, όπως ξέρετε, σήμερα οι γεωργοί της Ένωσης κερδίζουν το 1 τέταρτο της αξίας του γεωργικού προϊόντος. Αυτό το ποσοστό είναι παράλογο και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Αν θέλουμε να περάσουμε στην οικολογική γεωργική παραγωγή πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τις σχέσεις ισορροπιών μεταξύ των προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων. Γι' αυτό το κείμενο αυτή τη ιδιαίτερα αναμενόμενης οδηγίας είναι ένα καλό βήμα για, την, ναι, για τις νέες ισορροπίες και θέλω να εκφράσω την ευχή η οδηγία αυτή που δεν σταματά στα σύνορά μας άλλωστε να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, με βάση τις πολιτικές ομάδες βλέπουμε τα ονόματα, θα το διορθώσουμε. Αυτό ο κύριος Κάρας ε, έχει το λόγο τώρα. Έχω 1,5 λεπτό, ζήτησα να μιλήσω και μου είχαν δώσει 1,5 λεπτό. Ήμουν στον κατάλογο. Είμαι στον κατάλογο. Αλλά με ξεχάσατε. Θα το τσεκάρουμε. Συνεχίζουμε. Όπως έχω τα στοιχεία. Με βάση... Η κυρία Ριμπέιρο έχει το λόγο με βάση το δικό μου πρόγραμμα. Θα το τσεκάρουμε όμως, μην φοβάστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η θητεία μας φτάνει στο τέλος της. Οι πολίτες μας κοιτούν και Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδια ε, φοδιασμού τροφίμων. Εδώ και χρόνια έχουμε εργαστεί πάνω στο θέμα αυτό. Επιτέλους όμως ε, είδαμε αρκετή πολιτική βούληση ώστε να έχουμε μια οδηγία που να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους γεωργούς ε, και για να ε, εμποδίσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πρόκειται για σημαντική μέρα για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Απαγορεύονται λοιπόν ε, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές όπως είναι οι σε τροποποίηση των ε, συμβάσεων, η μετακύληση ε, των ζημιών στους γεωργούς για τα αλλοιώσιμα προϊόντα, κυρώσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην γραπτή σύμβαση. Είναι λοιπόν σημαντικό το βήμα προόδου, ιδιαίτερα για τις μικρές αγορές ε, όπου ε, δεν ε, υπάρχει ανωνυμία των διαφόρων φορέων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει λοιπόν περισσότερη προστασία στον Ευρωπαϊκό Γεωργό, γι' αυτό είναι καλή μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σημερινή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Οθώνουμε τα ονόματα στον πίνακα και θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Τζουφρίντα. Είναι πυλώνα, η Γεωργία είναι πυλώνα στην Ένωση, ωστόσο όλο και πιο συχνά υπόκειται σε κατηγορίες διότι οι γεωργοί μας ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα διαρθρωτικού χαρακτήρα και κόστους αλλά και αθέμητων πρακτικών από πλευράς των ε, επιχειρήσεων διανομής. Είναι η πιο αδύναμη κρίκη στην αλυσίδα και συχνά στρέφονται κατά της Ευρώπης και εναντίον μας που τους εκπροσωπούμε. Με την οδηγία αυτή αποδεικνύουμε ότι εν τέλει είμαστε με την μαζί τους με τους γεωργούς, με τους παραγωγούς, με τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Με τις περιφέρειες όπως τη δική μου, τη Σικελία που ζει από τη γεωργία και που έχει εκατοντάδες προϊόντων αριστείας που πρέπει να προστατεύονται. Αύριο αυτό θα καταστεί δυνατό χάρη στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο αντιπρόεδρο μα Ντεκάστρο στην Επιτροπή και όλοι εμεί όσοι παλεύουμε για χρόνια προ όφελο των γεωργών και προασπίζοντα τη δική μα γεωργική παραγωγή. Ο κύριος Κάρας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κύριε και κύριοι. Το δικό μας ευρωπαϊκό μοντέλο είναι η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτό σημαίνει η ρύθμιση της αγοράς. Σημαίνει να ρυθμίζουμε την αγορά σε μια κατεύθυνση ώστε να προστατεύουμε τους μικρότερους συμμετέχοντες στην αγορά για να μην έχουν μειονέκτημα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ πέρα. Πού απαγορεύουμε τις αθήνητες πρακτικές. Τελειώνουμε με τις ε, πρακτικές αυτές ε, που είναι εις βάρος ε, των γεωργών και άλλων εξαρτημένων προμηθευτών. Και τελειώνουμε με τις πρακτικές αυτές των καθυστερημένων πληρωμών ή την ακύρωση της παραγγελίας τελευταία στιγμή. Γιατί έτσι ε, μόνο θα προστατεύσουμε την ύπαρξη την οικονομική των Γεωργών. Τελειώνουμε επίσης με τις άδικες εμπορικές και μονόπλευρες εμπορικές σχέσεις. Με τον εμποδίζουμε το να μην ε, ε, είναι δυνατή πλέον η προφορική σύμβαση. Και υπάρχει βεβαίως και η δυνατότητα ανωνύμων καταγγελιών από γεωργούς και η δυνατότητα να φτιαχτεί ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Ευχαριστώ λοιπόν την Προεδρία του Συμβουλίου για τα όσα έκανε για να σταματήσουν επιτέλους οι ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Μόλις άκουσα ότι η οθόνη λειτουργεί έτσι ώστε το ΕΛΚ να είναι πάνω-πάνω ανα πάσα στιγμή. Οπότε να με συγχωρείτε. Εγώ συνεχίζω με τον αρχικό κατάλογο των ομιλητών. Σον Κέλλη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι στην Επιτροπή Γεωργίας. Είμαι όμως Ιρλανδός και η Ιρλανδία είναι σε μεγάλο βαθμό γεωργική χώρα και γι' αυτό με ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Στην πρώτη μου θητεία πριν από αρκετά χρόνια ήμουνα σε μια συνάντηση με ε, την ε, ε, Μέιραντ Μακίνες, με την Αν Μαρή Κοράτσα Βίλτ και ο Επίτροπος Χόγκεν ήταν εκεί και είπε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ε, πολλοί δεν τον πίστεψαν τότε, θεώρησαν ότι είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι το έχει πετύχει και να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα ε, τα θέματα των αθέμητων πρακτικών που συμπεριλαμβάνουν τις πληρωμές τα αλλοιώσιμα τρόφιμα κλπ. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ο συνάδελφος Νίκολσον είπε ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πραγματι είναι, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή στα κράτη-μέλη ώστε ε, να διασφαλίσουμε τα ωφέλη για τους γεωργούς. Ε, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, τιμές που πέφτουν και το Brexit, ε, πρέπει να φροντίσουμε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουν τους γεωργούς. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο ε, θα ισχύει και στην περίπτωση του Brexit, ε, παρόλο που ο κύριος Άγνιου δεν πιστεύει σε αυτό. Ελπίζω να έχει δίκιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαριάννα Πέτυρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η δημοσκόπηση που έγινε μεταξύ των παραγωγών για το θέμα αυτό έδειξε ότι η ζημιά από αυτές τις πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ακριβώς αυτές οι αθέμητες πρακτικές ε, εμποδίζουν τους νέους ε, από το να ασχοληθούν με τη γεωργία. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, τότε το μέλλον της γεωργίας πλέον θα αμφισβητηθεί. Οι αγρότες είναι ο κλάδος ε, με τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αισθάνονται καθόλου ασφάλεια. Οι ενδιάμεση εδώ είναι η πιο ισχυρή και παρόλα αυτά ρίχνουν το επιχειρηματικό ρίσκο στους ασθενέστερους, στους αγρότες ε, με τις προθεσμίες πληρωμής, με τις συνθήκες αποθήκευσης, στοιχεία δηλαδή τα οποία δεν επηρεάζουν οι αγρότες. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτήν την συμφωνία στο πλαίσιο του διαλόγου και ναι, νομίζω ότι πρόκειται για μια νίκη των μικρών αγροτών και θα διευκολύνει λίγο τη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σβάμπ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε για την καθυστέρησή μου στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά στη Γεωργία, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το έλεγε πάντα η ομάδα του ΕΛΚ και βεβαίως ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τον κύριο Ντεκάστρο. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η οδηγία δεν είναι τέλεια παντού. Γιατί η προστασία που περιλαμβάνεται εδώ πέρα πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τον μέχρι τώρα ορισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα ορισμού, αλλά αν είναι να κάνουμε αυτή την αλλαγή πρέπει να υπάρξει μία μελέτη επιπτώσεων. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουμε έτσι απότομα τον ορισμό των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η οδηγία αυτή ξεκινάει από την υπόθεση ότι υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στα ζητήματα της γεωργίας. Και πηγαίνει έτσι προς την κατεύθυνση της πλήρους εναρμόνισης ε, γιατί αλλιώς όπως αναφέρεται και στα εκτιμώντας 16 και 17 θα πάμε πάλι σε έναν κατακαιρματισμό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σβάμπ, δέχεστε ε, γαλάζια κάρτα από τον κύριο Μόη. Ναι. Παρακαλώ. Όχι. Δεν έχουμε ερώτηση. Από την Επιτροπή Ανάπτυξης, η Λίντα Μακέιβαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν πολλοί, η νομοθεσία αυτή είναι κάτι που ζητάμε εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστώ Επίτροπε Χόγκαν ε, που υποβάλλατε την πρόταση και ευχαριστώ τον Παύλο Δικάστρο που κατάφερε να ολοκληρώσει τις εργασίες πριν το τέλος της θητείας και πριν το Brexit. Μιλώ εκ μέρου τη Επιτροπής ανάπτυξη. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι η νομοθεσία αυτή καλύπτει όχι μόνο τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο νότιο ημισφαίριο, διότι και αυτοί βρίσκονται υπό πίεση όπω οι Ευρωπαίοι γεωργοί και έχουν πολύ λίγη διαπραγματευτική δύναμη. Ε, όταν αγοράσετε μια μπανάνα, το 4 έως 9% ε, παίρνει ο Γεωργός τελικά. Ε, ενώ ε, στο, στο, στον, στα προϊόντα του κοκοφίνικα έχουν πέσει οι τιμές κατά 30-40%. Πρόκειται για πολύ καλή νομοθεσία. Θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτήν και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους στην Ευρώπη που ζήτησαν την νομοθεσία αυτή, το ε, κίνημα Fair Trade και όλες τις οργανώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που ζήτησαν κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ότι το νέο κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με τα θέματα δίκαιου εμπορίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η επιτυχία των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό αποτελεί μεγάλο, μεγάλη επιτυχία για τους γεωργούς. Δείχνει ότι θέσαμε τέλος στον παράγοντα φόβο. Η αύξηση των πρακτικών που απαγορεύονται επίσης αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολύ περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες ε, απαγορεύονται οι αθέμητες πρακτικές. Φερρυπίν, καθυστερήσει πληρωμών. Η πληρωμή δεν μπορεί να καθυστερήσει ή να μην χορηγηθεί χωρίς αιτιολογία, δικαιολογημένη αιτιολογία. Ζητώ από όλα τα κράτη να υιοθετήσουν κατάλληλα βήματα και μηχανισμούς για να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι στην ημερήσια διάταξη. Γνωρίζουμε ότι στην πράξη δεν υπάρχει δίκαιο εμπόριο. Γνωρίζουμε ότι στην πράξη υπάρχει υπερεκμετάλλευση των αγροτών ακούστηκε άλλωστε ότι οι ίδιοι αγρότες το πολύ πολύ να πάρουν το 20% της συνολικής τιμής που πιάνει ένα προϊόν και αυτό διότι υπάρχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις υπάρχουν οι μεγάλες αλυσίδες διατροφής και διανομής των τροφίμων υπάρχουν οι εκβιασμοί από τον χοντρέμπορα, ο οποίος διαμορφώνει τις τιμές πολλές φορές πληρώνει με επιταγές εν συνεχεία δεν εξοφλεί και όλα αυτά βεβαίως οδηγούν σε μια πλήρη εξάρτηση των αγροτικό κόσμων. γι' αυτό χρειάζεται η πολύ συγκεκριμένη απαγόρευση των αθέμητων πρακτικών η στήριξη των γεωργών μας αλλά βεβαίως αυτό δεν είναι πανάκια. οι αγρότες πρέπει να στηριχτούν και με άλλες πρακτικές και κυρίως να υπάρξουν τράπεζες για να τους δώσουν φθηνές πιστώσεις για να αντιμετωπίσουν το ακριβό κόστος παραγωγής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλτε Βάουτμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χόγκαν. Θεωρώ ότι αυτή η οδηγία είναι απολύτως απαραίτητη για να επιζήσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες. Επιτέλους θα σταματήσουν 16, 16 αθέμητες εμπορικές πρακτικές αγαπητοί συνάδελφοι. Θα προσπαθήσουμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα πεδίο με ίσους όρους ανταγωνισμού. Θα σταματήσουν οι ακυρώσεις παραγγελίας τελευταία στιγμή. Θα σταματήσει η μονομερής αλλαγή των συμβάσεων και η άρνηση να υπογραφούν γραπτές συμβάσεις. Κύριε Επίτροπε, το 2017 το Ευρωβαρόμετρο έκανε μία δημοσκόπηση μεταξύ των αγροτών και 77% αυτών είπαν ότι τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Ελπίζω λοιπόν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή γρήγορα για να στηρίξουμε κάπως τους αγρότες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιγγέλ Βιέγκας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι Πορτογάλοι γεωργοί αυτή τη στιγμή λαμβάνουν μόλις το 20% της τελικής τιμής των προϊόντων τους. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, ενεργούν πολύ επιθετικά και πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές για τους παραγωγούς. Είναι θλιβερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πέντε τελευταία χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ε, τώρα όμως, ε, λίγο πριν τις εκλογές, ε, έχουμε την οδηγία αυτή και κάλιο αργά παρά ποτέ. Η πρόταση αυτή έχει μάλλον κάποιες θετικές πτυχές αλλά δεν απαντάτε το βασικό ερώτημα. Και Επίσης δεν έχουμε καμία εγγύηση για την τήρηση των κανόνων. Ε, έτσι λοιπόν δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα έχουν αξιοπρεπή ζωή οι γεωργοί μας. Ε, μπορεί να αποτελεί καλό βήμα πρόοδου η πρόταση αυτή, δεν εκπληρεί ε, όμως όλες τις επιθυμίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, πρέπει να έχετε σηκώσει η κάρτα για να μιλήσετε στο KTI. Δεν θέλετε. Έχετε τον λόγο. Δέχομαι θετικά την οδηγία αυτή που μετά από τόσα χρόνια εν τέλει προστατεύει τους γεωργούς από αθέμητες πρακτικές των αγοραστών και διανομέων μεγάλων επιχειρήσεων προς όφελος όλης της αλυσίδας διατροφίμων. Μπορώ να σας περιγράψω τι είχε γίνει στη Σαρδινία και από την περιφέρεια από όπου προέρχομαι και να δείξω την αλληλεγγύη μου στην κατάσταση εκεί. Ελπίζω η οδηγία να, ε, να αποκαταστήσει τα δικαιώματα των χιλιάδων ε, γεωργών που δούλεψαν για χρόνια χωρίς δικαιώματα. Αυτά ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Να, σας να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Ντεκάστρο. Η γεωργή και παραγωγή ξέρουμε ότι είναι ευάλωτοι σε αθέμητες πρακτικές. Ο κλάδος της ε, διατροφής έχει μεγάλες ανισορροπίες μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων οι τελευταίες επιβάλλουν ε, κακόπιστες ε, θέσεις και υποχρεώσεις στους γεωργούς εις βάρος εν τέλει των καταναλωτών. Χάρη στην οδηγία που συζητούμε σήμερα, εισάγουμε ένα ελάχιστο ποσοστό προστασία σε όλη την Ένωση με την απαγόρευση 16 θέμητων πρακτικών που επιβάλλονται μονομερώς από τον έναν εταίρο στον άλλον. Καθυστέρηση ε, Πληρωμήσει ή ακύρωση τελευταία στιγμή των παραγγελιών. Τα μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή στην Ένωση των κανόνων και μέτρων που περιλαμβάνει η οδηγία και που έχουν στόχο να προστατεύσουν του γεωργού και να παράσχουν προϊόντα ποιότητα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σετμαλόβα έχει το λόγο, η κυρία Όλγα Σετμαλόβα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υιοθετώντα το πρώτο ευρωπαϊκό μέσο για την προστασία των γεωργών και των μικρών εκμεταλλεύσεων από τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουμε τη διαδικασία που ξεκίνησαν το 2016 η κυρία Μακίνες και ο κύριος Τσέσακ. Πετύχαμε σχεδόν το αδύνατο Θα απαγορεύσουμε λοιπόν τώρα τις παραγγελίες τελευταία στιγμής και δεν θα πρέπει οι ασθενέστεροι να φοβούνται τα τύπινα. Οι αρχές θα πρέπει ε, να συνεργάζονται ε, μεταξύ τους, οι αρχές των διαφόρων κρατών μελών. Ε, θεσπίζουμε λοιπόν δίκες προϋποθέσεις για τους παραγωγούς και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο αποτέλεσμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Hogan. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επικροτώ την ευρεία στήριξη για την συμφωνία που πετύχαμε το Δεκέμβριο και πολύ θα χαρώ να δω η υποστήριξη αυτή να αντικατοπτρίζεται στην αυριανή ψηφοφορία. Ο κύριος Εντεκάστρο έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι αυτή η νομοθετική πράξη ε, θα προστατεύσει τους γεωργούς της Ευρώπης και μάλιστα θα προστατεύσει ε, το 97% των μικρών εκμεταλλεύσεων ε, στον αγροδιατροφικό τομέα. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις ακούσαμε σήμερα από τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος. Μία από τον κύριο Άγνιου που αποκάλυψε ότι το μυστικό που κρατούσε τόσα χρόνια ήταν ότι όσοι συμφωνούν μαζί του καταψηφίζουν την πρόταση της κυρίας Μέη και τελικά θέλουν να μείνουν στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι θα είσαστε εδώ σε ένα χρόνο. Ε, θα καταψηφίσετε την πρόταση αυτή για να παραμείνετε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου δεν ακούσαμε. Θα έχετε, είχατε πολύ χρόνο για να εκφράσετε τις απόψεις σας ε, κατά τη διάρκεια των ετών. Η άλλη θέση ήταν του κυρίου Κάρθη για την νομοθεσία αυτή. Ε, ο οποίος ε, δήθεν μιλά στο όνομα της ε, πολιτικής του ομάδας, ε, κρατάει όμως μια θέση απομονωτισμού. Ε, προστατεύει τους ισχυρούς εις βάρος των ασθενών και ε, με εκπλήσει αυτή η θέση του Sinn Féin ε, που προσπαθούν εδώ και χρόνια να παρουσιαστούν ως σοσιαλιστές. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους ασθενείς απέναντι στους ισχυρούς. θα θεωρούσα ότι την αρχή αυτή μπορεί να την συμμεριστεί το Sinn Féin. με εκπλήσει λοιπόν ε, που ο κύριος Κάρθη βρίσκεται με το μέρος των ε, μεγάλων ε, λιανοπολιτών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει, κύριε Κάρθη, ότι το μέτρο αυτό είναι πανάκια και ότι εν μία νυχτή θα λύσει το πρόβλημα. Είναι όμως ένα σημαντικό μέσο. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν πέρα από την οδηγία αυτή και ελπίζω να το κάνουν αυτό πόσο μάλλον λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε ο κύριος ε, Ανδριώ για την Γαλλία. Με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου αδράξαμε την ευκαιρία και αυτοί που συνεχίζουν να αντίκενται στην ε, νομοθεσία αυτή ε, αποτελούν μία ασύνδετη συμμαχία. Ο κύριος Νίκολσον και η κυρία Γκιλέρα έχουν δίκιο. Προστατεύουμε τους γεωργούς. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε κυρία Μαγκίνες, η κυρία Αγγιλέρα και άλλοι τόνισαν ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία σε απάντηση εκκλήσεων εκτός του Κοινοβουλίου για να προστατεύσουμε τους ε, ασθενείς. Γι' αυτό προστατεύουμε τους γεωργούς στην αγροδιατροφική αλυσίδια, απαγορεύουμε τις αθέμητες πρακτικές και νομίζω ότι η πλειοψηφία ε, είναι υπέρ μας κυρία Χόιπαχ, ε, μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογία. Μπορώ να σας πω όμως ότι έχουμε πετύχει πολλά όσον αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια στη Γεωργία με τον κανονισμό ε, όμνιμπους ε, στην αγροδιατροφική αλυσίδα και στο εγγύς μέλλον ε, θα παρουσιάσω και άλλες ε, τροποποίησεις. Έχουμε μπροστά μας το στόχο, αλλά θα πετύχουμε κάτι μόνο εάν ε, τα κράτη-μέλη αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ε, ο κύριος Νταντέν είπε ότι είναι ευγενής ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τη δουλειά της. Τώρα πια εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή. Ε, κύριε Αντριό και κυρία Ζωάνα και άλλοι, αναφέρατε την πρόταση της Επιτροπής να τονίσω ότι έχει την πλήρη υποστήριξη όλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Γιούνκερ το 2016 είπε ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς είναι δυνατόν το γάλα να είναι πιο φθηνό από το νερό. Ε, επίσης να πω στον κύριο Σφάμπ ότι καταλαβαίνω τις παρατηρήσεις του. Ε, είχαμε μια πολύ πιο φιλόδοξη πρόταση. Ε, πετύχαμε όμως συμβιβασμό τελικά. Επίσης εκπονήθηκε μελέτη αντικτύπου πριν υποβληθεί η πρόταση αυτή. Τίποτα στην ομοθετική αυτή πράξη δεν θα πρέπει ε, να δημιουργεί φόβους σε κανέναν στον αγροδιατροφικό ε, τομέα εφόσον φέρονται δίκαια απέναντι στους γεωργούς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπη. Το λόγο έχει ο κύριος Ντεκάστρο, εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και ευχαριστώ εκ νέου τον, κύριο, τον επίτροπο κύριο Χόγκανγκ που υποστήριξε τις θέσεις μας. Χωρίς αυτή την ομαδική δουλειά δεν θα είχαμε πετύχει συνάδελφοι. Οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση της πρότασης ε, καταφέραμε να έχουμε μια πολιτική συμφωνία το Δεκέμβριο. Θέλω να υπενθυμίσω την ομόφωνη υποστήριξη της πρότασης στο Συμβούλιο Γεωργίας ε, που δείχνει ότι αυτή και την υποστήριξη από όλους τους συναδέλφους και από αυτούς που ήθελαν περισσότερα και από αυτούς λίγοι είναι αλήθεια που δεν ήθελαν καθόλου την ολιγία. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε συνάδελφοι. Μια Ευρώπη που βοηθάει τις αδύναμες επιχειρήσεις, που προστατεύει τον καταναλωτή με κανόνες με διαφάνεια και που εξασφαλίζουν την ποιότητα. Να υπογραμμίσω ακόμα αυτό που είπε η, κυρία, η συνάδελφος κυρία Μαγκίνες. Ένα πρώτο βήμα είναι γιατί και πρέπει να περιμένουμε και την υλοποίησή της. Αλλά τονίζουμε ότι η οδηγία διευρύνει την αποτελεσματικότητα των εθνικών νόμων. Να θυμίσω στον κύριο Άγνιο ότι η, χάρη στην οδηγία οι, οι βρετανικές επιχειρήσεις θα είναι σε καλύτερη θέση, θα είναι προστατευμένες όταν εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μακέβαν που υπενθύμησε κάτι που, για το οποίο είμαστε περήφανοι. Εφαρμόζεται και σε παραγωγούς εκτός Ευρώπης η οδηγία. Η προστασία δηλαδή επεκτείνεται σε όλους τους μικρούς παραγωγούς που υφίστανται αθέμητες πρακτικές εδώ στην Ευρώπη. Εν τέλει, αγαπητέ Επίτροπε Χόγκα, κάναμε με την οδηγία αυτή ένα μικρό θαύμα. Την υποστηρίζουν όλες οι ομάδες με την μία εξαίρεση της συναδέλφου Ματίας. ευχαριστώ όλους και πραγματικά σήμερα είναι μια επιτυχία που θα ήθελα το κοινοβούλιο μας να επαναλάβει και στο μέλλον. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεκάστρο. Ολοκληρώνεται η διαδικασία. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Καλή τύχη. Προχωρούμε τώρα στην εξέταση κοινής, στην κοινή συζήτηση τη σύσταση ε, τη Αντιπροέδρου κ. Χέιντι Χάουταλα για την συμφωνία, εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή τη δασική νομοθεσία στη διακυβέρνηση και το εμπόριο και την ε, δεύτερη έκθεση πάλι τη κυρία Χάλα για την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ σχετικά με την εφαρμογή τη δασική νομοθεσία στη διακυβέρνηση και το εμπόριο στον δασικό τομέα. Το λόγο έχει η εισηγήτρια, αντιπρόεδρος κυρία Χάουταλα. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαιτέρως για το ότι οι εθελοντικές συμφωνίες για την δασοπονία, την διακυβέρνηση και το εμπόριο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνδυασμού εμπορικής συμφωνίας με την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αυτής της εθελοντικής συμφωνίας με το Βιετνάμ με την ε, Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα το κεφάλαιο 13 για την βιώσιμη ανάπτυξη της Συμφωνίας Ελευθερίου Εμπορίου που ακόμα δεν έχει κυρωθεί ε, κάνει αναφορά στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό μέσο για να αντιμετωπιστούν ελλείψεις ε, στον τομέα της διακυβέρνησης όχι μόνο της ε, δασοπονίας αλλά και στο κρατικό σύστημα στο σύνολό του. Μιλάω για τη λειτουργία των ε, τελωνίων, ε, τα κτλ. Το Βιετνάμ είναι η τρίτη χώρα η οποία έχει συνυπογράψει τέτοιες εθελοντικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρίτη ασιατική χώρα. Και αφορά σε αυτό το θέμα την ελάθρο Επισκέφθηκα την χώρα τον Ιανουάριο ως εισηγήτρια και μου τόνισαν ότι το Βιετνάμ σκοπεύει να γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων ξυλίας παγκοσμίω. Αυτό βεβαίω σημαίνει ότι αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτή η συμφωνία. Υπάρχει τώρα ένας νέος νόμος περί δασοκομείας από τον Ιανουάριο που απαγορεύει ξεκάθαρα τις εισαγωγές ε, παράνομης ξυλίας. Οπότε θα πρέπει πλέον να εισάγεται ξυλία παράνομα από την Καμπότζη. Και εδώ πέρα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει και με την Καμπότζη. Ε, αυτό το πρίσμα είναι πολύ ανησυχητικό ότι η οργάνωση Global Witness είδε μια αύξηση στις εισαγωγές από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα υψηλού κινδύνου κάτι το οποίο πρέπει να δούμε στο πλαίσιο της ε, εφαρμογής της εθελοντικής συμφωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν οι παράνομες εισαγωγές. Το να πάει η πηγή σε νέες χώρες υψηλού κινδύνου δεν είναι λύση και αναμένω βεβαίως να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία γρήγορα και αποτελεσματικά και να υπάρξει διαβούλευση με όλους του ενδιαφερόμενου και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει λίγο θόρυβο στην αίθουσα. Συμφωνώ και παρακαλώ του συναδέλφου. Όσοι θέλουν να μιλήσουν να φύγουν από την Ολομέλεια και να μην κάνουν θόρυβο γενικά. Μιλάει η Αντιπρόεδρος κυρία Χάουταλα εξηγώντα την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της θα πρέπει να διασφαλίσει επαρκείς πόρους για να στηρίξει το Βιετνάμ για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι στην διαδικασία σύνταξης ενός σχεδίου δράσης για την αποδάσωση καινοτομίε οι οποίες είναι παρόμοιες με την εθελοντική συμφωνία απαιτούνται ακριβώ για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια πρόκληση της αποδάσωσης. Μια πρόκληση η οποία πλέον γίνεται κρίσιμη καθώς η επιστημονική κατανόηση της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται. Εθελοντικέ αυτέ συμφωνίε είναι σημαντικό κομμάτι τη λύση, λοιπόν καθώ απαιτούνται νομικά μέσα για να καταπολεμηθεί η αποδάσωση παγκοσμίω. και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει ισχυρά μέτρα για να μην υπάρχει αποδάσωση για προϊόντα που εξάγονται προ την Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επί τη ευκαιρία η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα προϊόντα όπω ο καφέ, το κακάο και το φινικέλαιο το Βιετνάμ αντιμετωπίζει βεβαίως ε, ε, πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις αυτής της συμφωνίας, ε, κάτι για το οποίο είμαι βέβαιη ότι θα προσπαθήσει να κάνει με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Δεν μπορεί εδώ πέρα απλά να συμπληρώνουμε κουτάκι. Μόνο όταν το Κοινοβούλιο πιστεί για το ότι έχει σταματήσει η λαθροϊλοτομία θα μπορέσουν να δοθούν άδειε στο Βιετνάμ. Σας ευχαριστώ. Δεν σας διέκοψα νωρίτερα γιατί δεν ήθελα να εμποδίσω την πορεία της σκέψης σας αλλά να αμέσω μόλις ε, το σχολιάσατε κι εσείς. Δίνω αμέσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, αντιπρόεδρο κύριο Άντσιπ. Σας ευχαριστώ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συμμετάσχω στη συζήτηση που ολοκληρώνει την... Ε, Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Επίτροπος. Ζητώ συγγνώμη διότι αντικαθιστώ και ένα συνάδελφο και ε, μπέρδεψα τις σημειώσεις μου. Ζήτω συγγνώμη. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. η εθελοντική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Βιετνάμ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στι σχέσει μα με το Βιετνάμ και σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της παράνομη υλοτομία και αποδάσωση. καθώς και επιβεβαίωση Τη εγκυρότητα του μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα δάση, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο. Είναι η πρώτη συμφωνία ε, εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση, που είναι όχι μόνο σημαντικό εξαγωγέ, αλλά και σημαντικό εξαγωγέα ξυλία. Το Βιετνάμ βρίσκεται στο επίκεντρο του Παγκοσμίου Εμπορίου Προϊόντων Ξυλίας και γι' αυτό η θελοντική Συμφωνία εταιρική Σχέσης με το Βιετνάμ ε, όταν αρχίσει να λειτουργεί πλήρως ε, θα έχει σημαντικό θετικό ε, αντίκτυπο και πέρα από τα σύνορα της χώρας επιφέροντας κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη στους ανθρώπους του Βιετνάμ. Χαίρομαι που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με την αξιολόγηση αυτή. Μάλιστα φαίνεται ότι ε, συμφωνείτε και με τα δύο ψηφίσματα που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Μπορώ να συμφωνήσω με τα, τις βασικές παρατηρήσεις των εκθέσεων. Το Βιετνάμ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Μία σημαντική επιτυχία ήταν ε, η ανοιχτή και επικοτομητική συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων στη διαδικασία. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχίσει και στην φάση εφαρμογής της συμφωνίας. Το Βιετνάμ θα ε, επιβάλλει υποχρεωτικές, υποχρεωτικά μέτρα δέουσας επιμέλειας και Γνωρίζουμε ότι θα είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε η εφαρμογή να συνάδει με τα υψηλά πρότυπα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ξυλία. Το θέμα της νομιμότητας των εισαγωγών και ιδιαίτερα αυτών από την Καμπότζη βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης και δικαίως ε, συμβαίνει αυτό. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την διαδικασία. Ωστόσο, θα πρέπει να σα θυμίσουμε ότι οι έλεγχοι των εισαγωγών αποτελούν ένα μόνο στοιχείο ενός ολοκληρωμένου συστήματος που στόχο έχει να διασφαλίσει την νομότητα της ξυλίας και πέρα από τα σημεία εισαγωγής. Ε, η επεξεργασία, το εμπόριο και οι εξαγωγές επίσης καλύπτονται. Τέλος, ε, η επιτυχία της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ε, θα μετρηθεί κατά την εφαρμογή του συνολικού συστήματος. Δεν μπορεί να υπάρχει επιβολή του νόμου για τα δάση, ούτε αδειοδότηση των εξαγωγών χωρίς να συμβαίνει αυτό. Επικροτώ το θετικό μήνυμα από πλευράς των ε, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, προσβλέπω στη συνέχιση της ε, συζήτησης πάνω σε αυτήν την συμφωνία ορόσημο. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή Ανάπτυξης τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ζαχραντήλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγητής ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, στήριξα πλήρως ε, την εθελοντική αυτή συμφωνία με το Βιετνάμ. Είναι αναγκαία και χρήσιμη, καινοτόμος και με ε, λογικό μηχανισμό. Ξέρουμε πω το Βιετνάμ εξάγει προϊόντα ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλε χώρε στην Ιαπωνία, την Κίνα. Και η συμφωνία αυτή θα αποτελεί ένα αποτελεσματικό ε, μέσο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και προώθησης του αϊφόρου εμπορίου ξυλία. Να τονίσω κάτι. Χαίρομαι για την σύναψη της συγκεκριμένης συνθήκης, αλλά ανησυχώ από την άλλη για την ε, άλλη συνθήκη τη συνθήκη ελευθερία εμπορίου. Έχουμε σοβαρέ καθυστερήσεις και περιπλοκές και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να πιέσει λίγο την Ρουμανική Προεδρία για να προχωρήσουμε και με την άλλη συνθήκη να την ψηφίσουμε πριν από τις ευρωεκλογές το Μάιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Ζάχραντιλ. Ε, τώρα Ξεκινάμε με τις ε, παρεμβάσεις εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Βαλέσα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε άλλη μια εμπορική συμφωνία, η τελευταία αυτή της ε, θητείας μετά την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Χαίρομαι πραγματικά που ανοίγουμε τις αγορές μας σε εμπόριο υψηλών προδιαγραφών. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ των εμπορικών ε, συμφωνιών καθώς ε, προωθούν την διεθνή διαγωνιστικότητα των εταιριών μας και δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το ότι έχουμε ήδη πάνω από 70 τέτοιες εμπορικές συμφωνίες ε, Βεβαίω, προωθούμε την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και τι προδιαγραφέ και τι αξίε μα, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντο. Θεωρώ ότι το σώμα θα πρέπει να συνενέσει το ταχύτερο δυνατόν για να περάσουμε στην εφαρμογή για να την εκμεταλλευτούμε όλοι το στομότερο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Τζιλ έχει το λόγο ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε, Κυρία Χάουταλα, συγχαρητήρια για την ε, έκθεσή σας. Επικροτώ τη συμφωνία αυτή με το Βιετνάμ που τώρα δεσμεύεται να εισάγει μόνο νόμιμη ξυλία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι είναι κορυφαία η θέση του Βιετνάμ στα προϊόντα ξυλίας. Ε, η αποδάσωση είναι δεύτερος, η δεύτερη σημαντικότερη αιτία για την ε, υπερθέρμανση του πλανήτη. Ε, είναι λοιπόν σημαντική συμφωνία αυτή και για τους στόχου του Παρισιού και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω ωστόσο δύο ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχά θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη να ασχοληθούμε με την περιφερειακή διάσταση της παράνομη υλοτομία. Θα ήθελα να γνωρίζω τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την παράνομη υλοτομία σε χώρες όπως είναι το Λάος και η Καμπότζη. Επίσης, ε, τι συμβαίνει όσον αφορά την Εθελοντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ε, με την Κίνα. Και τέλος, σε τι βαθμό ο κανονισμός έχει θυχθεί στις διαπραγματεύσεις ε, με την Ιαπωνία, που επίσης είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελεύθερους και δημοκρατικούς, ε, ο η κυρία να έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόληψη της αποψήλωσης των δασών είναι κομβική σημασία για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και αυτό πρέπει να το, να το βλέπουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική διαμορφώνοντας μια σφαιρική προσέγγιση τοπικά, περιφερειακά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη είναι ένα παράδειγμα στον τομέα αυτό, η Φιλανδία ιδίω. Είμαι ικανοποιημένη γιατί συμφωνήσαμε με αυτή την ε, εθελούσια συμφωνία με το Βιετνάμ. Είναι μια χώρα που έχει κάνει σημαντικά και γρήγορα βήματα για να προστατεύει τα δάση της και να είναι νόμιμα τα προϊόντα ξυλίας που εξάγονται στην Ευρώπη ε, που είναι ένας κλάδος εξαιρετικά χρήσιμος άλλωστε για τη χώρα. Χρειαζόμαστε τέτοιες συμφωνίες το σύντομο το δυνατό γιατί αυτό θα δώσει καλύτερη ευημερία για το Βιετνάμ και περισσότερες θέσεις εργασία και για τις δύο πλευρές. Γι' αυτό θα πρέπει, τόσο πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες που είναι σημαντικοί θα γίνονται σεβαστοί σε κάθε επίπεδο. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Σόλτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί εισηγητές, η ομάδα μου χαιρετίζει την συμφωνία αυτή. Αποτελεί ένα ενδιαφέρον υπόδειγμα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε οικονομικές προοπτικές για τον λαό, ταυτόχρονα με την προστασία της φύσης και του κλίματος για να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 στην Νοτιοανατολική Ασία. Το Βιετνάμ έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ε, λαθρολοτομίας στην πράξη ε, ειδικά από το Λάος και την Καμπότζη. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να προσφέρουμε έμπειρια και οικονομικά μέσα, γιατί τα προγράμματα αυτά ήδη μείωσαν το παράνομο εμπόριο κατά 20% αλλά υπολογίζεται ότι ούτως ή άλλως οι απώλειες από την παράνομη λετομία είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε θα πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο για να περάσουμε σε μια αηφόρο υλοτομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Φρουντσούλικα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να τονίσω το ότι το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας ε, στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και μια πολύ δυναμική χώρα στην περιοχή. Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια πολλών ανάλογων συμφωνιών με χώρες ε, στην Αφρική, με την Ινδονησία και βασίζεται στον κανονισμό περιξηλίας του ΟΗΕ. Ω μέλο τη επιτροπή ανάπτυξη ε, πρέπει να πω ότι στηρίζω αυτή την συμφωνία. Επίση, ε, πρέπει να δούμε και τι κοινότητε των αυτοχθόνων που συχνά βασίζονται στα δάση και είναι συχνά θύματα της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος. Πρέπει να διασφαλίσουμε η συμφωνία αυτή να συμπληρώνει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο για μεγάλης κλίμακας εκμετάλλευση των δασών. Πρέπει να αποτρέψουμε τη μαζική αποδάσωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φρουντζουλίτσα και περνάμε τώρα ε, στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και ξεκινάμε με τον κύριο Μαριά. Grazie, το βιετνάμ είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ξυλίας στον κόσμο και βεβαίως σημαντικός εμπορικός εταίρος της ευρωπαϊκής ένωσης. η εθελοντική αυτή συμφωνία πραγματικά εάν τηρηθεί και εφαρμοστεί σωστά θα μπορεί να συμβάλλει στην ε, αντιμετώπιση της λαθροϊλοτομίας. είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να σταματήσει η αποδάσωση να στηριχθούμε στις προσπάθειες οι οποίες ε, πραγματικά ενισχύουν ε, συνθήκες περιβαλλοντικές τέτοιες που διασφαλίζουν ε, την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής. βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα διότι γίνεται παράνομη εισαγωγή ξυλίας στο βιετνάμ από την καμπότζη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη διαφθορά η οποία υπάρχει στα τελωνεία στις τελωνειακές αρχές του βιετνάμ. εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί προφανώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή και ορθή εφαρμογή της συμφωνίας την οποία βλέπουμε. επομένως είναι θέμα τήρησης εκ μέρους του βιετνάμ των όρων και των προϋποθέσεων της εθελοντικής αυτής συμφωνίας. ευχαριστώ. Ο κ. Σόσνιερτς έχει το λόγο. Χαίρομαι για αυτό το ψήφισμα και εγώ και οι ψηφοφόροι μου στην Πολωνία χαίρονται που θα προστατευτούν τα δάση του Βιετνάμ. Η μισή από τους ψηφοφόρους μου είναι υπέρ ε, των ποσοστώσεων υπέρ της Καμπότζης και η μισή κατά. Υπάρχει μεγάλη συναισθηματική φόρτωση ε, και παρακολουθούν αυτή την ε, συζήτηση. Σας διαβεβαιώ ε, οι ψηφοφόροι μας. Και δεν ακούνε μόνο οι δικοί μου ψηφοφόροι, αλλά ακούνε και όλος ο κόσμος για το θέμα αυτό και ότι έχει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, σοφούς ανθρώπους που συζητάνε τέτοια θέματα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρω ότι κατεβάζω λιγάκι το επίπεδο. Πάντως, χαίρομαι που δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω. Ε, οι Πολωνοί ε, ψηφοφόροι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για το θέμα ε, του μελιού που συλλέγεται στην Παραγουάη. Ελπίζω να το συζητήσουμε στην επόμενη σύνοδο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στην Επίτροπο στον Επίτροπο Άντσιπ, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ που επιστήσατε την προσοχή της Κομισιόν στα όσα σας απασχολούν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και την κατάσταση που επικρατεί στο Βιετνάμ. Ακούστε και ένα ερώτημα για μια, για μια περιφερειακή πρωτοβουλία. Υπάρχουν ε, εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με το Λάος, διάλογος με την Καμπότζη, διμερή συνεργασία με την Κίνα, όπου η νομιμότητα των προϊόντων ξυλίας είναι προτεραιότητα. Επίσης υπάρχει διάλογος και με την Ιαπωνία. Τα μηνύματα που ακούστηκαν σήμερα είναι ξεκάθαρα και βροντερά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους Βιετναμέζους εταίρους, ούτως ώστε να θέσουμε ε, ένα φιλόδοξο πλαίσιο, ούτως ώστε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Σας διαβεβαιώ ότι η Κομισιόν δεσμεύεται και είναι έτοιμη να κάνει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, η Κομισιόν έχει το βλέμμα στραμμένο προς τα εμπρός. Να βασιστούμε στη θετική εμπειρία που έχουμε με τις εθελοντικές ε, συμφωνίες εταιρική ε, σχέσης και, και την εφαρμογή της δασικής ε, νομοθεσίας διακυβέρνηση και εμπόριο και αυτό απέναντι στο Βιετνάμ. Εδώ έχουμε επενδυτικές συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες με το Βιετνάμ και συμφωνίες εθελοντικής, εθελοντικές συμφωνίες εταιρική σχέσης πάντα με το Βιετνάμ. Θα ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο στην εφαρμογή της ε, Θελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με το Βιετνάμ, της VPA, και πώς τα θέματα που θέτει το ψήφισμα αντιμετωπίζονται από τους Βιετναμέζους. Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω ότι με το να, ότι με το να δώσετε τη σύμφωνη γνώμη σας δεν υποστηρίζετε απλώς την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέσης, επαναδιατρανώνετε τη σημασία του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ε, δασικής νομοθεσίας που από το 2003 έχει διαμορφώσει τον αγώνα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παράνομης υλοτόμησης και η οποία ευθύνεται για την ε, αποδάσωση. Βλέπουμε ότι αυτό το σχέδιο δράσης είναι βασικό παράδειγμα εμπορικής πολιτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής που άλλο υποστηρίζονται. Χρειαζόμαστε τέτοια συνοχή στην πολιτική μας για να αντιμετωπίσουμε τις ευρύτερες προκλήσεις της αποδάσωσης. Και θα μας καθοδηγήσει καθώς αναπτύσσουμε περαιτέρω τις πολιτικές μας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Και τώρα, η εισηγήτρια έχει το λόγο, η Αντιπρόεδρος κυρία Χάουτολα. Χάιντε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ γιατί κάναμε εξαιρετική δουλειά μαζί. Χαίρομαι που βλέπω ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο φαίνεται ότι θα υποστηρίξει αυτή την εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Βιετνάμ. Είναι κατά πάσα πιθανότητα το πιο αποτελεσματικό εμπορικό εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τι αρνητικέ εξελίξει που δεν θα επέτρεπαν την πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και όπω είπαν και οι συνάδελφοι και ο, Επίτρο, ο κύριος Επίτροπος να έχουμε κατά νου την περιφερειακή διάσταση. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι ένα από τα τρία πιο σημαντικά σημεία αποψήλωση των δασών στον κόσμο. Το άλλο είναι το Κονγκό και η ε, Λατινική Αμερική. Σε όλου αυτού του τομεί έχουμε εθελοντικέ ε, συμφωνίε εταιρική σχέση οι οποίε βρίσκονται εν εξελίξη. Ε, αναμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει ιδιαίτερα σοβαρά τις αποκαλύψεις για οργανωμένο έγκλημα και για την ε, λαθροϊλοτόμηση στην Νοτιοανατολική Ασία όπως προσφάτως έχουν καταδειχθεί από φορείς προστασίας του περιβάλλοντος στη Μιανμάρ. Και επίσης τώρα έχουμε και αξιόπιστους ισχυρισμούς ότι το Βιετνάμ άρχισε να αντικαθιστά τις εισαγωγές από Καμπότζη με εισαγωγές από την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ε, λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό για παράνομη υλοτόμηση. Χαίρομαι που ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα διάφορα βήματα στην υλοποίηση αυτή τη εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση και πιστεύω ότι οι δύο επιτροπέ που ασχολήθηκαν περισσότερο με το θέμα, Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και Επιτροπή Ανάπτυξη, θα συνεχίσουν να, να έχουν βαρύνοντα λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να, να επικυρώσουμε τη συμφωνία και το μη νομοθετικό ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κοινή συζήτηση έκλεισε. Η ψηφορία θα γίνει αύριο. Προχωρούμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι η έκθεση το κύριο Σέπφλιν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαμασού, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Σέπφλιν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τις επιθυμίες ολόκληρου του Κοινοβουλίου για τον κύριο Σέπφλιν, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο για μια σοβαρή ασθένεια, ε, να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών έχει σαν σκοπό να δείσει στου πολίτε αν είναι επαρκή και έρχονται από το 1 τέταρτο ε, ευρωπαϊκών χωρών ένα δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας ανάλογο με αυτό που έχει το Κοινοβούλιο μέσω των ψηφισμάτων που ψηφίζουμε κάθε μήνα και το Συμβούλιο Υπουργών. Τη δυνατότητα δηλαδή να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την καλέσουν να νομοθετήσει σε ένα νέο τομέα ή να πάψει να νομοθετεί ή να τροποποιήσει μια παλιά νομοθεσία. Ο πρώτο κανονισμό, ο οποίος υιοθετήσαμε πριν από λίγα χρόνια για και αποτελούσε τη νομική βάση του συστήματος ήταν αρκετά απογοητευτικό γιατί μόνο τέσσερι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών κατέληξαν και έφτασαν στην τελική φάση της διαδικασίας. Γι' αυτό ακριβώ ε, ε, ε και ο Επίτροπος Τίμερμας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων συνεργάστηκαν για να ετοιμάσουμε μια νέα πρόταση ε, που οδήγησε σε μια συμφωνία σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου, η οποία εγκρίθηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων με 10 ψήφους υπέρ, καμία ψηφοκατά και τρει αποχές μόνο. Ο νέος κύκλος ζωής, ο οποίος εισάγεται τώρα σε αυτόν τον ε, κανονισμό για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών είναι πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και επιτρέπει μια πιο απλή διαδικασία, πιο προσπελάσιμη, λιγότερο δαπανηρή, πιο ε, διαφανή, με την εισαγωγή της δυνατότητα μιας μερικής καταγραφής της πρωτοβουλίας πολιτών με αρχικό σκοπό ε, όταν εκφεύγει των πεδίων της συνθήκης και με την υποχρέωση της Κομισιόν να παρουσιάσει τα συμπεράσματα ε, σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, έξι μήνες, και οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για την υποχρέωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οργανώνει μία συζήτηση πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφανθεί ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και και να έχει την ευθύνη το Κοινοβούλιο να υιοθετεί μία πρόταση ψηφίσματος γιατί θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο, εμείς δηλαδή, ε, τροποποίησε τον εσωτερικό του κανονισμό ούτω ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η δυνατότητα. Η ε, αναθεώρηση του κανονισμού εξασφαλίζει πιο διαφανή χρηματοδότηση, έχει προβλέπει σημεία επαφής, ε, αρχείο ε, online, ούτω ώστε να μπορούμε έτσι να διαχειριζόμαστε online όλη τη διαδικασία και προβλέπεται μέχρι το 2020 η Κομισιόν θα εφαρμόσει ένα σύστημα κεντρικό για την ε, συλλογή online των δηλώσεων ε, στήριξης. Αυτό το σύστημα υπάρχει ήδη, απλώς είναι απερχαιωμένο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να σταματήσει να... Θα, να, θα ολοκληρωθεί μάλλον μέχρι το τέλος του χρόνου και το ζητούσαν οι ΜΚΟ. Άλλες ΜΚΟ και άλλα άτομα τελευταία στιγμή ανησύχησαν για τη διαδικασία αλλά δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε το περιεχόμενο αυτού του τριμερούς διαλόγου και επομένως η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, συστήνει εδώ στην Ολομέλεια να επιβεβαιώσουν τη θαυμάσια συμφωνία που επετεύχθη σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λεμασούχ. Και εγώ θέλω να ευχηθώ εκ μέρου μου ε, καλή ανάρρωση στον κύριο Σέπφλιν. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά από την Επιτροπή και εγώ όπως και όλοι ευχόμεθα να επανέλθει στο Κοινοβούλιο υγιής και δυνατός. Ο κύριος Σάνσιπ έχει το λόγο τώρα, επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η συζήτηση αυτή κλείνει τη διαδικασία επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στο πλαίσιο της Επιτροπής Juncker. Επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρώπης να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει κάποια πρόταση για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Από τότε που άρχισε να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα πριν από περίπου 7 χρόνια, πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτε έχουν υπογράψει πρωτοβουλίες πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αποτελούν σημαντικό μέσο για την προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει στους πολίτες να ξεκινούν ευρωπαϊκές συζητήσεις και βοηθούν να προωθούν θέματα στην ημερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δύο ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών. Η οδηγία για το πόσιμο είδωρ και η οδηγία για την αξιολόγηση κινδύνων στην αλυσίδα τροφίμων, όπου τα θεσμικά όργανα έχουν καταλήξει σε ε, πολιτική συμφωνία. Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα αναθεωρημένο κανονισμό για την πρωτοβουλία πολιτών, ούτω ώστε να αποκτήσει το πλήρες δυναμικό της. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθούμε τους πολίτες και να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν το μέσο αυτό χωρίς να υπάρχουν εμπόδια στην πορεία αυτή. Το κείμενο στο οποίο έχει συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα δώσει τη δυνατότητα στις πρωτοβουλίες πολιτών να είναι περισσότερο προσιτές και περισσότερο φιλικές προς το χρήστη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για τους οργανωτές ε, πρωτοβουλειών να αποκτήσουν, να αποκτήσουν υποστήριξη μέσω ε, online πλατφόρμα στα κράτη-μέλη. Θα βοηθήσει τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας να έχουν καλύτερη διαδικασία καταχώρησης και θα τους δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερη ευελιξία στη χρονική στιγμή έναρξη τη εκστρατεία τους. Η Επιτροπή θα δίνει στους οργανωτές ε, μια δωρεάν εξυπηρέτηση για την ε, online συλλογή υπογραφών. Θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία τα οποία παρέχουν οι πολίτες ε, με ασφάλεια. Όλοι θα μπορούν να υπογράψουν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Επίσης θα υπάρχει περισσότερος χρόνος ε, για ευαισθητοποίηση, για συμμετοχή και για συζητήσεις πριν από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή ε, θεωρεί κρίμα το ότι κάποιες από τις, ε, κάποιοι, κάποιοι από τους στόχους που θέλαμε να επιτύχουμε στη μεταρρύθμιση αυτή δεν κατορθώσαμε τελικά να τους επιτύχουμε. Τελικά δεν μπορέσαμε να μειώσουμε ε, την ηλικία συμμετοχής στα 16 από τα 18 χρόνια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να μειώσει την ηλικία για τους δικούς της πολίτες, αν το επιθυμεί το κράτος μέλος αυτό. Ελπίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη θα μειώσουν την ηλικία συμμετοχής, διότι η φωνή της καινούριας γενιάς πρέπει να ακούγεται. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός επιφέρει ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης ε, στοιχείων, το οποίο παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δωρεάν. Θέλουμε να συνεχίσουν να έχουν την επιλογή οι οργανωτές να χρησιμοποιούν το δικό του σύστημα, αν το προτιμούν έναντι του κεντρικού συστήματος. Και συμβιβαστικά, αυτή η δυνατότητα ε, θα εκλείψει σταδιακά μέχρι το τέλος του 2022. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παρέχει ένα σύστημα υψηλής ποιότητας το οποίο θα αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους. Πιστεύω ότι έχουμε ε, επιτύχει το στόχο μας, δηλαδή η πρωτοβουλία πολιτών να γίνει περισσότερο προσιτή, λιγότερο δίσκαμπτη και πιο εύκολη στη χρήση της. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως ε, τον εισηγητή, τον κύριο Σέφλιν, για την δέσμευση την οποία επέδειξε για την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και για τη συμβολή του ώστε να επιτύχουμε αυτό το πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, ο κύριο Τζαμπάσκι. Η κυρία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως είναι εισηγητής της γνωμοδότησης αυτής για τη δική μας Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάπφλιν και όλους τους συνεισηγητές για την συνεργασία τους. Το αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε φτάσει είναι ισορροπημένο. Δίνει την ε, ευκαιρία στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτό το σύστημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό δημοκρατικό εργαλείο η πρωτοβουλία αυτή, διότι επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση συμμετοχή στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Οι αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα έπρεπε να γίνουν, γιατί ήταν πολύ περίπλοκο και δύσκολο να χρησιμοποιηθεί είχαμε παρατηρήσει σειρά εμποδίων τα οποία έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε. Διευκολύνεται η συλλογή υπογραφών και προστατεύονται καλύτερα τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα η πρωτοβουλία να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Στην Επιτροπή Αναφορών, ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Σέφλιν, για τη δουλειά που έχει κάνει. Να πω ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με τον Επίτροπο Τίμερμανς και με τους εκπροσώπους της Αυστριακής Προεδρίας. Τα αποτελέσματα είναι καλά. Θελήσαμε να μεταρρυθμίσουμε αυτή την πρωτοβουλία για να δώσουμε ένα χρήσιμο εργαλείο στους Ευρωπαίους πολίτες. και από πλευράς της Επιτροπής Αναφορών είναι σημαντικό το γεγονός ότι είναι δημόσια η ακρόαση εντός του Κοινοβουλίου στην οποία παρουσιάζουν λεπτομερώς οι φορείς τις πρωτοβουλίες τους έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό θέλαμε. Δεν καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να έχουμε την ύψιστη δυνατή εκπροσώπηση από πλευρά δύο αυτών ε, θεσμικών οργάνων. Ε, ήταν σα η διατύπωση. Ο Επίτροπος Τίμερμαν, αλλά και η Αυστριακή Προεδρία είπαν θα το δούμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί θα θέλαμε να γραφτεί στο κείμενο ότι ο πρόεδρο τη Επιτροπή ή ε, ε, ο, ο πρόεδρος της προεδρία Προεδρίας του Συμβουλίου θα παρίστανται για να έχουμε την ύψη στη δυνατή εκπροσώπηση. Ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τώρα, ο κύριος Σάκη. Πάλι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς οι Ευρωβουλευτές ανέκαθεν Λέγαμε ότι πρέπει να απλουστευτεί και να βελτιωθεί αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους πολίτες. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις προτάσεις των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος να γίνει μια πραγματική ένωση πολιτών. Να είναι πιο απρόσκοπτη διαδικασία με σαφέστερους κανόνες. Και από ό,τι φαίνεται αλλάζει η κατάσταση σήμερα. Με την πάροδο λίγων μηνών το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε δίκιο στους Ευρωπαίους πολίτες και καταδίκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλούμε για τις ε, μειονότητες και τα δικαιώματά τους. Ένα άλλο θέμα είναι η πολιτική συνοχή για την ισότητα μεταξύ των περιφερειών και για τη βιωσιμότητα των... της εκάστοτε περιφερειακής κουλτούρας. Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες είχαν απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δικαστήριο μας δικαίωσε. Γνωρίζουμε τώρα ότι αυτό ήταν λάθος. Η συλλογή υπογραφών για το Safe Pack μας έδειξε λοιπόν ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειάστηκε να συλλέξουμε πολύ περισσότερες υπογραφές από ό,τι χρειαζόταν και με βάση την απόφαση του δικαστηρίου από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει και δεύτερη συλλογή υπογραφών. Φαίνεται λοιπόν ότι το ζήτημα των μειονοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με, ε, με ιδιαίτερη έμφαση και αυτό είναι καλό. Ευχαριστώ. Και τώρα από τους σοσιαλιστές, Κάουφμαν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υπάρχει εδώ και 7 χρόνια περίπου. Από την ένταξη ισχύω του κανονισμού, πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτε έχουν δώσει την υπογραφή του για να υποστηρίξουν κάποια πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό δείχνει ότι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ε, ε, ενστερνιστεί αυτό το μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας. Η άλλη πλευρά του νομίσματος βέβαια είναι ότι ε, πολύ λίγες πρωτοβουλίες κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές σε πάνω από 7 κράτη-μέλη. Από την πράξη λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ε, ήταν τα θέματα που τους απασχολούν σε πρώτο επίπεδο περισσότερο. Είχαμε ε, θέματα που έχουν σχέση με διοικητικά ζητήματα. Είναι καλό λοιπόν το ότι έχουμε τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια. Καταρχήν, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, να υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία πολιτών. Δεύτερον, ε, σημεία επαφής ε, θα οργανώνονται στα κράτη-μέλη και θα έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται αυτά τα σημεία οι οργανωτές πρωτοβουλειών. Η Επιτροπή θα μπορεί να ελέγχει τις ε, πρωτοβουλίες πριν τις ε, ε, εγκρίνει πλήρως. Και τέταρτον, για την προετοιμασία της εκστρατεία, θα έχουν βοήθεια και θα μπορούν να αποφασίζουν για το χρονικό σημείο έναρξης της εκστρατεία τους. Και πέμπτον, θα μπορεί να διοργανώνεται και μια δημόσια ακρόαση ώστε να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών και έχει τροποποιηθεί αντιστοίχω και ο κανονισμό για να το ε, επιτρέπει. Θα είναι λοιπόν πιο φιλικέ προ το χρήση οι πρωτοβουλίε πολιτών. Η πολιτική μα ομάδα έχει συζητήσει πάρα πολύ ε, το θέμα τη πρωτοβουλία των πολιτών, ούτω ώστε να αποκτήσει πιο νεανικό χαρακτήρα, μειώνοντα ε, την ελάχιστη ηλικία. Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί, ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, θέλουν να υπερασπίσουν την άποψή του για θέματα που αφορούν την αλλαγή του κλίματο ή το ελεύθερο ίντερνετ. Θέλουν να συμμετέχουν και πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν επέτρεψε την μείωση της ελάχιστης ηλικίας. Έχει γίνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όμως, διότι τώρα τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνα τους για την μείωση της ηλικίας από τα 18 σε μικρότερη ηλικία. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια ζωντανή συζήτηση και θα μπορέσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό το ότι οι νέοι μπορούν να υποστηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τη συμμετοχή των νέων. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Και τώρα, από το ECR, ο κύριος Μαριάς. Νότι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία πολιτών είναι μια συγκεκριμένη έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενισχύεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι συμμετείχαν μέχρι στιγμής 9 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες Πρωτοβουλίε πολιτών δείχνει την μαζική συμμετοχή και το γεγονός ότι ήδη ξεκινά νομοθετική πρωτοβουλία για το πόσιμο είδωρ δείχνει την επιτυχία της προσπάθειας. όμως θα πρέπει η όλη διαδικασία να είναι πιο απλουστευμένη να μην έχει τον κυρίαρχο ρόλο η επιτροπή η οποία είναι αυτή την οποία καλούν οι πρωτοβουλίε να νομοθετήσει αλλά η ίδια ελέγχει κατά πόσο οι πρωτοβουλιε είναι ορθε ω εκ τούτου η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική το συζητήσαμε στην επιτροπή αναφορών και φυσικά το δικαίωμα των διοργανωτών να έχουν μια δημόσια ακρόαση και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο νομίζω ότι διευρύνει τη δημοκρατική πλευρά της λειτουργίας. στηρίζω την προσπάθεια να έχουμε τη μέγιστη συμμετοχή των νέων 16 ετών νέοι να μπορούν να συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια. το γεγονό ότι δεν το επιτρέπει το συμβούλιο είναι αρνητικό όμως τα ίδια τα κράτη μπορούν να δώσουν αυτή την ευκαιρία και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει την ευκαιρία αυτή. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υπάρχει ε, μία μπλε κάρτα των Σοφάουζερ. Τη δέχεστε? Παρακαλώ. Μίλησαν για μια πρωτοβουλία των πολιτών με 2 εκατομμύρια άτομα για τον σεβασμό ε, της ανθρώπινης ζωής από την ε, σύλληψη μέχρι το θάνατο. Την υποστηρίζω και εγώ. Αλλά δεν αναγνωρίστηκε και δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο, γιατί υποτίθεται ότι αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του Κοινοβουλίου, υποτίθεται. Θα ήθελα να μου πείτε τι ξέρετε και τι άποψη έχετε. Ευχαριστώ. Please. κοιτάξτε θα ήθελα να πω το εξής ότι η διαδικασία προβλέπει να υπάρχει και η θέση της κομισιόν και η θέση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. στο βαθμό όμως που υπάρχει διαφωνία θεωρώ ότι θα μπορούσαν οι αρμόδιοι να προσφύγουν στο δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης όπως έγινε και με τις άλλες πρωτοβουλίες και να κριθεί από εκεί και πέρα αν αυτό ήταν νόμιμο ή ήταν παράνομο. σε τελική ανάλυση η εφαρμογή της νομιμότητας διασφαλίζεται από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι αρμόδιοι. ευχαριστώ από τους φιλελεύθερους η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Επίτροπε. Η βελτίωση και η διευκόλυνση τη άσκηση τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια συνεισφορά στη δημοκρατία και είναι μια απαραίτητη γυτνίαση των πολιτών προ τι ευρωπαϊκέ υποθέσει. Είναι καλό νέο το να διαπιστώνουμε ότι πολλέ από τι βελτιώσει που έχουν εισαχθεί σε αυτή την έκθεση για να γίνει πιο χρήσιμη, πιο απλή η άσκηση αυτού του δικαιώματο ε, προέρχονται από του ίδιου του πολίτε. Όλα αυτά τα λέω γιατί έσα από πάρα πολύ κοντά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από μία από αυτέ τι πρωτοβουλίε, το Minority Safe Pack, ε, που κατάφεραν να το υπογράψουν ε, ο ελάχιστο αριθμό πολιτών σε 12 κράτη-μέλη, ώστε να παρουσιαστεί και να ληφθεί υπόψη. Έζησα όλε αυτέ τι δυσκολίε από πολύ κοντά. Ελπίζω αυτέ οι βελτιώσει αυξάνουν τον αριθμό των πρωτοβουλειών που υποβάλλονται και τον αριθμό των πολιτών που εμπλέκονται ε, και είναι μια καλή ιδέα αυτές οι πρωτοβουλίες να εξετάζονται σε δημόσια ακροάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συζητούνται στην Ολομέλεια και να οδηγούν σε πρόταση ψηφίσματος. Είναι θετικό και το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προθεσμίες. Επίσης, βελτιώνουμε τις πλατφόρμες και τις τεχνικές ε, προϋποθέσεις και τεχνικά μέσα που έχουν ε, αυτοί που τις προτείνουν. Επίσης, το γλωσσικό καθεστώς θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ε, ε, πολιτιστική ποικιλομορφία της Ένωσης. Της ε, Ένωσης. όσοι μιλούν μειωτικέ γλώσσε, διεκδικούν το Minority Safety Safe Pack. πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, είναι θέματα ευαισθησία και γυπνίαση. νομίζω ότι θα πρέπει και το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για να προωθηθεί αυτό το, έγγραφο, αυτό το εργαλείο συμμετοχής ε, των πολιτών. Σας παρακαλώ, από εδώ και πέρα, να μην ξεπερνάμε τα δύο λεπτά. Από τους πράσινους, ο κύριος Στερικάβρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δουλεύουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια για αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν είχε συμφωνήσει η ομάδα μου για την πρώτη εκδοχή, γιατί δεν ήταν αρκετά ισχυρή. Τώρα καταλήξαμε σε ένα τελικό κείμενο που έχει βελτιώσει κατά πολύ το παλαιό κείμενο, ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω τα θετικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας, παρότι επαναλαμβάνω κάτι που ήδη είπαν και οι συνάδελφοί μου. Τώρα οι οργανωτές έχουν τη δυνατότητα να καταγράφονται ως νομικές οντότητες. Δεύτερον, η μετάφραση του παρατήματος περιλαμβάνεται με ε, λογικό περιορισμό του αριθμού των χαρακτήρων. Τρίτον, οι οργανωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την ε, χρονική ημερομηνία που τους εξυπηρετεί. Ε, τέταρτον, μπορεί να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με τι διευθύνσει των πολιτών. Ε, πέμπτον, όλοι οι πολίτε θα μπορούν να υπογράφουν πρωτοβουλία πολιτών ανεξάρτητα από το που κατοικούν. Ε, έβδομο σημείο. Σημαντικό είναι η παρακολούθηση. Μία παρακολούθηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ακρόαση και μία μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά λοιπόν παρουσία και αυτό το δικαίωμα παρέμβαση και αυτό αποτελεί πολύ θετικό σημείο. Να αναφέρω και ένα αρνητικό σημείο όμως. Και εδώ διαφωνώ κάπως με αυτό που είπε ο κύριος Λαμασούρ σχετικά για το ατομικό σύστημα συγκέντρωση υπογραφών, το οποίο θα, θα επιτρέπεται μέχρι το τέλος του 2022 και όχι αργότερα, ε, είναι κάτι ένα του οποίου ε, διαφώνησαν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, μετεπιτάσεως μάλιστα το ατομικό σύστημα θα έπρεπε να συνεχίζεται. Τελικά όμως, αν εξετάσουμε συνολικά το θέμα, αν δούμε τα υπέρ και τα κατά, θα πρέπει να δεχθούμε ότι η συνολική πρόταση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Και γι' αυτό θα προτείνω στην ομάδα μου να ψηφίσει υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή είναι ήδη περασμένη η ώρα και έχουμε αρκετούς ομιλητές και έχουμε και άλλα θέματα. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο που σας δίδεται. Για την ΚΟΑ, κυρία Σπινέλη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Για τέσσερα χρόνια ασχοληθήκαμε με ένα εργαλείο που προβλέπουν οι συνθήκες, αλλά ήταν θνησιγενές, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους πολίτες. Προσπαθήσαμε να, την, της δώσουμε νέα πνοή για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος. Ε, τεράστια κρίση αντιμετωπίζει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας. Ε, οι επιθέσεις που δέχονται τα, η ΜΚΟ, τα συνδικάτα. Ε, και αυτό τι είναι, το αίτημα για μια άμεση δημοκρατία. Μια, ένα αίτημα το οποίο ε, γίνεται επικίνδυνο όταν δεν το ακούμε, όπως, έδειξαν, όπως μας έδειξε το Brexit. Χάσαμε την ευκαιρία εν μέρη και οι πολίτες δείχνουν την απογοήτευσή τους. Η πρωτοβουλία αυτή τεχνικά έχει βελτιωθεί μόνο. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι η πρωτοβουλία αυτή στέθηκε με επιτυχία. Αλλά το η δυνατότητα για να δοθεί νομοθετική συνέχεια είναι μονοπόλιο στα χέρια της Κομισιόν, ακόμα και η συλλογή των υπογραφών. Είναι, ε, μία, ε, είναι η νιωστή, νιωστή, ο νιωστός κόλαφο που δίνεται ε, στις ΜΚΟ. Είναι σαν να έχουμε φτιάξει ένα smartphone ε, πιο τέλειο, αλλά να έχουμε μπλοκάρει τις ε, κλήσεις. Είναι user-friendly, αλλά όχι citizen-friendly. Δεν έχει πεθάνει αυτή η πρωτοβουλία, αλλά είναι σε κόμμα. Κλείνουμε την πόρτα στη συμμετοχή των πολιτών στην πραγματικότητα, τη συγκεκριμένη στιγμή όπου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα Στι ευρωπαϊκέ κοινότητε, στι Ευρωπαϊκέ χώρε. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, που σα κόβω. Θέλω να σεβαστούμε το χρόνο. Σά παρακαλώ. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό από εδώ και πέρα. Πρέπει να είμαστε ευγενεί και προ του συναδέλφου. Αυτού που θα ακολουθήσουν τι δικέ μα παρεμβάσει. Η κυρία Εύη είναι η επόμενη από το EFTD για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την τροποποίηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, και κατά την άποψή μου έχουμε χάσει μια ευκαιρία για να φέρουμε πιο κοντά τον ε, πολίτη στην ε, Ευρώπη. Υποτίθεται ότι φτιάξαμε ένα εργαλείο για να καλύψουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Ο συμβασμό ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι αποδυναμώνει όμως αυτό το εργαλείο. Ε, είμαστε στα όρια που επιβάλλουν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει υποχρέωση για την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το θέμα που αποτελεί την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Ε, αν η συμφωνία επιβεβαιωθεί, όχι μόνο το αίτημα που προέρχεται απευθεία από ένα εκατομμύριο πολίτε θα μπορούσε να αγνοηθεί ή να παρακαμφθεί, αλλά θα μπορούσε να ακυρωθεί το σύστημα συλλογή υπογραφών ε, που θα το διαχειρίζονται οι διοργανωτές ε, που μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να, και, για να συλλεγχθούν οι υπογραφές και για να διευκολυνθεί η συζήτηση για το θέμα της πρωτοβουλίας. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα εργαλείο πολύ πιο δυνατό, ε, με σεβασμό των ε, συνθήκων, ε, με, αν είχαμε τρεις ακροάσεις. Μία κατά τη διάρκεια των υπογραφών, όταν φτάσουμε στο ένα εκατομμύριο υπογραφές και μία με, μετά το, με το follow-up. Και όχι με απλή αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, αυτό για να ακούσουμε περισσότερο τους πολίτες. Αλλά αυτό που πριτάνεσε τελικά ήταν η έπαρση αυτών που θεωρούν ότι όλα αποφασίζονται στα διάφορα γραφεία των Βρυξελών. Η Κομισιόν είναι, παίζει από μόνη της, παίζει ενού Δεν δίνει καμία λογοδοσία απέναντι στους πολίτες, κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα παίζουμε ένα παιχνίδι ε, παγιδευμένο από την αρχή ως το τέλος. Τα χαρτιά είναι παγιδευμένα. Αύριο θα ψηφίσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό κείμενο που όμως ε, έμεινε γράμμα κενό περιεχομένο. Ευχαριστώ κύριο Σκοέγιο. 1,5 λεπτό. Ε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς δεν δεχόμαστε μια Ευρώπη που δεν θα είναι κοντά στους πολίτες. Είναι σημαντικοί οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της συνθήκης Λισαβόνα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, που ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, που πρόθεσε τη συμμετοχή των πολιτών και ενέπλεξε περιττέρω τους ε, εκλογεί. Εκατομμύρια Ευρωπαίων από πολλές χώρες ε, συμμετείχαν ε, και πολλοί Πορτογάλοι συμμετείχαν. Αλλά δεν αρκεί αυτό για να ενισχύσει την, ε, την Ευρώπη των πολιτών, για να καταπολεμήσει την απάθεια και την αποχή από τις εκλογές, για να καταπολεμήσουμε τους δημαγωγούς. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την πρωτοβουλία, να την απλουστεύσουμε ακόμα περισσότερο, να την κάνουμε πιο προσπελάσιμη και να λάβουμε υπόψη μας την ανησυχία που υπάρχει για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θέλω να μειωθεί ο αριθμός των κρατών για την συμμετοχή. Θέλουμε περισσότεροι πολίτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν, ούτως ώστε όλοι να συμμετάσχουμε ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχουμε στις πρωτοβουλίες. Γιατί περισσότερη δημοκρατία σημαίνει καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι η συμφωνία που υποβάλλεται προς ψήφιση είναι ενδιαφέρουσα γιατί βελτιώνει σημαντικά το μηχανισμό πρωτοβουλίας από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών. Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσουν αυτούς που αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει πλέον ένα επίσημο σύστημα συγκέντρωσης ε, διαδικτυακών υπογραφών. Δίνεται περισσότερος χρόνος για τη συλλογή των υπογραφών. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη μπορούν να τροποποιήσουν την νομοθεσία τους έτσι ώστε όσοι είναι από 16 και πάνω να μπορούν και να ψηφίσουν και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Και θέλω να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διοργανώσει συζήτηση για τέτοιου είδου πρωτοβουλίας. Η βραχία ζωή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στην Ευρώπη απαιτεί μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις που εθελήθηκαν τώρα είναι καλές και μάλιστα πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες πρωτοβουλίες και μεγαλύτερη ε, συμμετοχή των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ για ένα μισή λεπτό, Βελέσσα. Από το 2012, πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει πρωτοβουλίες πολιστών δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως ε, το δυναμικό αυτού του μέσου. Η επικαιροποίηση της, της πρωτοβουλίας πολιτών θα μπορέσει να υποφεληθεί και από ηλεκτρονικά μέσα, από την online συγκέντρωση υπογραφών και από την σχετική πλατφόρμα. Και όλα τα στοιχεία θα μπορούν να είναι προσιτά και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή θα μπορεί να καταχωρεί εν μέρη την πρωτοβουλία σε θέματα όπου η Επιτροπή μόνο έχει δυνατότητα πρότασης πρωτοβουλειών. Και επί έξι μήνες μετά την καταχώρηση μπορούν οι οργανωτές να αποφασίζουν πότε θα αρχίσουν την εκστρατεία τους. Μεγαλύτερη ευελιξία που θα είναι προς όφελος των μικρότερων ομάδων διοργανωτών. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Τα πρότυπα θα είναι υψηλότερα και θα είναι και πιο φιλικό προς το χρήστη το σύστημα αυτό. Προσβλέπουμε λοιπόν ε, στην ε, ανάπτυξη αυτού του μέσου που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε περνάμε και στη διαδικασία Catch the Eye. Αντιπρόεδρος κ. Καστάλιντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το... Λέγαμε πολλά και γεννήθηκε και, και δημιουργήθηκε ένα τίποτα στην πραγματικότητα. Ακόμα μία φορά το κείμενο του τριλόγου δεν είναι στο ύψος των ελπίδων. Δεν είναι αποτελεσματικό. Η, κανονικά για να γίνει η σωστή πρωτοβουλία πολιτών θα έπρεπε να, τροποποιηθεί η, να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Γιατί είναι παράλογος ο λόγος της, ο ρόλος της Κομισιόν και υπερβολικός. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά παρόλα αυτά και χωρί συνθήκε. Θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε στι οργανώσει κοινωνία των πολιτών. Αλλά όχι. Το κείμενο, αυτό που ψηφίσαμε, μα πάει προ τα πίσω. Δίνει μονοπόλιο στην Κομισιόν. Μονοπόλιο στη χρήση και στη διαχείριση τη πλατφόρμα τη κεντρική αυτή, ε, αντί για τους διοργανωτές, αντί για εκείνους ε, που μέχρι τώρα διαχειριζόταν μεμονωμένα τις ε, πρωτοβουλίες. Ε, Δώσετε μεγαλύτερη πρωτοβουλία στους Ευρωπαίους πολίτες, δώστε μεγαλύτερη πρωτοβουλία στου οργανώσει ε, των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Καστάντο είχε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν τα χρησιμοποίησε όλα. Η κυρία Ward έχει ένα λεπτό. Uh, I welcome. Καλωσορίζω την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και το τρόπο με τον οποίο την αξιολογούμε. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να εμπλέκονται σε συμμετοχικές διαδικασίες. Για να μπορούν να το κάνουν όμως πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι και να καταλαβαίνουν τις ευρωπαϊκές αξίες, τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που του αναλογεί για να φτιάξουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου του 2016 πολλοί δεν καταλάβαιναν για το τι ψήφιζαν στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ και θεωρούσαν ότι δεν είχαν τη δύναμη να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες λοιπόν πρέπει να είναι πιο προσβάσιμες για όλους. Και χαίρομαι διότι θα υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν και νέοι 16 ετών και χαίρομαι διότι θα είναι βελτιωμένη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα έχει τονιστεί το πόσο η φτώχεια λειτουργεί ως τροχοπέδι ε, και δεν μπορεί κανείς να ασκήσει τα δικαιώματά του ως πολίτες. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη για να χτίσουμε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Διακόπτη ο Πρόεδρος, παρακαλώ. Κυρία Γουόρτ, συγγνώμη, αλλά ε, ε, δεν έχετε άλλο χρόνο. Κυρία Κούνεβα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να έχουμε τόσες διαφωνίες. Συγγνώμη, είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να έχουμε τόσες διαφωνίες και τόσες μετοντεύσεις από ορισμένες πολιτικές ομάδες. Πρόκειται για ένα εργαλείο άμεσης δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα μας φέρει πιο κοντά στους πολίτες για να ακούσουμε τις φωνές τους και είναι χρέος μας να απαντήσουμε με πράξεις. 80 μέρες πριν τις εκλογές είμαστε και βάζουμε τόσα εμπόδια στους πολίτες. θέλουν να μας προτείνουν να δημιουργήσουμε νομοθεσία για τα προβλήματά τους. μα τι πιο καλά από αυτό. αλλιώς γιατί να μας εμπιστευτούν γιατί να μας ψηφίσουν όταν εμείς δεν τους δίνουμε σημασία. αδύνατο να ψηφίσουμε το κείμενο ως έχει. δυστυχώς οι λίγες προοδευτικές δυνάμεις δεν αρκούν για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. να είστε σίγουροι κάποιοι από εμά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ προσωπικά. Κύριε Φλάνγκαν, ένα λεπτό. Τελευταίο ομιλητή στο ΚΑΤΣΔΙ. Ευχαριστώ πολύ. 67 ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε πολιτών έχουν ξεκινήσει. Μόνο τέσσερι πλήρωσαν τα κριτήρια, δηλαδή το 1 εκατομμύριο υπογραφέ. Μόνο δύο κατέληξαν σε νομοθετικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νερό και ε, ε, για την ε, αλυσίδα διατροφή και του κινδύνου. Στην περίπτωση ορισμένων ε, ετοιμάτων η Επιτροπή αρνήθηκε γιατί ήταν αντίθετη η πρωτοβουλία των πολιτών ε, σε σχέση με τα σχέδια της Επιτροπής. Δηλαδή η Επιτροπή ε, είναι και ο κριτής και αυτός που υλοποιεί την πρωτοβουλία. Ε, σιγά σιγά θα εκλείψει η δυνατότητα συγκέντρωσης μεμονωμένων πρωτοβουλειών και μετά το 2022 θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ολοκληρώνεται λοιπόν η διαδικασία κάψη διάρκεια και δίνουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Άνσιπ για να κλείσει με μια παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεισφορά του σε αυτή τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Επιτροπή έχει αποδείξει ότι όταν μια πρωτοβουλία είναι επιτυχημένη, της ε, δίνουμε όλη την πολιτική προσοχή η οποία της αξίζει. Οι πρωτοβουλίες των πολιτών έχουν πραγματική επίπτωση στις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην νομοθεσία που προτείνεται. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ένα εργαλείο το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο στη διάθεσή τους για να ζητήσουν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Η αναθεωρημένη ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα διευκολύνει τους πολίτες να ακούγεται η φωνή τους περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε. Ο κύριος Λαμασούρ εκ μέρους του εισηγητού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έλεγα ότι ο συνάδελφος Κάμπρας συνόψισε με αξιοθαύμαστο τρόπο την προστιθέμενη αξία που κομίζει αυτή η μεταρρύθμιση, αλλά και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί ενδεχομένως ε, σε, διάφορα, σε διάφορους κύκλες κύκλους. Υπάρχει μια παρανόηση για αυτό το πολύ κεντρικό σύστημα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα ήθελα να πω στον Αντιπρόεδρο κύριο Καστάλτο γιατί αν είχε γίνει αποδεκτό, αν έγινε αποδεκτό αυτό το σύστημα έγινε αποδεκτό κατόπιν αιτήματο των υποψηφίων που υιοθέτησαν αυτή την πρωτοβουλία και που ήθελαν να διασφαλίσουν ότι θα τύχουν απολύτως ισότιμης μεταχείρισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η κεντρική διαχείριση είναι τεχνική και εγγυάται την πολιτική ουδετερότητα και την νομιμότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων που υιοθετούν και ε, βρίσκονται στις απαρχές της ανάληψης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας. Από τη στιγμή που ξεκινά τριμερής διάλογος, Καμία τροπολογία δεν είναι αποδεκτή χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και άρα για να αλλάξουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ασχοληθεί το επόμενο Κοινοβούλιο και η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα να μην δώσουμε την εικόνα ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο για πέντε χρόνια έχει οθετήσει δεκάδες νομοθετικά κείμενα εκτός από το κείμενο που φιλοδοξεί να δώσει νέα εξουσία και νέα δύναμη στον Ευρωπαίο πολίτη. Ας μην δώσουμε αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συζήτησης αγαπητοί συνάδελφοι. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης έκθεση της κυρίας Σάντρα Καλνιέτη για την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Δεν θα υπάρχει διαδικασία catch the eye ούτε διαδικασία με μπλε κάρτες κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ξεκινούμε ευθύ αμέσω με την κυρία εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. President. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τίτλος της έκθεσής μου είναι έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Δεν ήταν εύκολο το έργο να εγκρίνουμε μια έκθεση για τις σχέσεις αυτές σε μια κατάσταση όπου επιθέσεις που υποστηρίζονται από το ρωσικό κράτος γίνονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της χρησιμοποιώντας υβριδικές τεχνικές ε, πολέμου. Ως αποτέλεσμα, Μεγάλο μέρος της έκθεσης αφορά την αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της για την αποτροπή των υβριδικών απειλών. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την κατοχή της Κρυμαίας, τονίζουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε στη φυσιολογική κατάσταση μέχρι ότου η Ρωσία αποκαταστήσει πλήρω την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη βάση των σχέσεών μας με τη Ρωσία, διότι δεν μπορεί πλέον να θεωρείται στρατηγικός εταίρος η ξεπερασμένη εταιρική σχέση, συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία με την Ρωσία θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του ΟΑΣΕ. δεν υπάρχει πια χρόνος ε, για ευγενική διπλωματική γλώσσα και δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος, ε, δεν υπάρχει τόπος για ε, νέες μεγάλες πρωτοβουλίες συνεργασίας με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να κατέχει τμήματα της Ουκρανίας και ε, επιφέρει υβριδικές επιθέσεις εναντίον άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Βεβαίως, θα πρέπει να συνεχίσουμε την επιλεκτική συνεργασία με τη Ρωσία σε τομείς ζωτικού συμφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν οι παγκόσμιες προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια στην ενέργεια, ψηφιοποίηση, μη διάδοση πυρηνικών όπλων, καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι κάποιες από αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί για τις κυρώσεις ε, τις οποίες θα πρέπει να ε, παρατείνουμε όσο συνεχίζονται οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία και θα πρέπει να είναι σαφέ το μήνυμά μα προ τη Ρωσία όσον αφορά τι κυρώσει, περισσότερε κυρώσει για περισσότερε παραβιάσεις και λιγότερε κυρώσει για λιγότερε παραβιάσει. Όσο βλέπουμε επιδείνωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί υιοθετώντα ένα ευρωπαϊκό νόμο, αντίστοιχο του Magnitsky Act, δημιουργώντας ένα καθεστώ κυρώσεων ε, σε σχέση με τι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κλειδί για πιο αποτελεσματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας είναι η συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Αυτό ισχύει απολύτω και για το Nord Stream 2, ένα έργο το οποίο αυξάνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο. Απειλεί την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και για την ε, διεθνή και ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Άρα θα πρέπει ο Nord Stream 2 να σταματήσει. Οι συστάσει ε, για το τι πρέπει να γίνει με τη Ρωσία στην έκθεσή μου δεν είναι πάρα πολλέ, αλλά κάποιε από αυτέ πρέπει να αναφερθούν συγκεκριμένα. Πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξη στι επαφέ μεταξύ πολιτών γενικότερα και συγκεκριμένα επαφέ